Good day, everybody. Buongiorno, come Good day, everybody. Thank you for being here. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και για να ξεκινήσουμε, να περάσω αμέσως στις ανακοινώσεις. Είναι μια από αυτές τις μέρες που είναι φοβερά πολύ άσχολη. Η Επιτροπή μας έχει φοβερά φορτωμένο πρόγραμμα. Έχουμε πάρα πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη, πρέπει να διατρέξουμε. Λοιπόν, ξεκινώ ανακοινώνοντας με έχετε ακούσει από το λέω, να είστε συνεργάσιμοι για να μπορέσουμε να προλάβουμε. Είναι μια μέρα που θα πρέπει πραγματικά να δώσουμε προσοχή στο χρόνο. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί στο πώς αποδίδουμε το χρόνο αγόρευσης. Όσοι προβλέπονται, ο συντονιστέ ή κάτι άλλο θα πάρουν δύο λεπτά και οι υπόλοιποι ένα λεπτό δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Διότι είναι μια τέτοια μέρα που δεν έχουμε λεπτό για χάσιμο. Ξεκινάμε λοιπόν εγκρίνοντα την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Οπότε περνάμε στι ανακοινώσει του Προέδρου. Ω προ το γλωσσικό καθεστώ, το βλέπετε, όλε οι γλώσσε, εκτό από φιλανδικά, λετωνικά, λιθουανικά και γελικά. Μετά, συστάσει των συντονιστών. Κρι Πίτερ, εισηγητή για την έκθεση Ιδίας Πρωτοβουλία για την πράξη ψηφιακών υπηρεσιών. Χαβιέρ Μορένο, εισηγητής για τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής ε, υπηκών των χωρών ε, για σκοπούς ε, απασχόλησης υψηλών δεξιοτήτων γαλάζια κάρτα. Έλενα Γιόντσεβα, εισηγήτρια για την ΕΑΖΟ. Μίριαμ Ντάλι, εισηγήτρια για την νόμιμη μετανάστευση και την εργασία. Άλλη Κούνκε, οριζόντια οδηγία ίσης μεταχείρισης. Και πάλι ε, είπαμε η μεταχείριση και η οδηγία της, μετά γνωμοδοτήσεις διαπραγματεύσει για τις μελλοντικέ σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Λοραν Βίντσε, Τάγκ, ε, βελτίωση τη εσωτερικής αγοράς ε, με την τη αγορά, Ασίτα Κάνκο, οι ηθικέ πτυχέ τη τεχνητής ευφυΐας Πάτρικ Τζακ Γιάκη, η τα θέματα κρατικής εξουσίας και ε, του διεθνούς δικαίου σε θέματα ε, ποινική δικαιοσύνης. Εάν δεν υπάρχουν εδώ λοιπόν αντιρρήσεις, να ανακοινώσω ότι έχουμε μια πολύ σύντομη ηλεκτρονική ψηφοφορία αύριο, στις 12 και 4. Παρακαλώ λοιπόν να το θυμηθείτε και να φέρετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Περνάμε λοιπόν στο πρώτο επί της ουσίας σημείο της ημερήσιας διάταξης, που θα μας απασχολήσει αρκετά, όλο το πρωί. Μια ειδική ακρόαση για την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνου, του λεγόμενου Δουβλίνου 3, περιμένοντας και αναμονή του Δουβλίνου 4. Τώρα θα ασχοληθώ με το Δουβλίνο 3. Αυτό ε, εφαρμόζεται και υλοποιείται εδώ. Θα συζητήσουμε λοιπόν τα πορίσματα της διαδικασίας υλοποίησης του κανονισμού δουβλίνου 3. Θα τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά για αυτό το θέμα που είναι ύψης της σημασία και γιατί θέλουμε να προχωρήσει το όλο πακέτο οι όλοι δεσμοί μέτρων για το άσυλο, ένα καθοριστική σημασία νομοθέτημα. Και επίση η Επιτροπή δεν έχει δημοσιεύσει εκθέσει για την υλοποίηση από το 2016. Οι συγγητέ και σκιώδει το έχουν επισημάνει πισταμένο αυτό. Και εδώ θα σας δώσουμε πληροφορίες για το ε, ιστορικό της σύνταξης και της χάραξης του νέου κανονισμού Δουβλίνο 3 για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό πόρισμα, τελική έκβαση αυτή τη νομοθετική διαδικασία που έχει μπλοκαριστεί τόσο καιρό. Εδώ λοιπόν σήμερα έχουμε ένα-δυο πάνελ. Πρώτο πάνελ ε, εθνικές αρχές ε, από Ελλάδα, Γερμανία, Σουηδία, Ισπανία και Ιταλία. Το δεύτερο πάνελ είναι ενδιαφερόμενοι και συμμετέχοντες ευρωπαϊκού επίπεδου. Και μετά θα ακούσουμε τον εισηγητή μας για το όλο θέμα, ή την εισηγητριά μας, την κυρία Κελέρ, και τους ε, Σκιώδη. Θα ακούσουμε και τους Σκιώδη. Και μετά θα έχουμε και λίγο χρόνο προσυζήτηση με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Όμως το λέω ευθύ εξ αρχή. Ένα λεπτό στον καθένα. Σκιώδη και εισηγητή, εισηγήτρια, δύο λεπτά. Τώρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κυρία Σάσα Αρλιουάλ. Αρλιουάι, αν τα λέω καλά. Αλριχάουι. Πώς σας λένε. Με συγχωρείτε. Προσπαθώ να το πω σωστά. Αλεριχάουι. Το Διεθνές Δίκτυο Προσφύγων. Προστασία για όσους έχουν δικαίωμα ε, στη διαδικασία του Δουβλίνου. Έχετε το λόγο για 7-10 λεπτά. Θα προλάβετε. 8. Ωραία. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πάρω το λόγο. Είναι σημαντικό προνόμιο για μένα να βρίσκομαι εδώ, να μοιραστώ την ιστορία μου και τις απόψεις μου για το Δουβλίνο. Καθότι μπορώ να θεωρήσω τον αυτό μου επιζήσασα της ε, ιστορίας του Δουβλίνου. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να ζητήσω από όλους εσάς ε, να σκεφτείτε μια στιγμή τα εξής ερωτήματα. Υπάρχει κανείς εδώ που να έχει κάποια εμπειρία ε, εξαναγκασμού να φύγει από την πατρίδα του, να αφήσει πίσω οικογένεια, φίλους, δουλειά, σπίτι. Κάποιος που να έχει ζήσει τον εκτοπισμό ε, ή την εξαναγκαστική μετανάστευση για διάφορους λόγους. Και τέλος, μπορείτε να φανταστείτε εσείς να βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση. Ελπίζω να μην βρεθείτε ποτέ φυσικά. Σε μια κατάσταση λοιπόν όπου όλοι εσείς και η οικογένειά σας αποφασίζετε να φύγετε. Μπορείτε να φανταστείτε σε ποια χώρα θα ζητήσετε άσυλο. Τώρα, και πάλι, καλημέρα, ονομάζομαι Σάζα, είμαι πρόσφυγας, μένω στη Γερμανία. Πριν δούλευα για την ύπατη αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες στη Συρία, και δούλευα με τους πρόσφυγες πριν ε, φανταστώ ότι μπορεί να γίνω και εγώ πρόσφυγας κάποια στιγμή. Πώς ξεκίνησε το ταξίδι μου. Εγώ λοιπόν ετήθηκα άσυλο στη Σουηδία, αλλά είχα αμερικανική βίζα. Μετά έμεινα για 1,5 χρόνο στην Σουηδία υπήρξε μια διαλκεστίνητα μεταξύ ΙΠΑ και Σουηδίας για το ποιο θα αναλάβει την υπόθεσή μου. Ξέρω ότι εκεί δεν πρόκειται για διαδικασία από το Δουβλίνο. Μου είπαν ότι υπάρχει κάποια άλλη σύμβαση, κάτι τέτοιο. Μετά από 1,5 χρόνο ελήφθη η απόφαση να μην με αναλάβουν είπα, αλλά και από τη Σουηδία αρνήθηκαν, απέριψαν το αίτημα μου. Είπαν ότι μπορεί να μείνει τέσσερα χρόνια εδώ και να ξεκινήσει και πάλι μια καινούργια υπόθεση. Κατά τη διάρκεια αυτού του 1,5 έτου δεν είχα το δικαίωμα να εργαστώ, να σπουδάσω ή να κάνω οποιαδήποτε άλλου είδους ε, φυσιολογική ζωή. Γι' αυτό αποφάσισα να φύγω από αυτή την κατάσταση. Δεν ήθελα να χάσω 1,5 χρόνο και μετά πάλι άλλα 4 χρόνια αναμένοντα νέα απόφαση του Σουηδία. Γι' αυτό και είπα ότι θα φύγω και θα ζητήσω άσυλο σε άλλη χώρα. Πήγα λοιπόν στη Γερμανία. Εκεί έκανα και πάλι αίτηση. Ήξεραν ότι είχε απορριφθεί το αίτημά μου στη Σουηδία, δεδομένου του συστήματος του Δουβλίνου, το γνώριζαν και είπαν εντάξει πρέπει να δούμε αν μπορούμε να σας δεχθούμε ή όχι. Ξεκίνησε λοιπόν πάλι μια διαδικασία ενό έτου, περιμένοντα μια τελική απόφαση για την υπόθεσή μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, δεν μπορούσα να ξεκινήσω τα μαθήματα ένταξη, τίποτα. Είχε σταματήσει η ζωή μου. Είχα όμως πάντα την ελπίδα, την φιλοδοξία να είμαι ενεργή, δραστήρια, να μάθω τη γλώσσα, να είμαι καλός άνθρωπος Είχα και όλες αυτές τις εμπειρίες από την προηγούμενη μου εργασία και ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ε, εμπειρία ε, για τη νέα μου χώρα. Τελικά όμως τι, έπαθα κατάθλιψη. Έχασα τις ελπίδες μου. Ήμουνα σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Με βάση τη δικασία του Δουβλίνου, λοιπόν, ε, Βλέπω ότι αυτή είναι μία από τις επιπτώσεις του Δουβλίνου στους πρόσφυγες. Πρέπει λοιπόν από αυτή την άποψη να εξετάσουμε το Δουβλίνο. Από την άποψη των, των κοινοτήτων που πλήττονται. Δεν έχει να κάνει λοιπόν αυτή η ιστορία μόνο με όσους κάθονται σε ένα γραφείο και μας ε, εξετάζουν ω στατιστικά στοιχεία ή υποθέσεις και φακέλους. Πρέπει να ακουστεί πραγματικά η υποθεσεις και φακέλου. πρεπει να ακουστει πραγματικα η φωνη μας. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εργαστούμε από κοινού. Να ακούσουμε σε ποιες περιπτώσεις έχει επιτύχει και σε ποιες περιπτώσεις έχει, έχει αποτύχει ο κανονισμός του Δουβλίνου γιατί πρόκειται για ανθρώπους πίσω από αυτά τα νούμερα, πίσω από αυτούς τους φακέλους. Έχουμε αλλάξει την προσέγγισή μας και πλέον μιλάμε μόνο για υποθέσεις, φακέλους και στατιστικά στοιχεία. Εγώ εργαζόμουν για την υπάτη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στο παρελθόν. Εργαζόμουν λοιπόν, ξέρω τον εργασιακό φόρτο. Δεν σκεφτόμουν ποτέ του ανθρώπου. Έλεγα: Έχω πολλή δουλειά, θα δω τι θα κάνω. Αλλά αν σκεφτείτε ότι στο δικό μου μικρό γραφείο έχουμε 20.000 φακέλους που αφορούν ανθρώπους, γυναίκες, ασυνόδευτα παιδιά. Και αν δείτε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και αλλού, δεν νομίζω ότι είναι μια σωστή προσέγγιση. Όταν αποφασίζουμε ελαφρά την καρδία για ανθρώπινες ζωές, χωρίς να σκεφτούμε κάτι παραπάνω, όπως έκανα και εγώ τότε. Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα βρισκόμουν ποτέ σε αυτή τη θέση εγώ, η αδελφή μου, ο αδερφός μου, η οικογένειά μου θα ανήκαν σε αυτή την κατηγορία που πλήττεται. Από πλευράς προσφύγων, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι το Δουβλίνο έχει αποτύχει σε ορισμένες περιπτώσεις. Αντί να υπάρχει επιμερισμός ε, των ευθυνών με τα κράτη-μέλη, ο ένας μετατοπίζει την ευθύνη στον άλλον σαν μπαλάκι πετάνε τους πρόσφυγες από τη μια χώρα στην άλλη. Κανείς δεν θέλει να τους αναλάβει. Όλοι λένε όχι δεν είναι δική μου ευθύνη, είναι δική σου. Και μέσα σε όλα αυτά οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι. Τους φερόμαστε πάρα πολύ άσχημα ενώ παράλληλα συζητούμε ποιο θα του αναλάβει και τι θα γίνει. Δεν μπορούν να πάνε ένα σχολείο σε κάποιε περιπτώσει, δεν μπορούν να εργαστούν να ζήσουν τη ζωή του. Εγώ λοιπόν από το δικό μου παράδειγμα δείχνει ότι το Δουβλίνο περιορίζει την κινητικότητά μας, τις δυνατότητες μας ε, να αναζητήσουμε ασφάλεια και προστασία. Το Δουβλίνο επίσης δεν ε, αποσκοπεί στην ε, ισομερή κατανομή των ευθυνών μεταξύ κρατών μελών. Για παράδειγμα, η Ιταλία έχει λάβει περίπου 1 τρίτο των ετούντων άσυλο που έχει μεταφερθεί από άλλο κράτος μέλος. Μπορούμε να μιλήσουμε για την Ελλάδα η Ουγγαρία σταμάτησε να δέχεται ε, πρόσφυγες με κάποιον τρόπο. Βλέπω λοιπόν ότι δεν δουλεύει καλά το σύστημα του Δουβλίνου. Μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει κάποιο είδους ε, παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων από αυτή την άποψη. Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση. Κάποιες φορές δεν εξετάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους ε, στα επιμέρους κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο. Αν δείτε, για παράδειγμα, στην Ελλάδα. Εκεί, στα κέντρα υποδοχής, έχετε δει πώς ε, ζουν οι άνθρωποι. Αν όλοι μας, λοιπόν, ως κράτη-μέλη, παρέχουμε τις ίδιες υπηρεσίες, δεν νομίζω ότι θα ε, υπάρχει κάποια διαφορά. Δεν θα πάνε στην, στη Γερμανία εάν έχουν τις ίδιες υπηρεσίες ε, στην Ελλάδα. Αναφέρεται στο Δουβλίνο ότι δεν εγγυάται κανεί ε, την χορήγηση ασύλου σε όλα τα κρατημέλη και δεν ε, ε, συμπεριλαμβάνεται η παρουσία ενό μέλου οικογένεια. Εμεί είχαμε ευθύνη έκκληση για σωστή συμμετοχή. Είχαμε ζητήσει από όλα τα κρατημέλη να έρθουν και να μιλήσουν απευθεία με τι θυγόμενε κοινότητε και να αναζητήσουμε από κοινού λύσει. Η δική μου σύσταση λοιπόν είναι η εξή η εμπειρία μου μου δείχνει ότι η λύση στο προσφυγικό θα ξεκινήσει από την εμπλοκή των ε, προσφύγων που έχουν ζήσει οι ίδιοι, έχουν βιώσει αυτά τα πράγματα. Παρότι οι επιμέρους ιστορίες μπορεί να διαφέρουν, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και οι λύσεις που θα πρέπει να αναζητήσουμε είναι ε, τρομερά παρόμοιες. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονό ότι ο περιορισμός της ε, μετακίνηση που απορρέει από το σύστημα του Δουβλίνου είναι μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγε σε όλη την Ευρώπη. Και για όλους εμάς ε, που τα καταφέραμε και είμαστε προνομιούχοι, αν θέλετε, ενώ δεν είμαστε στην ουσία. Δεν είναι προνόμιο το να χαίρουμε των δικαιωμάτων μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από αυτές τις υποθέσεις, πίσω από αυτά τα στατιστικά νούμερα υπάρχουν άνθρωποι. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα σύστημα που θα μεταχειρίζεται τους ανθρώπους με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μοιραστήκατε την μαρτυρία σας με ιδιαίτερη εντυμότητα και ειλικρίνεια και ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Να ξεκινήσουμε τώρα με το πάνελ να ξεκινήσουμε με του εκπροσώπου από τι διάφορε εθνικέ αρχέ που έχουμε προσκαλέσει. Απλώ να σα παρακαλέσω να σεβαστείτε το χρόνο. Η αρχική μου ε, πρόθεση ήταν να έχουμε 10 λεπτά ο καθένα. Αν μπορείτε να προλάβετε και σε 9, καλό θα ήταν. Ε, θα προσπαθήσουμε να μην χάσουμε χρόνο. Να ξεκινήσουμε χωρί περαιτέρω καθυστερήσει, λοιπόν. Ελλάδα, Γερμανία, Σουηδία, Ισπανία και Ιταλία. Από την Ελλάδα θα ξεκινήσουμε, αν έχω καταλάβει καλά. Μα ακούτε, θα ξεκινήσετε, έχετε το λόγο. Έχετε 9 λεπτά. Um, my name is Marcos Caravia. Λέγομαι Μάρκος Καραβίας και είμαι επικεφαλής υπηρεσίας ασύλου εδώ στην Ελλάδα και θα παρέμβω από την Ελλάδα Έχω την κυρία Παπαϊλιού δίπλα μου που είναι επικεφαλή τη μονάδα Δουβλίνου στη χώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σα για την πρωτοβουλία αυτή, για την πρόσκληση και για το γεγονό πω μας επιτρέπετε να λάβουμε μέρο μέσω ε, τηλεδιάσκεψης. Θεωρούμε ότι είναι η ενδεδειγμένη στιγμή για να αναθεωρήσουμε την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνου 2 και το κατά πόσο κατάφερε να πετύχει τους δεδηλωμένους στόχου δηλαδή να εξασφαλίζει τις οικογενειακές ενότητες, να στηρίζει τα δικαιώματα των ανηλίκων και με ταχύ τρόπο να αποφασίζει ποιο είναι το κράτο μέλος το οποίο είναι αρμόδιο για να χορηγήσει ή όχι ε, το καθεστώς προστασίας. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε καταρχήν υπό ποιε συνθήκες ε, σχεδιάστηκε το Δουβλίνο 3 και, εφαρμόστηκε. Και να σας πω πως ε, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε ε, το θέμα των προσφύγων, των προσφύγων θεωρήσαμε πως αυτό ο κανονισμός δεν είναι ούτε λύση για τη μαζική μετανάστευση, ούτε εργαλείο διαχείρισης αυτής. Το θέμα λοιπόν είναι, μπορούμε να ε, κοιτάξουμε το πώς εφαρμόστηκε η, ο κανονισμός Δουβλίνο 3 στα πλαίσια τα οποία διαμορφώθηκαν από τα γεγονότα τα οποία προηγούνται και ακολουθούν το 2015. Ακούστηκε πως αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια εποχή post κρίσεως, όπου ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου στην Ευρώπη μειώθηκε σε επίπεδα 2014. Η κατανομή των αιτήσεων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δίνεται με ίσο τρόπο, οπότε η ε, με άνισο τρόπο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα το σύστημα της υποδοχής ε, και διεκπαιρέσεις έχει ε, αντιμετωπίσει ιδιαίτερες πιέσεις λόγω ροών και από τα χερσαία σύνορα τα τελευταία χρόνια αλλά και από τα νησιά. Και οι ροές αυτές το τελευταίο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκαν ριζικά. Το 2019, εν συντομία, η υπηρεσία ασύλου καταχώρησε 77.287 ετούντες άσυλο. Στο νησί της Λέσβου 22.252 ε, κατέθεσαν αίτηση ασύλου για το έτος 2019. Αν λοιπόν η Λέσβος ήταν ε, εθνικά κυρίαρχο κράτος μέλος, θα είχε καταχωρήσει ε, τον 10 τον, δέκατο πιο υψηλό ρυθμό αιτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφαρμογή λοιπόν του κανονισμού. Θέλουμε να σας δώσουμε κάποιο feedback από την ε, οπτική γωνία της Ελλάδος. Τώρα, αν δούμε τα κριτήρια ιεραρχικά όπως έχουν αναφερθεί στον κανονισμό, η επανένωση ε, ε, οικογενειών και κυρίως η επανένωση ανηλίκων με την οικογένειά τους είναι πρωταρχικός στόχος. Και από τα 10.560 αιτήματα που έχουμε στείλει ως μονάδα Δουβλίνου στην Ελλάδα, που είναι η μονάδα που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του κανονισμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία έχει να κάνει με την οικογενειακή επανένωση. Στην πράξη προέκυψαν μία σειρά από θέματα για την εφαρμογή των άρθρων 8 με 11 που αφορούν κυρίως την οικογενειακή επανένωση. Και θα ήταν ασφαλές να πούμε πως υπάρχει μια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις ε, αρμόδιες μονάδες Δουβλίνου στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ένα από τα ζητήματα που ε, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η τεκμηρίωση. Η τεκμηρίωση που χρησιμοποιείται, όπως επίσης ε, ε, τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους οικογενειακούς δεσμούς. Κάποια κράτη-μέλη υποδοχής επιβάλλουν ένα, μια απέτηση τεκμηρίωσης πολύ υψηλή και θεωρούν πως οποιασδήποτε ε, έμεσες, ε, οποιασδήποτε έμεσα στοιχεία ε, τεκμηρίωσης δεν γίνονται αποδεκτά. Για παράδειγμα, ζητούν να γίνουν τεστ DNA για να αποδειχθεί ο οικογενειακός δεσμός. Κάποια άλλα κράτη-μέλη δέχονται τις μερικές, τα, μερικά, τα μερικώς τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία, όπως επίσης και τα περιστασιακά ή τα έμεσα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πως επειδή αργεί η οικογενειακή επανένωση λόγω δυσκολίας τεκμηρίωσης, πάρα πολλές από αυτές τις ε, ε, υποθέσεις ε, χάνουν χρόνο. Τώρα, για τους ανηλίκους μπορώ να σας πω πως έχουμε αυτό το οποίο εμείς αναφέρουμε ως ερμηνευτικές αποκλήσεις. Κάποια κράτη-μέλη θεωρούν πως το νομικό καθεστώς των ε, μελών της οικογένειας είναι διαφορετικό. Δηλαδή, αν έχει ε, υπηκότητα, αν ε, έχει άδεια διαμονής, όλα αυτά καθορίζουν το καθεστώς και την διεκπαιρέωση που γίνεται για την επανένωση. Κάποιοι δεν εφαρμόζουν καθόλου το άρθρο 8. Αν ο συγγενής ή το μέλος οικογένειας έχει, ε, για παράδειγμα, ε, απαγόρευση επανένωσης ε, με είσοδο στη χώρα ή προσωρινή άδεια διαμονής. Επίσης, εντωμεταξύ από τη στιγμή της αίτησης, αν εντωμεταξύ έχει ενηλικιωθεί ο ανήλικος, δεν τον δέχονται καταπατώντας το 7.2 του κανονισμού. Επίσης, ξεχνούμε πολύ συχνά ε, πως υπάρχει η θεμελιώδης απέτηση του ε, ε, συμφέροντος του ανήλικου που πρέπει να, λάβετε, να λαμβάνετε υπόψη στο άρθρο 24 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άλλων διεθνών μεσών που θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη και πολλές φορές δεν γίνονται σεβαστά. Για τους ανήλικους να συνεχίσω λέγοντας πως η μονάδα Δουβλίνου στην Ελλάδα έχει σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία, την ΕΑΣΟ και άλλους ε, εμπλεκόμενους ε, φορείς ε, ένα εργαλείο για την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος και ένα ερωτηματολόγιο, μια κατάσταση ελέγχου checklist για να απαντά τα ερωτηματικά που θέτουν τα άρθρα του κανονισμού του Δουβλίνου. Και για τα ασυνόδευτα ανήλικα που ζητούν ετούνται ε, διεθνή προστασία στην Ελλάδα με συγγενείς που διαβιούν σε άλλο κράτος ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούμε το εργαλείο που για μας είναι το πιο άριστο εργαλείο για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντα του ανήλικου. Και βέβαια χρειαζόμαστε συνεργασία με τα άλλα κράτη-μέλη για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ε, κανονισμού Δουβλίνου. Με την εργαλειοθήκη αυτή ε, επιδιώκουμε να μαζέψουμε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να σεβαστούμε τα κριτήρια που θεσπίζει ο κανονισμός. Και με στόχο αυτό, για να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση, συνεντεύξεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με το παιδί, και οι πληροφορίες που λαμβάνονται ε, τεκμηριώνονται με τα απαραίτητα παραστατικά. Έτσι ώστε να καταθέτουμε αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες όταν στέλνουμε ένα αίτημα ε, μέσω αυτού του εργαλείου του, της αξιολόγησης του βέλτιστου ε, του συμφέροντος του παιδιού και αυτό έχει ε, διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων Δουβλίνου και τελικά έχει ε, βελτιώσει τη διαδικασία επανένωση οικογενειών με ανήλικα μέλη. Τώρα, για τα εισερχόμενα αιτήματα που λαμβάνουμε εμείς ως μονάδα Δουβλίνου με τις άτυπες ε, διελεύσεις και ε, με την στέγαση των ετούντων ε, και αυτό ε, το κάνουμε λαμβάνοντας υπόψη τα hit που έχει λάβει βάση Eurodac, ε, έχουμε κάποιο περιθώριο ε, ερμηνείας. Παρόλα αυτά, το κριτήριο της χώρας πρώτης εισόδου, πρώτης διέλευσης, καταλαβαίνετε, επιβαρύνει ιδιαίτερα τα κράτη που είναι στα σύνορα και κυρίως τα εθνικά συστήματα υποδοχής. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος εδώ να σημειώσει πως έχουμε δεχτεί στη μονάδα μας το 19 710 τέτοια αιτήματα σε ε, σύγκριση με το 229 αιτήματα του 2018. Παρόλο λοιπόν την αυξημένη πίεση βλέπουμε ότι έχουμε έναν αριθμό ε, υποθέσεων ε, που εφαρμόζονται οι διατάξεις. Για να καταλήξω, μια και έχουμε περιορισμένο χρόνο, ενδεχόμενες ελλείψεις του κανονισμού Δουβλίνο 3 ενδεχομένως συνδέονται με τον τρόπο που έχει δομηθεί και όχι μόνο με την εφαρμογή στην πράξη. Δηλαδή, είναι ε, περίπλοκος, είναι γραφειοκρατικός, είναι, ε, δίνει δυνατότητα ε, διαφορετικών ερμηνειών με ε, τρόπο που μπλοκάρει την εφαρμογή του. Είναι τα κράτη-μέλη στα σύνορα που αντιμετωπίζουν την πίεση των νέων αφήξεων και πιέζονται να αναλάβουν και την ευθύνη ε, για τα οτσετούντες άσυλο που υποβάλλουν ε, ε, χορήγηση ασύλου σε παραπάνω από ένα κράτος μέλος. Οικογενειακή επανένωση. Τα, οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα κράτη-μέλη και υπάρχουν και κάποιες ρήτρε ε, οι οποίες ε, θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για να παραμένουν μαζί οι οικογένειες και ε, εφαρμόζονται με, ανάλογα με τη διακριτική αξιολόγηση κάθε κράτους μέλους. Χρειάζεται λοιπόν αναθεώρηση σύμφωνα με εμά ο κανονισμός αυτός, ένα σύστημα που θα πρέπει πρώτον να λειτουργεί και δεύτερον να είναι ανθεκτικό σε τέτοιου είδους κρίσεις. Δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογα βαρύ για κάποια κράτη-μέλη, όπως συμβαίνει σήμερα, και θα θα πρέπει να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε μία μόνιμη κρίση μέσω αυτού σε κάποια κράτη ε, στα σύνορα. Λείπει λοιπόν ε, το στοιχείο της δικαιοσύνης, της δίκαιης κατανομής που θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Καραβιά που εκπροσωπείτε την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου. Ωστόσο θα επιμείνω. Οι επόμενοι παρεμβαίνοντες, παρακαλώ σεβαστείτε το όριο ε, χρόνου. Έχουμε φοβερά φορτωμένη μερισσία διαταξή δύο πάνελ και πρέπει να προλάβουμε να ακούσουμε και τους εισηγητές και τους σκιώδεις και να έχουμε και χρόνο για συζήτηση. Παρακαλώ οι υπόλοιποι προσπαθήστε να σεβαστείτε το χρόνο για να τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε κύριε Καραβία. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, δική σας κατάθεση. Θα ακούσουμε τώρα την, τον Γερμανό εκπρόσωπο, τον κύριο Λέσερ, από το Υπουργείο Εσωτερικών και ε, υποδιευθυντή για τα θέματα του νόμου ασύλου και της διαδικασίας ασύλου. Και τον κύριο Σφίμελ Φένινγκ, ε, ο οποίος είναι από το Μοσπονδιακό Γραφείο Μεταναστών και Προσφύγων στον Πόχουμ. Παρακαλώ προσπαθήστε σε 9 λεπτό, 9 λεπτά, 10 το πολύ διότι ενώ όλοι πάνε στα 11, δεν θα τα καταφέρουμε. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Λέγομαι Σίμελ Φένικ και είμαι υπεύθυνο στον Πόχουμ για τα θέματα του Δουβλίνου. Ήθελα αρχικά από πρακτική σκοπιά να παρουσιάσω τα προβλήματα τη υλοποίηση του Δουβλίνου 3 στην Γερμανία. Η Γερμανία, όπω ξέρετε, είναι ομοσπονδιακό κράτο. Οπότε υπεύθυνη για την εξέταση των αίτησεων ασύλου είναι ομοσπονδιακή υπηρεσία στη χώρα μας. Το ίδιο και για τις διαδικασίες του Δουβλίνου. Στην ε, Γερμανία μοιράζονται στα διάφορα ομοσπονδιακά κρατήδια οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Εκεί καταγράφονται οι ετούντες, εκεί γίνονται οι έλεγχοι και η εξέταση του κατά πόσον βρίσκονται σε ευάλωτες, ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Επίσης, ελέγχονται τα στοιχεία τους στο σύστημα ΒΙΣ και μέσω των εθνικών βάσεων δεδομένων που διαθέτουμε. Οι ετούντες επίσης ελέγχονται βάσει των προϋποθέσεων της διαδικασίας του Δουβλίνου. Έχουμε ένα Έχουμε τρία κέντρα στο Βερολίνο, στο Μπάιρεουτ, στο Μπόχουμ και στο Βερολίνο. Τρία κέντρα που ασχολούνται με τις διαδικασίες του Δουβλίνου και εξετάζουν τις αιτήσει ε, σε κεντρικό επίπεδο. Όταν έχουμε επαφέ με άλλα κρατημέλη, ελπίζουμε να έχουμε θετική απάντηση για να ελεγχθούν οι πληροφορίες και έχουμε και συγκεκριμένη προθεσμία για να λάβουμε τις απαντήσεις. Ανάλογα λοιπόν με την απόφαση που τα λάβουμε, συνεργαζόμαστε και με την ε, αστυνομία και τις τοπικές αρχές. «49.000 αιτήσεις ε, έχουν γίνει και 8.400 άτομα ε, είναι όσοι εξετάστηκαν για να καλυφθούν ε, τα πρώτα κενά του συστήματος. Εδώ στην Γερμανία ε, έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε ένα τρίτο των αιτήσεων. Κατά την υλοποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου, λοιπόν, και με την καθημερινή μας εμπειρία, αντιμετωπίζουμε διαφορετικά προβλήματα. Έχουμε διαφορετική διάρθρωση των, ε, της εκτάσεως των αιτήσεων, όμως ανάλογα με την κάθε περίπτωση υπάρχει και διαφορετική ερμηνεία. Οπότε καταλήγουμε να έχουμε και κάποιες φορές απόρριψη για διαφορετικούς λόγους. Το βασικό είναι να, υπάρχει, ε, να υπάρχουν ξεκάθαρα αποδεικτικά στοιχεία και ένα παράδειγμα είναι ο ορισμός του άρθρου 12, εδάφιο 4, για το πόσο ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα, μια ενισχύς θεώρηση ή όχι. Και πώς ε, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν τα διάφορα κράτη-μέλη. Βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού. Μεταξύ των 100 μελών Υπάρχουν σε επιμέρου τομεί δυνατότητε συνεργασία μεταξύ των κατών μελών, σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση τη αιτήση ασύλου για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με το Δουβλίνο αναγκαστικά και υπάρχουν όργανα και μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όταν δεν έχουμε πληροφορίες για τον ετούντα άσυλο. Με διάφορα ερωτηματολόγια. Όταν δεν είναι δυνατή λοιπόν η επιμέρους επαλήθευση όλων των στοιχείων, εκεί ε, χρειάζεται η περαιτέρω συνεργασία και πολλές φορές υπάρχει και ακύρωση όταν είναι πολλά τα προβλήματα που συσσωρεύονται σε μια συγκεκριμένη ε, περίπτωση. Οι δυνατότητα συνεργασίας με τα άλλα κράτη-μέλη βέβαια πολλές φορές έχουν να κάνουν και με το κατά πόσον είναι απρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μας οι άσυλο. Έχουμε μόνον 8.500 άτομα των οποίων έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία. Πάντως, διαρκώς προκύπτουν νέες περιπτώσεις, διότι ξέρουμε ότι πολλές φορές χωρίζονται οι οικογένειε ε, και φτάνουν ξεχωριστά στη Γερμανία επίτηδε για να μπορέσουν μετά να επικαλεστούν την ε, επανένωση. Έχουμε πολλές φορές παιδιά τα οποία αποστέλλονται όπως λέμε ως άγκυρε, ως ε, πρώτο μέλος για να τραβήξουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία της οικογενειακή επανένωση. από την άποψη της διάρθρωσης και του πώς εφαρμόζεται ο κανονισμό του Δουβλίνου, αυτό που βρίσκουμε εμείς προβληματικό είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετική κατανομή των αρμοδιοτήτων και όχι μόνο βάση της προθεσμίας. Δηλαδή, όταν ε, εκπνέει η προθεσμία εξέταση μιας πρέπει να μπορεί κάποιος να αποταθεί σε άλλο κράτος μέλος γιατί ο κανονισμός προβλέπει παράταση 18 μήνες και 12 εφόσον υπάρξει σύλληψη. Ευχαριστώ. meiner Seite. Ähm, Καλημέρα σας και από τη δική μου την πλευρά λέγομαι Λέσερ και είμαι υπεύθυνο της Υπηρεσίας Ασύλου στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο μας. Θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω την παρουσίαση του συναδέλφου. Το Δουβλίνου στη Γερμανία είναι σημαντικό σύστημα, σα το παρουσίασε ο συνάδελφο. Οι διαδικασίε έχουν βελτιωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε παρόλα αυτά ότι διαρκώ υπάρχουν ελλείψει. Ελλείψεις που δεν οφείλονται μόνο στις εθνικές μας αδυναμίες, αλλά λόγω για τις διάρθρωσες του κανονισμού Δουβλίνου 3. Είναι πολύ μακρές και γραφειοκρατικές οι διαδικασίες και είναι πολύ μεγάλο το γραφειοκρατικό άχθος για τα κράτη-μέλη και για τους ετούντες. Όμως, εάν το συγκρίνουμε ε, στην ε, πράξη, ε, είναι σημαντικά τα στοιχεία. Είναι 5% στη Γερμανία το σύνολο των αιτήσεων ασύλου που τελικά ε, καταλήγουν ε, με επιτυχημένη εξετάση μέσω του συστήματος Δουβλίνου να πάνε σε άλλο κράτος μέλος και να ε, τακτοποιηθούν εκεί οι υποθέσεις τους, ενώ προηγουμένως είχαμε ένα 3%. Είναι πολύ μεγάλες επίσης οι ελλείψεις συμμετρικότητας που προκύπτουν και από τα πρώτα κράτη και τα κράτη στόχο των μεταναστών, όπως η Γερμανία οι αιτούντες άσυλο δεν μπορούν να συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο στα ίδια μέρη που όπως ξέρουμε έχουν υπερβολικό φόρτο λόγω της ε, σημαντικής συγκέντρωσης ανθρώπων εκεί. Ε, επίσης υπάρχουν υπηρεσίες που δεν είναι υπεύθυνε για τον κανονισμό του Δουβλίνου 3 και πρέπει να ασχοληθούν με αυτό. Κατά τη δική μας άποψη έχει αποτύχει το Δουβλίνο 3. Χρειαζόμαστε κατεπηγόντως ε, μια μεταρρύθμιση του συστήματος, μια νέα αρχή και σκοπός εδώ ε, είναι ε, αυτό που πρότεινε πρόσφατα και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, ε, δηλαδή κάποιε ιδέε για το πώ θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό του Δουβλίνου. Εδώ είναι τρία τα βασικά σημεία τα οποία ήθελα να παρουσιάσω. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται ένα σύστημα με πολλέ διαφορετικέ αρμοδιότητε. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα γνωρίζετε αυτά, γιατί στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία είχατε υποβάλει έτοιμα για ένα τέτοιο, είχατε υποβάλει ιδέε για τέτοιο σύστημα σύστημα, δηλαδή να υπάρχει ένα σύστημα κατανομής και ευθύνης θα πρέπει να μην εξαρτώνται όλα από την εκπνοή της προθεσμίας και να εξετάζεται δίκαια και αντικειμενικά η αίτηση του ασύλου. Μετά θα πρέπει με την μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση, να λάβουμε δραστικά μέτρα. Θα μπορούσα εδώ να δώσω πολλές ιδέες προτάσεις, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν κάθε λόγο να καταπολεμήσουν την παράνομη, τη λαθρομετανάστευση. Και εδώ χρειάζεται ένα καθεστώς κατανομής των ευθυνών, διότι δεν μπορεί να είναι διαρκώς ε, διαφωνία και αντιπαλότητα τα κρατημέλη μεταξύ του. Θα πρέπει το δικαίωμα του ασύλου να το καταρτήσουν, να το θεμελιώσουν και να γίνει πραγματικά ευρωπαϊκό. Και το τρίτο που θέλω να αναφέρω είναι ότι εδώ ε, θα πρέπει να έχουμε καλό έλεγχο των εξωτερικών ε, σύνορων, αλλά και εσωτερικώς ε, στα χερσαία σύνορα. Θα πρέπει να δούμε ε, τι ακριβώ συμβαίνει στα εξωτερικά μα σύνορα και όσοι δεν έχουν δικαίωμα να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην λαμβάνουν το δικαίωμα αυτό. Σα ευχαριστούμε κύριε Σίμελφένη. Ε, πραγματικά αυτά που ε, μας παρουσιάσατε δείχνουν ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιημένη με την κατάσταση του Δουβλίνου. Ευχαριστούμε. Και τώρα να προχωρήσουμε. Ε, επόμενο πάνελ από τη Σουηδία η κυρία Σόπολτ Λίλιμπλατ, υπεύθυνη της υπηρεσίας Δουβλίνου και ο κύριος Άξελσον, σύμβουλος της υπηρεσίας για την μετανάστευση στη Σουηδία και της μονάδας για το Δουβλίνο. Σουηδική κυβέρνηση λοιπόν, πείτε μας τι κάνει για το θέμα αυτό. Προσπαθήστε 9 λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και μία παρουσίαση PowerPoint, αλλά μόνο την πρώτη διαφάνεια θα σας δείξουμε για να έχετε μια εικόνα. Σήμερα λοιπόν μας καλέσατε να μιλήσουμε για την διαδικασία του Δουβλίνου ε, στη Σουηδία και για να θίξουμε και ορισμένα επιχειρησιακά ζητήματα κατά την εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου. Αρχικά λοιπόν θέλω να σας δώσω μια επισκόπηση της κατάστασης. Βλέπετε στην οθόνη σας λοιπόν μια γενική εικόνα ε, της διαδικασίας των βημάτων ε, που κάνει ένας ε, ενήλικας τον άσυλο για τους ε, ανηλίκους είναι διαφορετική διαδικασία, αλλά επειδή είναι πιο συνήθις για τους ενήλικες, γι' αυτό σου παρουσιάζουμε αυτήν. Έχουμε τρία βήματα λοιπόν. Πρώτον, το στάδιο της αίτηση, ε, η εξέταση της αίτηση και η διαδικασία της μετακίνησης. Την ευθύνη για το σύνολο της διαδικασίας έχει η Σουηδική Υπηρεσία Ασύλου. Και μόνο σε ορισμένε περιπτώσεις εμπλέκονται και άλλες αρχές. Η διαδικασία αίτηση γίνεται με ομοιόμορφη ενιαία αίτηση στη Σουηδία. Έχουμε την καταχώρηση του, της αίτηση, αναζήτηση στο Eurodac και στο VIS και συνέντευξη. Να πούμε εδώ ότι τα πρώτα τρία βήματα της διαδικασίας γίνονται εντός ορισμένων ημερών από την ε, υποβολή της ε, αίτησης ασύλου. Και η συνέντευξη ακολουθεί το άρθρο 5 του κανονισμού του Δουβλίνου. Και αυτή λοιπόν γίνεται πολύ νωρί στη διαδικασία. Και κανονικά είναι η μοναδική περίπτωση όπου υπάρχει τέτα τέτ συνέντευξη του ετούντος ε, πριν ε, την απόφαση, χωρίς της απόβασης. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνέντευξη. Έχουμε καταλήξει σε πολύ καλά οργανωμένα ε, πρότυπα συνεντεύξεων. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντική διαδικασία και για τον ετούντα. Συνήθως η διαδικασία υποβολής της αίτησης ε, ιεραρχείται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες εντός της υπηρεσίας γιατί έχουμε και πολύ αυστηρά πλαίσια χρονικά από τον κανονισμό. Μετά λοιπόν τη διαδικασία της αίτηση, η υπόθεση παραπέμπεται στην ομάδα του Δουβλίνου, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του νόμου. Βάσει των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει κατά το πρώτο στάδιο, η ομάδα Δουβλίνου εξετάζει, ε, προσδιορίζει το αρμόδιο κράτος μέλος, και η Σουηδική ομάδα Δουβλίνου είναι αρμόδια και για τα εισερχόμενα και για τα εξερχόμενα αιτήματα. Μετά την έκδοση της απόφασης μετακίνησης, ε, υπάρχει κοινοποίηση προς τον ενδιαφερόμενο και είναι αρμόδιοι και για την, ε, την οργάνωση και εκτέλεση της μεταφοράς. Μόνο αν ο ε, δηλώσει ότι ε, δεν συμμορφούνται με, την, με τον κανονισμό ή διαφύγει, μόνο τότε εμπλέκεται η αστυνομία. Τώρα, για του ε, ασυνόδευτου ανηλίκου, γιατί διαφέρει ε, κατά τη διαδικασία σε σχέση με αυτού των ανηλίκων. Εν γέννη είναι πιο μακροσκελής και εκτεταμένη, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν, περισσο... ανήλικοι έχουν περισσότερη επαφή με τις ε, υπηρεσίε από ότι ένα ενήλικα και όλοι έχουν και έναν ε, νομικό εκπρόσωπο μαζί του. καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία. Σε περίπτωση αμφιβολία για την ηλικία του ετούντος και δεν έχουμε επίσημε αποδείξει. γίνεται μια αξιολόγηση, μια εκτίμηση τη ηλικία του ετούντος και η μεταναστευτική υπηρεσία έχει την δυνατότητα μαζί και με άλλες ε, αρχές να κάνουν οι ιατρικές ε, διαργασίες εκτίμησης της ηλικία, αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, είναι δύσκολο να τα προλάβουμε όλα αυτά. Και για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, η υπηρεσία μετανάστευσης και ο Δήμος ε, που είναι ε, αρμόδιος για τον ασυνόδευτο ανήλικο εργάζονται από κοινού για την υπόθεση. Αυτά είναι συντομία για τους ε, ανηλίκου. και τώρα η Μαρία θα σας ε, μεταφέρει θετικές και αρνητικές εμπειρίες ε, σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση του ζητήματος. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η εμπειρία μας προκύπτει απευθείας από την ομάδα Δουβλίνου στη Σουηδία δεν είναι μια πολιτική τοποθέτηση για τη Σουηδία, γιατί η ομάδα υπηρεσία μετανάστευσης είναι μια ανεξάρτητη αρχή σε ό,τι έχει να κάνει με την ε, επεξεργασία και διεκπαιρέωση των υποθέσεων. Για το θετικό σκέλος των εμπειριών μας, θα ήθελα να πω ότι η καλύτερη εμπειρία είναι όταν ε, ο κανονισμός του Δουβλίνου λειτουργεί όπως ε, πρέπει να λειτουργεί, ιδίως ό,τι έχει να κάνει με την επανένωση οικογενειών όταν έχουμε συγγενείς που έχουν χάσει επαφή με τους αγαπημένους τους και ε, τους ξαναβρίσκουν. Μια άλλη θετική εμπειρία είναι ο κανόνας της αλυσίδας. Η Σουηδία, όπως και άλλα κρατημέλη, έχει υιοθετήσει αυτόν τον κανόνα Θεωρούμε ότι η εφαρμογή αυτού του κανόνα της αλυσίδας είναι ένα καλό παράδειγμα όταν πολλά κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει επί μιας ε, εύλογης και δίκαιης ερμηνείας ε, των διατάξεων του κανονισμού, παρότι ο ίδιος ο κανονισμός δεν παρέχει ξεκάθαρες κατευθύνσεις. Τώρα, για το αρνητικό σκέλος ή τις προκλήσεις, όπως εμείς θέλουμε να τις αποκαλούμε. Όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι στην Ελλάδα και στη Γερμανία, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ότι ο κανονισμός ε, επιδέχεται πολλών ερμηνεών από τα κρατη και τα εθνικά δικαστήρια. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Για να μιλήσω συγκεκριμένα, είδαμε ότι οι υποθέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων είναι οι πιο δύσκολες ιδίω ό,τι έχει να κάνει με ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στον κανονισμό. Αν ο ανήλικο δεν έχει δώσει διαβατήριο ή άλλα προσωπικά έγγραφα και υπάρχουν αφιβολίε για την δηλωθήσα ηλικία, είναι δύσκολο για εμά να ε, αξιολογήσουμε επαρκώ την ηλικία του εντό του χρονοδιαγράμματο. Επίση, η απόφαση C47-17 του δικαστηρίου έχει καταστήσει πιο δύσκολη την διαδικασία προσδιορισμού της αρμοδιότητας σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί δεν μπορούμε πια να διατηρήσουμε ανοιχτές τις υποθέσεις με το αρμόδιο κράτος μέλος για να εκτιμήσουμε την ηλικία. Είναι δύσκολο επίση να εφαρμόσουμε γενικά την δικαστική αυτή απόφαση, γιατί το δεύτερο κράτο μέλο μπορεί να αποφύγει την ευθύνη, ε, αποφεύγοντα να απαντήσει στο αίτημα. Μία άλλη πτυχή του κανονισμού ε, που είναι δύσκολη για εμά είναι η ε, αποχρέωση παροχή αποδεικτικών στοιχείων, γιατί συνήθω έχουμε προφορικέ δηλώσει και συχνά οι αιτούντε δεν μπορούν να τεκμηριώσουν ε, τις δηλώσεις τους με άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Τα κράτη-μέλη ερμηνεύουν την εγκυρότητα των προφορικών δηλώσεων με διαφορετικό τρόπο και αυτό ε, δυσχεραίνει την διαδικασία προσδιορισμού της ευθύνης. Συχνά έχουμε τέτοια ζητήματα λοιπόν είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε ε, και υπάρχουν πολλές ερμηνείες για την ε, επιλογή του εντούτος να αποχωρήσει από την επικράτεια. Μετά έχουμε το άχθος απόδειξης, ε, στο άρθρο 12.4 για τις θεωρήσεις. Και αυτό είναι δύσκολο σημείο για μας. Μια υποχρέωση για την εφαρμογή του άρθρου είναι ο ετών να έχει αξιοποιήσει την θεώρηση για να εισέλθει στην επικράτεια του κράτους μέλους. Κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι το ετών κράτο μέλο, Η δική του ευθύνη να αποδείξει ότι εισήλθε όντω ε, ο ετών άσυλο με τη θεώρηση στην επικράτεια. Όσο ο ετών άσυλο δεν ε, δείχνει το διαβατήριό του, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό τα περισσότερα κράτη-μέλη θεωρούν ε, λογικό να θεωρήσουν, να υποθέσουν ότι χρησιμοποιήθηκε θεώρηση για την είσοδο στη χώρα. Όλα αυτά δυσκολεύουν τα πράγματα. Μία άλλη διάταξη που είναι πρόκληση για μας είναι το ζήτημα της οικογενειακής επανένωσης, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με το ε, συμφέρον του ανηλίκου. Είναι πολύ δύσκολο να εξετάσουμε υποθέσεις όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους δυο σας, κυρία Λίλι Μπλάτ και κυρία Άξελσον, για τη συνεισφορά σας. Ευχαριστούμε που μας παρουσιάσετε το εθνικό σας στήσιμα και πώς το οργανωμένοι στις εθνικές σας υπηρεσίες. Περνάμε στους επόμενους πανελίστ. Μαρία Μπολόκη από την Ισπανική Υπηρεσία Ασύλου. Και εσείς, αν μπορείτε το πολύ, 10 λεπτά. Παρακαλώ. Καλημέρα να σας παρουσιάσω και την δική μας την πρόπτικη. Σκοπός μου είναι να σας παρουσιάσω κάποιους αριθμούς που ε, εξηγούν την κατάσταση, του πώς έχει το ισπανικό σύστημα. Και να σας εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το ισπανικό σύστημα ασύλου. Ε, μερικούς γενικούς αριθμούς, για να δείτε ότι το 2019 120.000 από τις 720.000 στην Ευρώπη είναι ισπανικές. 139.000 είναι οι ε, παράνομες διελεύσεις και δεν θα πρέπει να λέμε πως όλοι οι αιτούντες άσυλο έχουν φτάσει παρανόμως στη χώρα. Για παράδειγμα, μειώσαμε τις ε, παράνομες εισόδους κατά 50% και παρόλα αυτά είχαμε αύξηση των αιτήσεων της ε, διεθνούς προστασίας πάνω από 100%. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πως έχουμε διαφορετική περίπτωση ε, στη χώρα μας από ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη. Για το Δουβλίνο να σας πω ότι τρέχουν παράλληλα διάφορες διαδικασίες, ε, πιέζεται πολύ το σύστημα και τα αιτήματα και οι φάκελοι του κανονισμού Δουβλίνου αυξήθηκαν κατά 10% το 2019, ενώ οι αιτήσει ασύλου αυξήθηκαν κατά το 100%, το οποίο σημαίνει ότι η κατάσταση δική μας είναι πολύ διαφορετική από ό,τι σε εσάς υπόλοιπους. Και να σας πω πως οι χώρες καταγωγής για μας είναι 90% από τη Λατινική Αμερική. Αυτοί ζητούν προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ισπανία. Κυρίως Βενεζουέλα, Κολομβία, Ονδούρες, Ελ Σαλβαδόρ και Νικαράγουα αποτελούν αυτό το 90% των αιτήσεων. Να μιλήσουμε λοιπόν και για την εφαρμογή του Δουβλίνου και να σας πω πως ακούσαμε τι είπαν οι υπόλοιπε αρχές και σε γενικές γραμμές η εμπειρία μας είναι παρόμοια με την εφαρμογή του κανονισμού, με την διαφοροποιημένη ερμηνεία, με τις ε, διατάξεις περί οικογενειακής επανένωσης που ερμηνεύεται ε, ανάλογα με το κράτος μέλος, ε, τις δυσκολίες με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως τα ασυνόδευτα άτομα ή τα άτομα τα εξαρτώμενα μέλη οικογενειών και έχουμε δυσκολίε επίσης θέματα με την αποδοχή ε, φακέλων από άλλα κράτη-μέλη. Επίσης αναγνωρίζουμε πως υπάρχει και ένα κόστος ε, μεταφοράς που είναι πολύ μειωμένο γενικότερα και στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ισπανία, οπότε θεωρώ πως η δική μας εμπειρία είναι παρόμοια με τα όσα είπαν οι υπόλοιποι εδώ στο πάνελ το να περιορίσουμε τις ε, ροές είναι το βασικό για μας, γιατί έτσι δεν έχουμε δευτερογενείς ροές, κάτι το οποίο ανέφεραν κάποιες αρχές. Και την ώρα που θα σκεφτούμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά στον κανονισμό του Δουβλίνου, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη την, καταγωγή τη δική μας ιστορικά. Δηλαδή, Καταρχήν, έχουμε ε, την ε, αρχή της ευθύνης του, της χώρας πρώτης εισόδου. Αυτό συνέβη ε, τη δεκαετία, την τα τέλη τη δεκαετία του 90, όπου είχαμε πιέσει μεταναστευτικές και είναι κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα. Όμως, όπως είπαν και οι υπόλοιπε αρχές, φτάνει κάποια στιγμή που είτε λόγω της κρίσης του 2015, είτε λόγω της ε, τρέχουσας συγκυρίας που έχουμε κρίση σε αριθμητικό επίπεδο τουλάχιστον, καλό θα ήταν να ξανασκεφτούμε αν αυτή η αρχή που ε, προϋποθέτει μια ισόρροπη ε, είσοδο από όλα τα κράτη-μέλη και μέσω αεροπορικών οδών ε, δεν επιβαρύνει υπερβολικά τις χώρες πρώτης εισόδου που αυτή τη στιγμή μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιβαρύνονται υπερβολικά από την τρέχουσα συγκυρία. Αυτό να το λάβουμε υπόψη προετοιμάζοντας τον επόμενο κανονισμό γιατί είναι, να είναι πιο αποτελεσματική η διεκπερίωση των αιτήσεων χορήγησης ε, προστασίας γιατί Ποιο είναι ο στόχο του Δουβλίνου, να αποφασίζουμε ταχύτητα ποιο είναι το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για μία αίτηση ε, χορήγησης προστασίας, διεθνούς προστατείας, για να προστατεύεται και ο ετών και για να έχουμε μια επεξεργασία ε, αποτελεσματική είτε υπό κανονικέ συνθήκες είτε στη διάρκεια μια κρίση. Άρα λοιπόν για τις χώρες πρώτης εισόδου να σας πω πως γενικότερα θα πρέπει να ε, μην τι επιβαρύνουμε δυσανάλογα ή επιπλέον επειδή ακριβώ γεωγραφικά βρίσκονται στα σύνορα. Αυτό πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Το στοιχείο αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε, γιατί μας έχει ξεπεράσει η πραγματικότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη το 2016 πρότεινε αυτή η κατάσταση να ληφθεί υπόψη και πρότεινε ένα σύστημα κατανομής υποχρεωτικής και ε, ταχύτατης για τους ετούντες ε, διεθνούς προστασίας, ε, λαμβάνοντας υπόψη συνδέσμους που έχουν με διάφορα κράτη-μέλη, οπότε θα μπορούσαν να ζητήσουν να εξεταστεί η αίτησή τους εκεί που έχουν αυτούς τους δεσμούς. Αυτή η γρήγορη και ανάλογη κατανομή των ετούντων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην πρόταση κανονισμού έτσι ώστε να λειτουργεί καλύτερα ο κανονισμός που έχουμε σήμερα. Άρα λοιπόν η εφαρμογή των οικογενειακών ρήτρων με διευρυμένη ερμηνεία, λαμβάνοντας υπόψη αδέλφια, ασυνόδευτους ανηλίκους, τα δικά του ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Οι άλλε ε, ευάλωτες ομάδες θα πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη στις διαδικασίες ε, για να εφαρμόζονται εύκολα και στην πράξη. Γιατί μία από τι που διαπιστώσαμε ήταν ε, η διαφοροποιημένη ερμηνεία των διαφορών διατάξεων που έχουμε στο Δουβλίνο ή η μη η, όμοια ή παρόμοια εφαρμογή. Και για όσους δεν έχουν δεσμούς με ένα κράτος μέλος ή δεν έχουν μείνει στο ο, κράτος μέλος αυτός ή δεν έχουν θεώρηση, δεν έχουν συγγενείς κάπου αλλού, θα έπρεπε να σκεφτούμε στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να τους κατανείμουμε με ισορροπημένο τρόπο και με ισότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σύστημα αντικειμενικό, με στοιχεία προαποφασισμένα, τα οποία θα επιτρέπουν να υπάρχει νομική βεβαιότητα σε κάποιο βαθμό, με μια κατανομή ισόρροπη, ισότιμη ε, μεταξύ κρατών μελών. Δηλαδή, ένα σύστημα μόνιμο, Δηλαδή να δρά και με προληπτικό τρόπο, γιατί δεν θα εφαρμόζεται η εφαρμογή του μόνο σε στιγμές κρίσης. Και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό το σύστημα τούτο να λαμβάνει υπόψη και την εξέταση μέσα σε σύντομη προθεσμία, έτσι ώστε οι διαδικασίες να τρέχουν αποτελεσματικά. Να μην έχουμε ανθρώπους που περάνε πάρα πολύ χρόνο ε, σε αυτή το... Ε, σε αυτή την αοριστία χωρίς να γνωρίζουν τι θα συμβεί ε, στο μέλλον και για αυτούς που φτάνουν ε, στις ακτές μας μέσω θαλάσσιας διάσωσης και αυτοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί, Γιατί ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε, να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που έχουμε και να δούμε πώς μπορούμε να ε, βοηθήσουμε να μην γίνεται και κατάχρηση των ε, διεθνών δατάξεων. Δηλαδή θα πρέπει εδώ και στα πλαίσια της αναθεώρησης ε, των διαδικασιών χορήγησης ασύλου μέσα στο Δουβλίνο να κάνουμε κάτι με κάποιες ρήτρε πιο ε, ε, συγκεκριμένο για τις απορρίψεις και επίσης το τι γίνεται με τις επαναπροωθήσεις. Γιατί έχουμε και αυτή την περίπτωση όπου το ένα κράτος πασάρει το βάρος στο άλλο. Για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα κλειστά κέντρα ε, που θα ιδρυθούν στην Ευρώπη, όπου θα μπορεί να μένει ο κόσμος απεριόριστο χρόνο. Ποια είναι η ευθύνη του κράτου μέλου πρώτη εισόδου. Γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση για το ποιο έχει τη μόνιμη ευθύνη και ποια είναι η ευέλικτη ε, αλληλεγγύη που μπορούμε να δείξουμε εμεί και που έχουμε δείξει εδώ και τέσσερα χρόνια. Έχουμε κάποιο συμπέρασμα. Πώ πρέπει να γίνει η κατανομή. Τι θα γίνει με όλα αυτά τα ζητήματα, τι σημαίνουν οι συνθήκες που έχουμε για την ευθύνη, τη δικαιοσύνη στην κατανομία και την στήριξη των όσων χρήζουν προστασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για το ότι προσπαθήσατε να τα πείτε πάρα πολύ σύντομα και για το όραμα το οποίο παρουσιάσατε βασιζόμενοι στην ισπανική εμπειρία για τη διαχείριση των αιτήσεων ασύλου και για τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά που έχει αυτό το υψηλό ποσοστό νόμιμων διελεύσεων ετούντων άσυλο που έχετε στην Ισπανία, γιατί αυτό είναι διαφορετικό από το τοπίο που περιγράφουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των ετήσεων ε, χορήγησης ασύλου προέρχεται από παράτυπες εισόδους. Θα περάσουμε λοιπόν στο επόμενο Αυτή της συνάντησης και θα ακούσουμε την εκπρόσωπο της, ΕΤΗ της Ιταλίας. Υπεύθυνη της Ιταλικής Υπηρεσίας Δουβλίνου. Ο λόγος εσάς για 10 λεπτά. Ελπίζω να προλάβω σε 9 λεπτά, γιατί και οι προηγούμενοι συνάδελφοι ήδη έχουν ε, περιγράψει μια εικόνα ε, πολύ διεξοδική για το τι προβληματισμοί προκύπτουν από τον κανονισμό του Δουβλίνου που φαίνεται να είναι κοινή για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε μια από τις θεμελιώδει αρχέ που, στις οποίες εδράζεται ο ισχύων κανονισμός του Δουβλίνου. Η αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης ιδίω σε ό,τι αφορά τα αποδεκτικά στοιχεία. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια βάση ε, εμπιστοσύνη για να οικοδομηθούν και να ανθίσουν οι αρχές της αλληλεγγύης και τη συνεργασίας όπως προβλέπονται από τι συνθήκε. Θα έπρεπε να λειτουργεί το νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση και για όλους τους άλλους κανόνε. Οι ιστορικοί λόγοι ήδη έχουν αναφερθεί επαρκώς η σημερινή λοιπόν κατάσταση φαίνεται να είναι μια κατάσταση μεταβατική. Η πολιτική κατάσταση στη Λιβύη, η πολιτική αναταραχή είναι ένα θέμα και είπαμε ότι με τον κανονισμό του Δουβλίνου δεν επιλύουμε πολιτικά προβλήματα, Όμω είναι σαφές ότι οι σημερινές συνθήκες θα πρέπει να μα προβληματίσουν. Θα πρέπει να κοιτάξουμε το ε, απότερο μέλλον και να προσπαθήσουμε να προβάλλουμε τα σημερινά γεγονότα στο τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον και να κοιτάξουμε να υπάρχει μια πραγματική μεταρρύθμιση, γιατί το είπαν και οι Γερμανοί συνάδελφοι πολύ ξεκάθαροι. Ε, υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου. Στην Ιταλία η κατάσταση της υλοποίησης του κανονισμού του Δουβλίνου έχει αλλάξει με τα χρόνια. Γιατί προφανώς υπήρξε μείωση των ροών, των ε, ε, αφήξεων και να θυμίσω ότι τα εξωτερικά μας σύνορα στην Ιταλία είναι αποκλειστικά θαλάσσια. Άρα οι παράτυπες είσοδοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται μόνον διαφελάσεις. Ε, απέναντία στα χερσαία σύνορα, στο βορρά, είναι εσωτερικά σύνορα. Οπότε όλες οι αφήξεις που καταγράφονται κυρίως στα βόρειο-ανατολικά αφορούν περιπτώσεις ετούντων ασύλου που ούτως ή άλλως υπάγονται στο σύστημα Δουβλίνου. Ε, το 2019 και στην Ιταλία η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη, όπως και στην Ισπανία. Είχαμε περίπου 1.500 αφήξεις ε, Όμω όμως είχαμε 40.000 αιτήσεις ασύλου και οι μεταφορές του Δουβλίνου ήταν περίπου λίγο λιγότερες από 6.000. Ε, τι σημαίνει αυτό, ότι υποδεχτήκαμε με το σύστημα υποδοχής μας στην Ιταλία τουλάχιστον το μισό των νέων δικαιούχων βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα κριτήρια που ήδη συζητήθηκαν στον κανονισμό του Δουβλίνου ήδη σήμερα ε, προβλέπουν μια ιεράρχηση των χωρών, δηλαδή χώρα πρώτης εισόδου βάσει του αρθρού 13 τελικά δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Ε, γιατί μετά ε, υπερισχύουν τα άρθρα 7, 8 και ούτω καθεξής. Τελικά ποιο είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που υπόθηκε και προηγουμένως. Η δυσκολία το βάρος της ευθύνης να το χειριστούμε έτσι ώστε να προστατεύσουμε και τους ανηλίκους, ανηλίκους ασυνόδευτους που έχουν διαφορετικά δικαιώματα σε σχέση με την οικογενειακή επανένωση, τα μέλη της οικογένειάς τους που βρίσκονται σε άλλα κράτη-μέλη και ταυτόχρονα η απόδειξη για τους οικογενειακούς δεσμούς. Η εμπειρία μας στην Ιταλία από την εφαρμογή του κανονισμού Βουβλίνου είναι πολύ παρόμοια με αυτή που είχαν οι Έλληνες συνάδελφοι στην Ιταλία. Ε, δηλαδή, πολλοί ήταν αυτοί που ετήθηκαν ε, διεθνή προστασία και είχαν πιστοποιητικά γεννήσεως Αλλά όχι πάντοτε, ήταν η εξαίρεση αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να ζητήσει κανεί ε, έγγραφα που να αποδεικνύουν του οικογενειακού δεσμού. Πολλέ φορέ συμβαίνει μεταξύ ε, γονέων και τέκνων, αλλά είναι δύσκολο να αποδείξει κανεί ε, του οριζόντιου δεσμού και ιδίω αν το μέλο τη οικογένεια διαμένει σε άλλο κάτω μέλο. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να έχουμε υπόψη την αρχή τη αμοιβέ εμπιστοσύνη. Ακριβώ γιατί το να έχουμε ταχείε διαδικασίε κάποιε φορέ θα έπρεπε να μεταφράζεται και σε διασφάλιση μια κοινή ερμηνεία. Κοινή ερμηνεία γιατί και το πρόγραμμα κοινή ερμηνεία του κανονισμού, η πρόθεση αυτή, υπογραμμίστηκε και από του άλλου παρεμβαίνοντε εδώ στο πλαίσιο μιας τέτοιας κατάστασης κρίσης που επίκειται κιόλα, υπάρχει ο κίνδυνος το κάθε κρατος μέλος να έχει την τάση να ερμηνεύει τις διατάξεις όπως το συμφέρει. Χρησιμοθυρικά. Για να το πω έτσι. Ε, και κάποιες φορές πράγματι υπάρχει πρόβλημα, πρόβλημα χρόνου στο πώ ελέγχονται τα αποδεκτικά στοιχεία που πετούνται για του οικογενειακού δεσμού, στο πώ ελέγχεται η ηλικία για του ε, τρίτους, ανηλίκου τρίτων χωρών. Αυτό είναι ένα μαζικό πρόβλημα. Οι απορρίψει, οι αρνήσει λόγω τη τεκμηρίωση, τη ελληπού ε, τεκμηρίωση, είναι ένα πρόβλημα. Ακόμα η χώρα μας Ε, εμπλέκεται σε προσπάθειες διάσωσης στην θάλασσα. Ως προς την ερμηνεία, λοιπόν, είναι πολλές περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τι συμβαίνει μετά από μια διάσωση στη θάλασσα. Είναι παράνομη ή παράτυπη η είσοδο βάση του άρθρου 13 ή όχι. Η αρχή αυτή, όπω υπόθηκε υποθηκε επανειλημμενος και για τη δική μας τη χώρα πρέπει να ε, μείνει πίσω μας, διότι η θέση κάποιων χωρών, η φυσική θέση κιόλα, τις φέρνει πραγματικά σε μια κατάσταση αδυναμίας, επειδή βρίσκονται ακριβώ στα εξωτερικά σύνορα. Και είναι εντελώ άδικη η μεταχείριση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών. Ε, θέλω να διαβεβαιώσω την την κυρία Αριχάβη, η οποία μίλησε πρώτη, ότι το δίκτυο των υπηρεσιών μας προσπαθεί πάντοτε να κοιτάζει και να θυμάται ότι πίσω από τα ταξιδιωτικά έγγραφα, πίσω από τα χαρτιά και την τεκμηρίωση υπάρχουν άνθρωποι ε, αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνονται σοβαρέ προσπάθειε στα κατημέρια για να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε μια κοινή γραμμή. Να ξεπεράσουμε αυτήν την αρχή τη πρώτη εισόδου. Πρέπει να υπάρξει επιτέλου ένα μοντέλο ίση ανάληψη ευθυνών. Να υπάρξει μια ίση κατανομή των ετούντων ασύλων στο, ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Μια αρχή αλληλεγγύη. Μια αλληλεγγύη ε, ε, ε, υπαρκτή ηλικής, όχι μόνο μεταξύ των ετούντων ασύλου και των κρατών πρώτης εισόδου. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την συνεισφορά σας κυρία Σπινέλη. Και τώρα περνάμε απευθείας στην αποτίμηση αυτής της σειράς μαρτυριών από τους υπαλλήλους των εθνικών υπηρεσιών θα έλεγα να ακούσουμε την εισηγήτριά μας, την κυρία Κελέρ και τους σκιώδη μα. Παρακαλώ δύο λεπτά το πολύ και προσπαθήστε αν μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις που θα μας απαντήσουν οι υπάλληλοι των εθνικών υπηρεσιών. Όσο είναι ακόμα μαζί μας, γιατί μετά θα έχουμε και ένα δεύτερο πάνελ. Και θα τους δώσουμε τον χρόνο βεβαίω να απαντήσουν στις ερωτήσει σα. Ε, σας θυμίζω ότι το δεύτερο πάνελ πρέπει να ξεκινήσει 10 και 35. Δύσκολο, αλλά πρέπει να τα καταφέρουμε ε, για να προλάβουμε στις 12.30 και μετά έχουμε και τους συντονιστές. Έχουμε απίστευτα φορτωμένη σε διάταξη και απίστευτη πίεση χρόνου. Παρακαλώ κυρία Κελέρ, τώρα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ειλικρινά τους ε, αρμοδίους και εκπροσώπους ε, των ομάδων Δουβλίνου στα επιμέρους που ε, δέχθηκαν ε, και κατάφεραν να κάνουν αυτές τις ιδιαίτερα εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις υποπίεση χρόνου. Μας δείχνουν όμως μια ολοκληρωμένη εικόνα που λειτουργεί συμπληρωματικά από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Σε τρία σημεία θα ήθελα να σταθώ. Αρκετοί από εσά μίλησαν για διαφορετικέ ερμηνείε των επιμέρους διατάξεων του κανονισμού του Δουβλίνου. Πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, τι προτείνετε για να υπάρχει σύγκληση, να προχωρήσουμε μαζί, να έχουμε πιο κοντινές ε, ερμηνείες που θα τηρούν το πνεύμα περισσότερο από το γράμμα του κανονισμού που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Και εδώ επισημάνατε τον ε, περιορισμένο χρόνο και το δύσκολο, ε, πόσο δύσκολο είναι να αποδείξουμε την ε, ηλικία του ετούντος και, και τα άλλα που αναφέρατε πάλι. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για να υπάρχει καλύτερη μεταχείριση των ανηλίκων. Τέλος, οι Γερμανοί συναδελφοί μίλησαν για το εξωτερικά σύνορα, τις παράνομες διαλέψεις, άλλοι μίλησαν για τους διακινητές για αυτό το ζήτημα. Ε, κάτι το οποίο μπορεί να βρίσκουμε κατά τη διαδικασία υπό τον κανονισμό του Δευλίνου, που μπορεί να μην το είχαμε εντοπίσει στην αρχή κατά την ε, καταχώρηση. Και πάλι υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει, ιδέε, λύσει για να έχουμε καλύτερο έλεγχο των συνόρων, καλύτερη εφαρμογή ε, και του χώρου Σέγγεν και πώ μπορούμε να καταπολεμήσουμε του διακινητέ. Ευχαριστούμε. Πραγματικά είστε εξαιρετικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τον χρονικό περιορισμό. Παρακαλώ, ο κύριος Τουμπέ, ο Σκιώδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ε, ομιλητές για τις ε, παρεμβάσεις τους. Είναι προφανές ότι δεν λειτουργεί καλά το Δουβλίνο σήμερα. Ένα σαφές ζήτημα είναι ότι έχουμε ε, τεράστιο αριθμό δευτερογενών μετακινήσεων. Ένα ερώτημα έχω, γιατί είναι αρκετά σαφές νομίζω. Συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται εναρμόνιση των συστημάτων ασύλου των κρατών μελών και αυτό μάλιστα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Έχω όμως το εξής ερώτημα. Έστω ότι θα τα καταφέρουμε να εναρμονίσουμε τα συστήματα ασύλου μας. Θεωρείτε ότι αυτό φτάνει, αν θέλουμε να αποτρέψουμε τις δευτερογενείς μετακινήσεις, ή πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλες ευρωπαϊκές ενέργειες για να αποτρέψουμε τις δευτερογενείς μετακινήσεις, για να μπορέσει να λειτουργήσει ένας νέος κανονισμός του Βλήνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Μπάρτολο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ακούσαμε όλοι αυτά τα στοιχεία της συζήτηση αυτής και ακούμε ότι το κανονισμό του Δοβλίνου δεν λειτουργεί, τουλάχιστον δεν λειτουργεί καλά. Δεν υπάρχει συντονισμό μεταξύ των 100 μελών. Η υλοποίηση του κανονισμού του Δοβλίνου επίση γίνεται μια προσπάθεια αρμονία, αλλά αυτά τα επιβεβαίωσε και το Συμβούλιο τη Ευρώπη που συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα με την εισηγήτρια, την κυρία Κελέρ. Μιλάμε για οικογενειακή επανένωση. Μιλάμε για το ύψιστο συμφέρον των ανηλίκων και για άλλες δυσκολίες, ε, για περιπλοκότητα, για δυσκολία ερμηνείας και εφαρμογής του κανονισμού του το λέω λοιπόν και υπό την ε, λογική ότι το άρθρο 80 για την, τις συνθήκες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει την αρχή της αλληλεγγύης και της ίσης κατανομής των ευθυνών. Είναι λοιπόν ε, απαραίτητο να υπερβούμε, να ξεπεράσουμε επιτέλους αυτή την αρχή της ευθύνης του πρώτου κάτους εισόδου. Το ακούσαμε εδώ. Ε, και το είπαν οι παρεμβαίνοντε, το είπε και το Ευρωκοινοβούλιο στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Πρόταση μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου που θα πρέπει να ε, προβλέπει ίση κατανομή μεταξύ των κρατών μελών. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί Εφόσον ένα κοινό πρόβλημα δεν ε, ε, αντιμετωπίζεται αυτό το αδιέξοδο και έχει παραμείνει μπλοκαρισμένο δύο χρόνια στο Συμβούλιο των Υπουργών. Νομίζω λοιπόν λύση όλων αυτό και γι' αυτό έχουμε έρθει σήμερα εδώ για να τα συζητήσουμε. Λύση θα ήταν ακριβώς να εγκριθεί, να προωθηθεί αυτό που έχει ζητήσει ήδη από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, το κοινοβούλια. Αυτή επιτέλους η ευλογημένη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Καρέμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους εκπροσώπους των ε, εκπροσώπων των αρχών για τις μαρτυρίες τους. Όπως τα είπε και ο κύριος Μπάρτολο, ε, πράγματι όλοι το ίδιο λένε. Αποτυχία του συστήματος Δουβλίνο 3. Το είπαν όλοι. Από το διαφορετικό μετερίζει τους, ε, διαφορετική ερμηνεία του κανονισμού, έλλειψη αλληλεγγύη. Ε, κακή κατανομή ευθυνών μεταξύ των κατομιλών, ε, προβλήματα με του ασυνόδευτου ανηλίκου. Το είδαμε να μα το λέει πριν από λίγε εβδομάδε ο Έλληνα Υπουργό. Ε, απευθύνει έκκληση στου Ευρωπαίου Υπουργού για την μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Το είδαμε και πώ αντέδρασε η Δημοκρατία τη Πορτογαλία. Εδώ λοιπόν καιρό είναι να αρχίσουμε να ανασκουμπονόμαστε και να συνοδευτούν και από πράξεις τα λόγια μας χθε ε, ε, μετρήθηκε ότι από το Σεπτέμβριο του 2015 είναι 600 τα παιδιά, 640 τα παιδιά που έχασαν τη ζωή του στην ε, Μεσόγειο. Πνίγηκαν. Θυμόμαστε την φωτογραφία εκείνη από το παιδάκι στην παραλία ε, και ε, αυτή δεν θέλω να την ξεχάσουμε. Επίση, όταν μιλάμε για διέλευση, για παράτυπη ή παράνομη διέλευση των σύνορων, τι σημαίνει παράτυπο και παράνομο. Κάποιο που διώκεται, που είναι υπαπειλή, ε, πού να τη θεώρηση για να μπει νομίμω. Θα πρέπει λιγάκι να σκεφτούμε ε, και όλη την, όλο το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε και το πώς ε, το αντιλαμβανόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, καιρός λίγο να κοιτάξουμε και την πράξη. Ευχαριστούμε. Ταρντίνο. Ταρντίνο έπρεπε να έχετε μιλήσει προηγουμένως, αλλά έτσι είχα τον κατάλογο. Σας δίνω το λόγο τώρα. Όχι, δεν μίλησα προηγουμένω Εγώ, εγώ σα ζητώ συγγνώμη, έπρεπε να έχετε μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σε ένα πράγμα συμφωνούμε όλοι προφανώ. Ότι ο κανονισμό χρήζει άμεση μεταρρύθμιση. Ακούστηκαν διάφορε παρατηρήσει επικριτικέ, δυσκολίε εφαρμογή, ερμηνεία και γραφειοκρατικό άρθρο. Ε, οι αριθμοί ήταν ξεκάθαροι. Το είπαν οι μιλητέ μα. Ήθελα απλώ να προσθέσω ότι το 2017 ε, σε σχέση με 700 αιτήσει ε, της ασύλου Μόνο το 13% εξετάστηκαν, 2.100. Ε, ε, Είναι λοιπόν ένα από τα βασικά στοιχεία αυτό που πρέπει να σκεφτούμε, το, η διάσταση της οικογενειακής επανένωσης. Υπάρχει έλλειψη διαλλακτικότητας και ελαστικότητας εδώ, δυσκολίας, να καταλάβουμε τις ε, οικογενειακές ανάγκες και δεσμούς. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τη βασική αρχή, τη βασική αρχή της πρώτης εισόδου. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιούν, να μην το βλέπουν αυτό όσοι μιλάνε για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Πώ μπορεί να είναι υπεύθυνο το κράτο ε, πρώτη εισόδου και πώς θα ε, ε, γίνει πραγματικότητα η αλληλεγγύη, πώς θα υπάρξει μεταρρύθμιση της αρχής της οικογενειακής επανένωση αν συνεχίζει να ισχύει η ευθύνη του κάτω πρώτου εισόδου. Ευχαριστούμε, κυρία Ένστ. Ευχαριστώ. Για το 2011 είδαμε ακριβώς ε, τι έγινε, τι ελπίζαμε με την Αραβική Άνοιξη. Ε, όπως τότε ελπίζαμε να πετύχει, Πάλι και το Δουβλίνο αναλόγω έχει αποτυχεί τελείω. Το ακούσαμε. Γονεί χωρισμένα τα παιδιά του, παιδιά μόνα του. Μετά, το 2015, τέσσερα χρόνια μετά, είχαμε το πρόγραμμα για τη μετανάστευση και το 2017 είχαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο να εμ, περνάει μια πρόταση για τη μετανάστευση που να μην γίνεται καν δεκτή υπήρχαν πολύ καλές ιδέες επιτάπητος και εγώ θα είχα χαρεί πάρα πολύ εάν ένας από τους πανελίστες μας εδώ είχε πει τουλάχιστον μία πρόταση ότι υπάρχει κάτι ως πρόταση ως τώρα που θα μπορούσε κανείς να το πιάσει και να κατευθύνει την ε, μεταρρύθμιση. Εντάξει, μεταρρύθμιση δεν έχει γίνει, δεν έγινε δεκτή η πρότασή μας. Αλλά τέλος πάντων τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, κατανομή. Όλοι είπαν ότι το σύστημα κατανομής πρέπει να αλλάξει. Πρέπει όμως να δούμε τι προτάσεις υπάρχουν στην Ισπανία, την Ιταλία, ε, ε, στα διάφορα κράτη, την Ελλάδα, ε, πώς μπορεί πραγματικά να γίνει η κατανομή των μεταναστών, ποια είναι η δική σας πρόταση. Και μετά βλέπουμε ότι από τις 19 Μαρτίου του 2019 ή μετεγκατάσταση ε, σε συνθήκες απάνθρωπες ή μη εξωπρεπής απαγορεύεται. Εδώ λοιπόν είναι θέμα πώς θα υλοποιηθεί η αρχή αυτή. Και επίσης ήθελα να μου πείτε επειδή πολλοί είναι αυτοί που έχουν ταυτόχρονα αρμοδιότητε και θα έπρεπε να υπάρχει δίκαιη κατανομή των αρμοδιοτήτων είπαμε, και των ευθυνών. Ε, θα πρέπει ποιο κράτος μέλος να αναλαμβάνει την ευθύνη και πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την έννοια της υποβολής αποδεκτικών στοιχείων. Ε, θα πρέπει να γίνεται στα εξωτερικά σύνορα πριν μπουν οι μετανάστες ένα ε, τεστ ε, αποδοχής. Σας υπενθυμίζω, 10 και 35 ξεκινάμε με το δεύτερο πάνελ. Μια μικρή καθυστέρηση, όχι όμως πολύ μεγάλη. Σας παρακαλώ πολύ. Έχω σημειώσει πως έχουμε δύο μέλη που θέλουν να κάνουν επιπλέον ερωτήσεις. Από ένα λεπτό ο καθένας. Η κυρία Γκυγιόν παρακαλώ να ξεκινήσει. Να το πω πολύ γρήγορα γιατί θεωρώ πως όλοι κατανοούν πως η, αρχή, η βασική αρχή που, στην οποία βασίζεται το Δευλίνο ξεκινά από το γεγονός πως όλος οι υπηρεσίες σύλλου και οι διαδικασίες σύλλου στα κράτη-μέλη είναι παρόμοιες. Αυτό Βλέπουμε λοιπόν πως αφενός η αρχή της πρώτης εισόδου δεν λειτουργεί, βλέπουμε πως ο, ο αριθμός των μετακινήσεων είναι πολύ μικρός και αστεία ακριβώς και χρειάζεται να βρει μια λύση το κοινοβούλιο που να περνά από άλλες αρχές. Δεν ξέρω αν εδώ οι ομιλητές μας είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την κατάλληλη θέση για να μας απαντήσουν ή την όρεξη για να μας, να μας απαντήσουν, αλλά τι θα κάνουμε στο Συμβούλιο έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους με, μια άλλη, ε, με έναν άλλο τρόπο, γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο από την αρχή δεν λειτουργήσε ποτέ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Φεράρα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλου του ε, πανελίστε. Θα επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Σε ό,τι αφορά τη χώρα και το κριτήριο τη πρώτη εισόδου. Ε, ένα κριτήριο το οποίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται τόσο πολύ και τελικά γίνεται αυτό που το εφαρμόζουν περισσότερο από όλα όλοι. Με ευνηδίε ε, παρέμβαση των υπευθύνων τη Γερμανία για τη διαδικασία του Δουβλίνου. Λένε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μοντέλο ίση ευθύνη, διότι θα πρέπει να υπάρξουν και διαδικασίε φιλτραρίσματο. Όσοι δεν έχουν δικαίωμα εισόδου να μένουν εκτό. Αυτό πραγματικά μου προκαλεί αμφιβολίε και μου θυμίζει κάτι που είχε αναδειθεί από το κείμενο το οποίο είχε ε, ε, ε, απορριφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2016. Όταν προβλέψουμε μια τέτοια προληπτική αποδοχή, μια ε, πρώτη φάση ε, εξέτασης της αίτησης, ε, όπως αυτό που έλεγε το κείμενο του Ευρωκοινοβουλίου, υπάρχουν πρακτικά προβλήματα. Ε, δηλαδή πώς θα γίνεται αυτός ο έλεγχος και τι διαδικασία θα εφαρμόζεται. Ε, και δικονομικά. Δηλαδή πάλι τα κράτη πρώτη εισόδου αναλαμβάνουν τη δυσκολία να εξετάσουν τις αιτήσει σε πρώτη φάση και να επαναπατρίσουν αυτούς που έρχονται να αιτηθούν άσυλο. Για τις δευτερογενείς τώρα μετακινήσεις, τι πράγμα. Πιο αργά Προσπαθώ να προλάβω το χρόνο τη ομιλία, αλλά να μιλήσω και αργά για τη Γερμανία. Τέλο πάντων. Ε, εδώ λοιπόν οι αμφιβολίε που μου προκύπτουν είναι οι εξή. Είναι πολιτικό το θέμα ε, και νομικό. Δηλαδή, οι Ιταλικές αρχές έχουν εντοπίσει ορθώ, δικαίω κατά την άποψή μου, την αρχή τη αμοιβή εμπιστοσύνη, ε, που πραγματικά λείπει και κάποιε από τι άλλε αρχέ έθεσαν το ζήτημα των διαφορετικών ερμηνεών. Πραγματικά είναι πολιτικό ζήτημα η ερμηνεία των ευρωπαϊκών διατάξεων. Ίσως, αλλά είναι μόνο ε, πολιτικό ή είναι νομικό. Εκεί μπορεί να υπάρχει μια νομική δυσκολία και το θέμα είναι πώ θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Διότι το τελικό δίκαιο προβλέπει την λεγόμενη αυθεντική ερμηνεία, την οποία μπορεί μόνο ο νομοθέτη να την ε, ε, αποφασίσει Αλλά αν υπάρχει ευρωπαϊκή ερμηνεία, πώ θα επιληθεί το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν, έχουμε πέντε εθνικές διοικήσεις στο πάνελ, τις ακούσατε. Είχαμε σχόλια, ερωτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσετε για τα πιο ουσιαστικά σημεία τα οποία σας αφορούν. Στον πρώτο γύρο θα ξεκινήσουμε με εσά, κύριε ε, Καραβία. Μπορείτε να τα πείτε σε ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό, έτσι ώστε να μην καθυστερήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις, πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα για τις δευτερογενείς ε, μετακινήσεις και, δε... και στις διαφορετικές ερμηνείες. Για το θέμα των δευτερογενών μετακινήσεων, εάν πρόκειται να θεωρήσουμε πως συνδέονται με τις ελλείψεις του Δουβλίνου και του κανονισμού του σχετικού, αν αυτό το σενάριο εφαρμοστεί, τότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας κανονισμός Δουβλίνου που να λειτουργεί. Και η θέση μας είναι όσο ο κανονισμός του Δουβλίνου θα, θα λειτουργεί ε, και θα είναι δεκτικό της κρίσης αν υπάρχει στοιχείο δικαιοσύνης. Αν υπάρχει λοιπόν αυτή η ρήτρα δικαιοσύνης ή δίκαιες κατανομής που θα ε, είναι στα θεμέλια της τροποποίησης. Βέβαια, πάντα σε κάθε κανονισμό υπάρχει δυνατότητα ερμηνείας, αλλά παράλληλα υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές και θα πρέπει πάνω σε αυτές να βασίζεται η ερμηνεία που λαμβάνουμε. Δηλαδή, η ανάγκη εξασφάλισης της οικογενειακής ενότητος, η ανάγκη διατήρησης πάντα ε, ως στόχο ε, του συμφέροντος του παιδιού. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών. Δηλαδή να προσθέσουμε στοιχεία που θα διευκρινίζουν το πώς θα χρησιμοποιείται ο κανονισμός στο μέλλον. Αλλά στην εφαρμογή του κανονισμού θα πρέπει να το κάνουμε λαμβάνοντας υπόψη μία αρχή ε, θεμελιωδών αρχών σαν αυτές τις οποίες μόλις ανέφερα. Όπως επίσης και να υπάρχει αμοιβή εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν η γερμανική πλευρά. Κύριε Λέσσερ, κύριε Σίμελφένικ, ένα, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Η εναρμόνιση του συστήματος ασύλου έχει προχωρήσει αρκετά. Πιστεύουμε ότι η εναρμόνιση, η είναι σημαντικότατο στόχος, αλλά δεν φτάνει μόνη της. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα δώσουμε κίνητρα ε, στους ετούντες άσυλο, αλλά και στα κάτι μέλη. Δηλαδή, ε, η διάφορες ε, ασυμμετρίες ε, μεταξύ των κρατών μελών, η επιβάρυνση συγκεκριμένων κρατών μελών, αυτή η έλλειψη ισορροπίας και αυτές οι διαρκείς αντιπαραθέσεις μεταξύ κρατών και οι διαφωνίες δεν μπορεί να συνεχιστούν. Εάν ε, έφευγαν αυτές οι ασυμμετρίες από τη μέση, θα είχαμε πολλά καλά στοιχεία. Θα λύναμε ζητήματα όπως τη δευτερογενούς μετανάστευσης στην Γερμανία η θέση της κυβέρνησης είναι να έχει προτείνει ένα σύστημα κατανομής των ευθυνών. Και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωρίζω ότι έχουμε δει την πρόταση αυτή. Έχουμε κοιτάξει και τις δικές σας απόψεις περί κατανομής των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών και τι εκτιμούμε. Εάν καταφέρνουμε να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα δίκαιης κατανομή των ευθυνών, το πρόβλημα των ε, πολλαπλών και διαφορετικών ερμηνεών θα το αντιμετωπίζαμε εν μέρη. Το θέμα όμω σήμερα είναι το ερώτημα ποιο, ποιο είναι αρμόδιο, δεν απαντάτε. Όταν ακόμα συζητάμε γι' αυτό, το ποιο είναι αρμόδιο, κράτο μέλο, άνθρωπο που πρέπει να το αποφασίσει. Ε, ποιο κράτο μέλο, μάλλον, είναι αδύνατο να το αποφασίσει ένα υπάλληλο από άλλο κράτο μέλο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο σύστημα. Και ευθύ εξ αρχή θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη κατανομή ευθυνών. Το έχει πει η Άζο. Μιλάει κανεί για ε, αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό θα ήταν ίσω ένα σύστημα. Και το Eurodac θα έπρεπε επίσης να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και να φαίνεται ε, από το Eurodac ποιος αναλαμβάνει τι και όχι διαρκώς τα κατημέρια να αντιπαρατήθεται μεταξύ τους. Turn. Mr. Axelson and Mr. Ο Ευχαριστώ. Ναι, ήθελα και εγώ να μιλήσω για το ζήτημα των ε, ερμηνεών του κανονισμού του Δουβλίνου. Κατά πόσο πρόκειται για νομικό ή πολιτικό ζήτημα. Σαφώ και πρόκειται για νομικό ζήτημα, γιατί τα δικαστήριά μα ε, θα ερμηνεύσουν ε, τον νόμο και κανεί άλλο. Γι' αυτό μπορεί να διαφέρουν αυτέ οι ερμηνείε από χώρα σε χώρα. Θα μπορούσε κανεί να θίξει και το ζήτημα τη εναρμόνιση του συστήματο Εγώ πάντα μιλώ βάσει της εμπειρία που έχουμε αποκομίσει στο γραφείο μας, στην υπηρεσία μας και μπορώ να σας πω ότι πράγματι τα διαφορετικά συστήματα ασύλου ε, βοηθούν τους ετούντες να κινούνται από τη μία χώρα στην άλλη. Οι διαφορετικοί κανόνες λοιπόν σίγουρα επηρεάζουν το σύστημα. Ευχαριστώ. Ωραία. Η ε, κυρία Μπολοκή, παρακαλώ. Αν μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν η εναρμόνιση. Να ξεπεράσουμε τη σημερινή κατάσταση λοιπόν μέσω εναρμόνισης και αυτό είναι κάτι το οποίο συμμεριζόμαστε όλοι. Στη δική μας περίπτωση θεωρούμε πως η ευθύνη του κράτους μέλους και το σχετικό κριτήριο με τις γενικές γραμμές που ενέκρινε το Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να είναι μια καλή τακτική, μια προσέγγιση για να κάνουμε μια διαρθρωτική αλλαγή και το σύστημα να είναι πιο αποτελεσματικό τα επόμενα χρόνια και να επιτρέπει να διαχειριστούμε και κρίσεις όταν αυτές ξεσπούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σιμονέλη, Σπινέλη, η κυρία Σιμώνα Σπινέλη διορθώνει ο πρόεδρος. Mm, ναι, και κατά τη δική μου την άποψη, η πρώτη είσοδο είναι ένα κριτήριο που θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μα ω το βασικότερο όλων. Και από τεχνική πλευρά, μια από τι αρχέ που θα πρέπει να εφαρμοστεί για να υπάρξει περισσότερη αμοιβή εμπιστοσύνη θα, είτε, θα ήταν αντιστροφή του βάρου ευθύνη, ε, απόδειξη. Ε, εδώ δηλαδή για περίπτωση οικογενειακής επανένωσης, μόνο εφόσον είναι αντίθετο ή αρνητικό για το συμφέρον του ανηλίκου, θα έπρεπε να μην γίνει η οικογενειακή επανένωση ας πούμε. Τώρα για τις δευτερογενείς ε, μετακινήσεις και μετανάστευση θα πρέπει να κοιτάξουμε το σύστημα υποδοχής, διότι αυτό κάνει όλη τη διαφορά σε σχέση με τις χώρες, που, το ποιες χώρες δηλαδή θέλουν οι περισσότεροι μετανάστες. Το να παραμένει κανείς σε ένα συγκεκριμένο τόπο έχει να μοιάζει πολλές φορές με φυλάκιση. Είναι σαν στέρηση της ελευθερίας. Το θέμα είναι λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθούν τα σωστά κίνητρα και στους μετανάστες για να μπορούν να μετακινηθούν από τη μια χώρα στην άλλη. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας και ευχαριστώ που κάνατε ό,τι μπορούσατε για να απαντήσετε συγκεκριμένα στις ερωτήσεις που τέθηκαν στο πρώτο πάνελ. Πραγματικά σας ευχαριστούμε όλους και τις πέντε υπηρεσίες που πήρατε μέρος στη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμε συνεισφορέ σα. Πραγματικά μα ανοίξατε τα μάτια, ε, μα διαφωτίσατε για τη δουλειά που μα αναμένει. Για να ε, φέρουμε στα σωστά μέτρα τον κανονισμό του Δουβλίνου και τι προτάσει μα. Τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ απευθεία, χωρί καμία καθυστέρηση. Διότι τελειώ δεν πρέπει να προλάβουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους του πανελίστε που πήραν μέρο. Και να περάσουμε αμέσω στο δεύτερο πάνελ. Γιατί έχουμε διάφορες παρουσιάσει, οι οποίες θα γίνουν από τους εμπειρογνώμονε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό θα χαρώ να καλωσορίσουμε του εκπροσώπου εδώ που είναι και οι παίκτε σε αυτή την προσπάθεια της αναλυτικής αξιολόγησης του κανονισμού του Δουβλίνου όπως έχει σήμερα. Εδώ λοιπόν θα ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση που θα μας κάνει ε, η κυρία Κάθριν Γούλαρντ και ο κύριος Σταύρος Παπαγεωργόπουλος ε, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν πώς έχει γίνει η εφαρμογή ε, του EPRS. Θα μας εξηγήσουν λοιπόν η πρώτη ως διευθύντρια και ο δεύτερος ως νομικός σύμβουλος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους εξόριστους και τους πρόσφυγες. Ξέρετε πώς έχουμε καθυστερήσει. Σας παρακαλώ πολύ και έχετε το χρόνο μένει για 10 λεπτά, αλλά αν μας τα πείτε σε 9 ακόμα καλύτερα. Εγώ θα παρουσιάσω εδώ ένα έγγραφο που θα σας παρουσιάσουμε την Παρασκευή και δυστυχώς δεν μπορώ να σας ακοινώσω ε, οποιασδήποτε εκπλήξεις. Είναι μία ε, έρευνα που βασίστηκε σε εντολή που λάβαμε από, την, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, την Κομισιόν και έχει να βασιστεί στις αρχές που έχουμε στη λειτουργία του, του Δουβλίνου δεν ψάχνουμε για εναλλακτικέ διατάξεις, δεν ψάχνουμε για καινούριε αρχές. Στο ερευνητικό αυτό, στην ερευνητική αυτή μελέτη θα σας πω πια σε οποιαδήποτε αξιολόγηση πρέπει να είναι ε, εξειδικευμένοι, γιατί έχουμε κενά στην ενημέρωση για το πώς λειτουργεί το Δουβλίνο και αυτό έχει να κάνει με τις αιτήσει, ε, με τη διάρκεια, με τις αποσύρσεις αιτήσεων, με την ε, διαδικασία και το χρόνο της, ε, των προσφυγών, όπως επίσης και με αποτυχημένες προσπάθειες μετακίνησης. Μετά Μιλήσαμε για την εφαρμογή του Δουβλίνου 3, λαμβάνοντας υπόψη το εργαλειοθήκη για την καλύτερη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλες τις αρχές που καλύπτει, όπως την συνέχεια, τη συνέπεια, την αλληλεγγύη και την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Η μελέτη μας δείχνει πως δεν είναι νομοθετικά αποτελεσματικό ο κανονισμό αυτό γιατί δεν εξυπηρετεί του στόχου που έχουν τεθεί. Ο πρώτο στόχο είναι η ταχεία πρόσβαση στη διαδικασία και όπω είπαν οι και κυρίως, όπως μας είπε η Σάζα, ε, δεν ε, επιτυγχάνεται αυτό. Ο δεύτερος στόχος ήταν ε, να σταματήσουμε τις πολλαπλές αιτήσει. και αυτό που διαπιστώνουμε στη μελέτη είναι πως έχουμε συνέχεια όλο και περισσότερες πολλαπλές αιτήσει. Είναι ένα φαινόμενο που ε, συνεχίζεται και το Δουβλίνο δεν αντιμετωπίζει τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Έχει ε, ένα κυρωτικό χαρακτήρα ο κανονισμός μετά τις μεταρρυθμίσεις του 16, αλλά δεν αντιμετωπίζει τους λόγους για τους οποίους μετακινούνται οι άνθρωποι, που έχει να κάνει με κακές συνθήκες υποδοχής, αλλά και με τις προσπάθειες που κάνουν να επανενωθούν με μέλη της οικογένειας και πολύ περίπλοκους άλλους λόγους. Τρίτον, η ιεραρχία και η ιεράρχηση των κριτηρίων που θέτει ο Δουβλίνο 3 δεν γίνεται απόλυτα σεβαστή και η μελέτη δείχνει πως ε, συχνά γίνεται ένα άλμα ε, προς την αρχή της ε, ε, πρώτης εισόδου ενώ αυτό θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως default. Ο Δουβλίνο 3 μοιάζει να είναι αναποτελεσματικός. Το οικονομικό κόστος είναι υψηλό και μάλλον δυσανάλογο, δεδομένου πως ο βασικός στόχος δεν δεν έχει επιτευχθεί. Το χρηματικό κόστος όμως είναι δύσκολο να το αξιολογήσουμε, τουλάχιστον ένα δις ευρώ το χρόνο, παρόλο που δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και έχουμε μεγάλες επενδύσεις σε μεταφορές και μετακινήσεις που δεν γίνονται από αυτούς που χρησιμοποιούν το σύστημα, Γαλλία και Γερμανία, γιατί τα αιτήματα δεν οδηγούνται τελικά σε μεταφορά ανθρώπων. Και στέλνει διάφορους ανθρώπους σε διάφορες κατευθύνσει με αναποτελεσματικό τρόπο το Δουβλίνο. Επίσης, το ανθρώπινο κόστος. Άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται καταναγκαστικά, συχνές συλλήψεις και άνθρωποι που ζουν ε, σε κάποιο είδου ε, ασάφεια. Καλύτερη λοιπόν νομοθέτηση, καλύτερα κριτήρια, οι στόχοι εξακολουθούν να είναι σωστοί αλλά επειδή δεν υπάρχει κεντρικοποιημένη διαδικασία λήψη απόφαση σε κοινό σύστημα για το άσυλο, είναι ουσιαστικό η νομοθεσία να κατανέμει ευθύνη σε συγκεκριμένο κράτο, το οποίο θα βρίσκεται μέσα στο κεντρικό αυτό σύστημα. Παρ' όλα αυτά, η μελέτη μα και άλλε μελέτε καταλήγουν στο ότι έτσι όπως έχει ο Δουβλίνο 3 αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αμφισβητηθεί. Συνοχή. Αυτό το κριτήριο που είναι το τέταρτο. Είναι ε, αδύναμη η συνοχή με διάφορους τρόπους. Πρώτα απ' όλα εσωτερική συνοχή. Αυτό λείπει. Λόγω των διαφορετικών ερμηνεών των κομβικών άρθρων από τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, συνοχή με τις θεμελιώδεις αρχές. Αδύναμη. Γιατί έχει ελλείψεις και στο σχεδιασμό και στη διατύπωση και στην εφαρμογή. Τρίτον, συνοχή με το κεκτημένο ασύλου. Δεν είναι τέλεια κυρίως λόγω ε, διατύπωσης και ερμηνεών όπου έχουμε ε, διαφορές μεταξύ Δουβλίνου και ε, οδηγίας για το χωρίς ασύλου. Προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, το τελευταίο. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Είναι δεδομένη στο να έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τυποποιημένες προσεγγίσεις στην ευθύνη και στην ε, υποχρέωση τεκμηρίωσης. Όταν έχουμε ένα κοινό σύστημα το οποίο δεν έχει κεντρικοποιημένη ε, κεντρική λήψη αποφάσεων, αυτό χρειάζεται. Όταν υπάρχει και νομοθεσία ε, ευρωπαϊκή, προφανώς υπάρχει ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία όταν αποφασίζεται η εφαρμογή. Αλλά οι αδυναμίε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του Δουβλίνου δημιουργούν ερωτηματικά για το κατά πόσο έχει προστιθόμενη αξία αυτό ο κανονισμό, όπω έχει αυτή τη στιγμή διατυπωθεί. Να καταλήξω με τα εξή συμπεράσματα, τα οποία, στα οποία καταλήξαμε από τη μελέτη την οποία την Παρασκευή θα διαβάσετε με λεπτομέρειε. Θα λέγαμε καταρχήν πως οι αδυναμίες έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό και με την εφαρμογή. Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα καλύτερης εφαρμογής, που είναι η αξιολόγηση που γίνεται από κάποιες αξιολογήσεις καλύτερης νομοθέτησης. Εδώ είναι ο σχεδιασμός της, ε, του νόμου που είναι ε, προβληματικός, είναι ασαφής, είναι άδικος και αφήνει υπερβολικές επιλογές στη χάραξη πολιτικής στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι περίεργο για κανονισμό. Αλλά βέβαια ε, πρόκειται για ένα νομικό μέσο που έχει στόχο να αποφεύγονται τέτοιου είδους προβλήματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στις πολιτικές επιλογές στη στιγμή της εφαρμογής και έχει να κάνει με τις προσπάθειες ελαστιστοποίησης των ευθυνών και αυτό έχει να κάνει με τα όσα είπε η Σάζα. Εφαρμογή λοιπόν, έλλειψη πόρων, διευρυμένη ερμηνεία. Θα πρέπει να καλύψουμε και τον σχεδιασμό του κειμένου και την εφαρμογή. Καλύτερη εναρμόνιση για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Τότε να έχουμε πλήρη συμμόρφωση με την ιεράρχηση που είναι μέσω πολιτικών επιλογών καλύτερες οικογενειακές ε, επανενώσεις, ε, χρήση τεκμηρίων, χρήση άρθρου 16 για τα εξαρτώμενα μέλη, καλύτερη χρήση και μεγαλύτερη του άρθρου 17 που είναι οι ρήτρε διακριτικής ευχέρειας για ε, θέματα οικογενειακών μελών ευρύτερη οικογένεια, μετακινήσεις που βασίζονται βασίζονται σε αιτήματα ε, ε, επαναπροώθησης και κυρίως όταν οι ανθρωπιστικές συνθήκες της χώρας προς τις οποίες ε, μετακινούνται οι άνθρωποι δεν είναι οι κατάλληλες. Επίσης, πολιτική για την αναστολή αυτών των μετακινήσεων ε, όταν έχουμε ε, κατάφερει καταπάτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την αποτελεσματικότητα. Καλύτερο σύστημα υποβολή αναφορών για να καλύπτονται τα κενά στην ενημέρωση και ε, σαφήνεια και κατευθυντήρε γραμμέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συστάσει για τη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ θα καταγράψω πω η δουβλινοποίηση πλέον είναι ρήμα που χρησιμοποιείται ε, ε, σε ευρωπαϊκές χώρες και χρησιμοποιείται και ως επιθετικός προσδιορισμός. Είναι η δούβλο δουβλινοποιημένη. Αυτό είναι ένας χαρακτηρισμός άρχιμος. Μιλάει για ανθρώπους κακομεταχειρισμένους και ταλαιπωρημένους. Η νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για την αναστολή ε, των μετακινήσεων αποδεικνύει πως δεν χρειάζεται συστηματική καταπάτηση δικαιωμάτων. Προτεραιότητα λοιπόν στα δικαιώματα του παιδιού, στο συμφέρον του παιδιού, στην ενημέρωση των ετούντων που λείπει, στην ελαχιστοποίηση των ε, κρατήσεων, στην οικογενειακή επανένωση, όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συγκριθούν με τι έχουμε στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην αξιολόγηση να συμπεριλάβουμε και τους άμεσα εμπλεκόμενους περισσότερη χρήση του άρθρου 17 και τη ρήτρα 1 και, τη, και την διάταξη 1 και τη 2 που είναι οι ανθρωπιστικοί λόγοι. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα όσων μετακινούνται και κυρίως όταν μιλάμε για κοινωνικές σχέσεις, ε, πρόσβαση στην απασχόληση, δικαιώματα κινητικότητα ε, εφόσον χορηγηθεί το καθεστώ και η οικογενειακή επανένωση. Τέλος, συστάσει για την αλληλεγγύη. Χρήση του άρθρου 33 στις δύσκολες περιπτώσεις, προληπτική δράση από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι παράλυση και πολιτικός πανικός που είναι αυτό που είδαμε όταν τα άρθρα αυτά δεν ε, χρησιμοποιήθηκαν. Άρθρο 17 για την κατανομή ευθυνών για συγκεκριμένες ομάδες ε, αφήξεων και τέλος οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα πρέπει να κάνει πιο δίκαιη την κατανομή της και πιο αλληλέγγυη την κατανομή. Διαφορετικά δεν έχει νόημα οποιαδήποτε αναδιάρθρωση. Αυτή ήταν και η κριτική που ασκήσαμε στις προτάσεις του Βλήνο 4. Ξέρουμε πως είναι δύσκολες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, αλλά το να ανεχόμαστε τόσο κακή νομοθεσία για πάντα επίσης είναι προβληματικό. Το Δουβλίνο 3 παραμένει το νομικό πλαίσιο και όσο συμβαίνει αυτό βασιζόμαστε ε, στη συμμόρφωση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και είπα να τονίσουμε την προηγούμενη μελέτη μας και να πούμε πώς το Δουβλίνο 3 μπορεί να είναι πιο ε, σύμμορφο με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στον τρόπο που εφαρμόζεται. Ευχαριστώ. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως ήταν και για, τις, ε, για τους εκπροσώπους των υπηρεσιών. Παρακαλώ, κάνετε ό,τι μπορείτε για να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα. Το λόγο τώρα έχει ο Αλεξάνδρ Δεσσαλού. από την ύπατη αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες και την αντιπροσωπεία της ε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά ζητήματα θα μας παρουσιάσει τα πορίσματα της μελέτης της υποτισαρμοστίας για την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο 3. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο τη τη Αρμοστία στο ΙΕ για του πρόσφυγε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την ε, δυνατότητα που μου δίνει να συμμετάσχω σε αυτή τη συνεδρίαση σήμερα. Δεν είχα τη δυνατότητα να δω την έκθεση ΕΚΡΕ, αλλά με ενδιαφέρον άκουσα την προηγούμενη παρέμβαση γιατί πολλά από τα ευρήματα συνάδουν με τα όσα είχαμε δημοσιεύσει στη δική μας έκθεση, τα οποία, την οποία μπορείτε να βρείτε και στο διαδίκτυο. Σε σχέση με την έκθεσή μας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ε, σκιαγραφίσω τα βασικά πορίσματα, ε, μετά να σταθώ σε κάποιες βασικές συστάσεις και να μιλήσω και για ένα άλλο paper που έχουμε στο τέλος για το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην προσωπική συνέντευξη. Υπάρχουν γενικέ προκλήσει που έχουμε προσδιορίσει και εντοπίσει στην έκθεσή μα, που είναι η έλλειψη ε, διερμηνέων και σωστά ε, καταρτισμένου προσωπικού, περιορισμένοι πόροι στι αρμόδιες εθνικέ αρχές και δημοσιονομικοί περιορισμοί σε ορισμένε περιπτώσεις που επηρεάζουν ε, δευτερεύοντα ζητήματα, βοηθητικές υπηρεσίες όπως είναι η διερμηνία και οι δυνατότητε ε, εκτύπωσης εγγράφων. Ε, υπάρχουν δυσκολίε βέβαια ότι έχει να κάνει με τι αρχέ να παράσχουν πληροφορίε και ενημέρωση. Κάποιε φορέ είναι πολύ περίπλοκε διαδικασίε και δεν μπορούν να τι κατανοήσουν οι ετούντε. Οι συνεντεύξει δεν χρησιμοποιούνται όσο αποτελεσματικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Πιο συγκεκριμένα, δεν δίνεται ε, επαρκή έμφαση στην συλλογή αποδεικτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον σωστό προσδιορισμό της αρμοδιότητας. Και συχνά δεν ε, ε, αναζητούνται αυτές οι πληροφορίες προοπτικά σε ό,τι έχει να κάνει με ε, τις διαδικασίες βλέπουμε έλλειψη ομοιομορφίας, έλλειψη καθοδήγησης και κατάρτισης ε, πάντα προ όφελο ε, του συμφέροντος και έτσι καταλήγουμε σε διαφορετικές προσεγγίσεις. Καθυστερήσεις, ό,τι έχει να κάνει με την χορήγηση εκπροσώπου και ασυνέπειες σε ό,τι έχει να κάνει με την επιμελητία σε διάφορα για την ιχνηλάτηση των μελών τη οικογένεια, πάλι υπάρχουν δυσκολίε, ε, όπω και υπάρχει και η περιορισμένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Πέραν των ε, υποχρεώσεων ε, του Δουβλίνου 3, εντοπίσαμε και άλλα ζητήματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κριτήρια οικογενειακή επανένωση και τη ρήτρα εξάρτηση, η μελέτη μα εντόπισε δυσκολίε όπω η χνηλάτιση μελών οικογενείας που δεν γίνεται όσο θα έπρεπε υψηλά πρότυπα αποδεκτικών στοιχείων και περιορισμένο χρονοδιάγραμμα που επηρεάζει τη δυνατότητα οικογενική επανένωση των ετούντων, ε, καθυστερήσει που αφορούν και τους ανηλίκου και τους ενηλίκους, ε, περιορισμένοι ορισμοί της οικογενείας που περιορίζουν την οικογενική επανένωση και τέλος έλλειψη σαφήνειας σε σχέση με τα κριτήρια ή τα όρια, κατόφλα και διαφορετικές ε, απαιτήσει ε, σε ό,τι έχει να κάνει με την εφαρμογή του άρθρου 16 ρήτρα εξάρτησης. Για τις ε, ρήτρε διακριτικής ευχέρειας ε, βρήκαμε ότι η προσέγγιση γενικά είναι περιοριστική στην πράξη. Υπάρχει έλλειψη κατευθυντήριων γραμμών σε ό,τι έχει να κάνει με την εφαρμογή αυτών των διατάξεων και οι όροι και προποθέσεις ποικίλουν και μπορεί να έχουν και πολιτικές προεκτάσεις. Και πάλι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ε, απαιτήσεων ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία και αυτό είναι ζήτημα. Κάποιες συστάσεις τώρα από πλευρά μας. Ε, κατά τη γνώμη μας, ο κανονισμός του Βουλήνο 3 έχει τη δυνατότητα ε, βραχυπρόθεσμα πριν την μεταρρυθμισή του να βοηθήσει τις οικογένειες να επανενωθούν αρκεί όμω να χορηγηθούν επαρκεί πόροι για τη λειτουργία του, για την υλοποίηση του του και με την περαιτέρω στήριξη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ασύλου. Εντοπίσαμε λοιπόν τα κενά και την έλλειψη εναρμονισμένη προσέγγιση στην εφαρμογή του συστήματο ε, Δουβλίνου, κάτι το οποίο συμβάλλει ε, στην έλλειψη εμπιστοσύνη και των ετούντων άσυλων και των κρατών μελών. Αυτό αντανακλάται με αρνητικό τρόπο και στην εμπιστοσύνη των κρατών μελών με δυσμενείς επιπτώσεις ε, στους ετούντες άσυλο που μένουν ε, ε, ξεκρέμαστε αν θέλετε σε μια μεσοβέζικη κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τον κανονισμό Δουβλίνο 3 και τι ε, ε, ρήτρε διακριτική ευχέρεια, προκειμένου να έχουμε ισχυρότερη οικογενειακή επανένωση. Δεν θέλουμε επιπρόσθετε ε, διατάξει που να αποτρέπουν την οικογενειακή επανένωση. Οι περιορισμένοι και περιοριστικοί ορισμοί των μελών οικογενείας παρεμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του συστήματος και προωθούν τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Πρέπει να στηρίξουμε την οικογενειακή επανένωση. Όταν οι οικογένειε ε, διαφορετικά θα ήταν χωρισμένε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιοποιούν τη διακριτική του ευχέρεια για να διασφαλίζουν την οικογενειακή ενότητα. Ε, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες γέρος, να υπάρχει σωστή χρήση των προσωπικών συνεντεύξεων και προδραστικά να συλλέγονται πληροφορίες που ε, βοηθούν στον προσδιορισμό του αρμοδίου κρατούς μέλους για την εξέταση μια αίτηση ασύλου είναι επιπρόσθετα μέτρα που μπορούν να διευκολύνουν την ε, λειτουργία του συστήματος μακροπρόθεσμα θα μας βοηθήσουν ε, στην ε, διασφάλιση και της ε, τήρησης των υποχρεώσεων του Δουβλίνου από τους ετούντες. Πρέπει λοιπόν οι πληροφορίες να χορηγούνται όσο γίνεται πιο γρήγορα και προφορικός και γραπτός και ακόμα και πριν από την υποβολή της αίτηση. Πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των χωρών που αποστέλουν και δέχονται αιτήματα και αιτούντες για να υπάρχει σωστή μετακίνηση υπό τον κανονισμό δουβλίνων. Πρέπει Έχουμε και την παρουσία επιτετραμένων αξιωματούχων σε άλλα κρατημέλη, το οποίο φάνηκε ότι είναι σημαντικό εργαλείο. Μηχανισμοί ταυτοποίηση θα πρέπει να θεσπιστούν για την ταυτοποίηση των ετούντων με συγκεκριμένε ε, ανάγκε. Να του δίνονται πληροφορίε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. ελεύθερη και ποιοτική νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Αυτό βοηθά στην έγκαιρη ενημέρωση και στη σωστή κατανόηση του συστήματος. Έλλειψη αμοιβαία ε, κατανόηση σε σχέση με τις ε, απαραίτητες ε, αποδείξεις για την τεκμηρίωση των οικογενειακών δεσμών είναι βασικό πρόσκομα στην οικογενειακή ενότητα πρέπει να υπάρχει σωστή συνεργασία ε, για αυτό τον λόγο. Τα παιδιά συχνά βλέπουμε ότι περνούν από μακροσκελείς διαδικασίες χωρίς την απαραίτητη στήριξη. Οι υποθέσει που έχουν να κάνουν με τα παιδιά και την οικογενειακή ενότητα πρέπει να ιεραρχηθούν ω προτεραιότητε. Βλέπουμε στη μελέτη μα ότι υπάρχει ανάγκη θέσπιση των απαραίτητων διαδικασιών και μηχανισμών για να βοηθήσουμε την συνεργασία ε, στις διαδικασίες αυτές βέλτου του ενδιαφέροντο και ηχνηλάτηση ε, και εντοπισμού των μελών οικογενεία. Αυτό υποστηρίζει τις ε, ταχύτερε διαδικασίε και περιορίζει το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος. Ένας θα πρέπει ε, να προσδιορίζεται και να διορίζεται όσο γίνεται πιο γρήγορα μετά την άφηξη του ανηλίκου στο κράτος μέλος. Θα πρέπει να είναι παρόν ο κυδεμόνα σε όλα τα στάδια για να προάγει τα συμφέροντα του, του ανηλίκου. Ήθελα τέλος να αναφέρω ότι έχουμε και ορισμένες συστάσεις εν ώψη του νέου ε, συμφώνου που ε, δημοσιεύσαμε τον Ιανουάριο και το είχατε και εδώ. Βέβαια τα περισσότερα αντίτυπα έχουν φύγει, το οποίο είναι καλό. Μπορείτε όμως να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Είναι λοιπόν μια, ένα νέο έγγραφο το οποίο είναι μελλοντοστραφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πραγματικά πολύ γεμάτη αυτή η αναφορά. Εμείς θα παρακολουθήσουμε το ρόλο της είπα, της Αρμοστίας ε, εδώ και βεβαίως ε, σεβόμαστε πολύ τη δική σας ε, συνεισφορά. Το ίδιο βέβαια ισχύει για κάθε μέλος του πάνελ που έχουμε καλέσει σε τούτη τη συνεδρία και αυτό συμβαίνει και για τους επόμενους. Η κυρία Γιωχάννα Ντάρμενιν από την DG Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Κέλλερ που έχει βοηθήσει στο να οργανωθούν αυτές οι συναντήσεις και να σας υπενθυμίσω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 ξεκίνησε μια αξιολόγηση που οδήγησε στην προτινόμενη ε, μεταρρύθμιση του Δουβλίνου 3, ε, η οποία ακόμα βρίσκεται στο τραπέζι γιατί δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε το κείμενο. Η δική μου παρέμβαση θα βασιστεί σε δύο ε, κυρίως σημεία Καταρχήν, η διακυβέρνηση που γίνεται του υφιστάμενου κανονισμού Δουβλίνου, όπως επίσης και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό και τη λειτουργία του τρέχοντος κανονισμού, βασιζόμενο στην αξιολόγηση και στα στατιστικά. Για το θέμα της διακυβέρνησης, να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 36, έχουμε τη δυνατότητα για διοικητικές ε, ε, διαδικασίες που μπορούν να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη για να διευκολύνουν την εφαρμογή του κανονισμού και κυρίως για την δημιουργία ε, αξιωματικών συνδέσμων ή στην περίπτωση απλούστευσης των διαδικασιών τη εντόμηση των προθεσμιών για τα αιτήματα ε, επιστροφών ε, και μετακινήσεων. Αυτά θα πρέπει να ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό. Από το 2016 και μετά, πέντε τέτοιες ε, διοικητικές διεκπαιρεώσεις ή ε, διαδικασίες έχουν θεσπιστεί. Στα πλαίσια του υφιστάμενου κανονισμού έχουμε την Επιτροπή Άρθρου 34 που ενέκρινε τον κανονισμό των 118 του 14 που ε, ε, ε, αναθεώρησε και επικαιροποίησε τον 1560 του 2003 και πολύ συχνά ε, καλούμε συναντήσεις στα πλαίσια της ομάδας ε, εμπειρογνωμόνων. Είναι η ε, Επιτροπή Επαφών, Contact Committee, για την ερμηνεία, συζήτηση και εφαρμογή του κεκτημένου του Δοβλίνου. Και συγκεκριμένα έχουν άλλες απόψεις μετά από δικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα διάφορα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή αυτή συναντάται σε αιτήσια βάση και καμιά φορά δις το έτος με στόχο να συζητηθούν οι διαφορετικές ερμηνείες και να βρίσκονται λύσεις. Να σας εξηγήσω έχει κατατεθεί μια έκκληση για μεγαλύτερη συνεργασία για τα θέματα τεκμηρίωσης και ανταλλαγών τεκμηρίων μεταξύ κρατών μελών. Θέματα, για παράδειγμα, που συζητήσαμε στην Επιτροπή αυτή ήταν πολλαπλές αιτήσει απόσυρση αίτησης και κατόπιν υποβολή αίτησης σε άλλο κράτος μέλος, δύο αλλεπάλληλε παράνομες διαλέψει συνόρων και οικογενειακή επανένωση. Κάτι το οποίο ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ελλάδος, όπως επίσης και κανόνες εφαρμοστικοί. Στον κανονισμό σήμερα στο άρθρο 37 υπάρχει η διαδικασία ε, συνδιαλλαγής, η συμφιλίωσης για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει μεταξύ κρατών μελών τη στιγμή της εφαρμογής του κανονισμού. Να υπενθυμίσω πως αυτή η διαδικασία μπορεί να κινηθεί κατόπιν ετηματος ενός από τα κράτη-μέλη που συμπεριλαμβάνεται στη διένεξη, αλλά θα πρέπει βέβαια στη χρήση αυτής της διαδικασίας συμφωνήσει και το έτερο κράτος μέλος. Έχουν προσπαθήσει διάφορα κράτη-μέλη να κινήσουν αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί είτε γιατί ατύπως μεταξύ κρατών μελών τα θέματα έχουν ε, επιληθεί, είτε γιατί δεν υπήρξε βούληση από το έτερο κράτος μέλος να μπει στη διαδικασία. Για τη διακυβέρνηση. Η ΕΑΣΟ έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. The issue of governance of the, of the Dublin system για την εφαρμογή του συστήματος διπλίνου με την περιοδική ε, αναθεώρηση της εφαρμογής του ε, κανονισμού, της δημιουργίας των δικτύων ε, μονάδων Δουβλίνου που ήταν χρήσιμα για καλύτερη συνεργασία και διάδοση πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2016 έτσι ώστε να μπορούν άμεσα να επικοινωνούν οι εμπλεκόμενες χώρες και εμπειρογνώμονες να υπενθυμίσω κάποια από τα θέματα που προκύπτουν με την εφαρμογή. Ακούσαμε πολλούς ομιλητές να μιλάνε για την εφαρμογή και το σχεδιασμό και να σας πω πως έχουμε στατιστικά δεδομένα να σας δώσουμε για τις διάφορες διαδικασίες. Κυρίως για την ανάληψη ευθύνης και τα αιτήματα επιστροφής. Συνολικό αριθμό αιτημάτων που έγιναν δεκτά, δηλαδή ανάληψη ευθύνη και επιστροφή. Από τις 28.000 το 2012 φτάσαμε τις 94.000 και κάτι το 2018. Αν δούμε τον αριθμό μετακινήσεων που Έγινα στην πραγματικότητα. Το 12 ήταν 9.000 περίπου, που έφτασε τις 25.000 περίπου το 18. Αν δούμε την κατανομή αυτών των μετακινήσεων, αν τη συγκρίνουμε δηλαδή με τα αιτήματα, έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις από χρόνο σε χρόνο, αλλά ποτέ δεν ξεπέρασε πάνω από το 35% από το 12 και μετά και έφτασε και το 20% το 15%. Για παράδειγμα, το 18% ήταν 26%. Αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσω και αυτό αναφέρθηκε από την ΕΚΡΕ πως θα πρέπει η μετακίνηση να συνδέεται με αίτηση και με άτομο. Αφού ο αριθμός αιτήσεων δεν ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα άτομα, αλλά ένα άτομα μπορεί να αιτηθεί μετακίνηση σε αρκετά κρατημέλη πολλαπλές φορές, πριν κάποιο κράτος μέλος κάνει τη μετακίνηση, τα στατιστικά δεν αποδεικνύουν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων έχουν κάνει πολλαπλές αιτήσει και έχουν οδηγηθεί σε μία μετακίνηση. Αυτό το είπε και κάποιος προηγούμενος ομιλητής. Δεύτερον, κατανομή μεταξύ ε, ετοιμάτων σε ανάληψη ευθύνης και επιστροφής. Καταρχήν έχουμε προβλήματα διαδικαστικών ε, αδυναμιών στα συστήματα των κρατών μελών. Στην επιστροφή, λοιπόν, έχουμε τις περισσότερες διορθώσεις που γίνονται στα πλαίσια του κανονισμού Δουβλίνου. Οι εγκεκριμένα αιτήσει από τις 21.000 το 2012 έφτασαν τις 65.000 το 18 και στις εγκεκριμένε ανάληψεις ευθύνης βλέπουμε πως από 7.000 περίπου το 12 έφτασαν κάτι παραπάνω από 30.000 το 18. Για την κατανομή βλέπουμε πως τα αιτήματα επιστροφής είναι τα 3 τέταρτα περίπου των αιτήσεων που γίνονται. 75% αυτών το 12, 69% αυτών των αιτημάτων το 18. Και Κάτι που θα πω ακόμα. Οι διαδικασίες αυτές έχουν και χρονικές πρεθασμίες οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και για την αίτηση και για την απόκριση και για την εκτέλεση της μετακίνησης. Και αν δεν γίνονται σεβαστές οι προθεσμίες, τότε η αρμοδιότητα μετακινείται στο κράτος μέλος που δεν σεβάστηκε τη χρονική προθεσμία. Οι κανόνες αυτοί κάνουν τις διαδικασίες περίπλοκες και δημιουργούν ε, διενέξεις και διαφορές μεταξύ κρατών μελών, υποσκάπτουν την νομική βεβαιότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος και δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο ε, ε, ενισχύει τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Κάτι το οποίο έχουμε πει συχνά. Για το θέμα της εφαρμογής των μετακινήσεων η αξιολόγηση δείχνει και αυτό το επανέλαβε ένας αριθμός ομιλητών στην αίθουσα, το χρονικό πλαίσιο είναι πολύ διαφορετικό. Φτάνει από τις τρεις μέρες με τις έξι μήνες. Κάποια κράτη-μέλη έχουν θέματα με τα χρονικά όρια γενικότερα και για την αξιολόγηση 20 κράτη-μέλη δήλωσαν οι 18 μήνες που προβλέπονται συνολικά είναι ένα από τα θέματα τα οποία δυσκολεύουν την κατάσταση. Το είπε και ο εκπρόσωπος Γερμανίας νομίζω. Αυτά ως ενημέρωση και τα στατιστικά δεδομένα για το πώς εφαρμόζεται το Δουβλίνο. Για τα κριτήρια ε, κατανομής ευθύνης βλέπουμε πως τα κριτήρια που ευθύνονται περισσότερο για την μετακίνηση είναι διαμονή, θεώρηση και είσοδος, διέλευση δηλαδή, στα εξωτερικά σύνορα, το είπαν σήμερα άλλωστε και πάλι, και οδηγεί σε καταστάσεις όπου οι ετούντες αποφεύγουν τη δακτυλοσκόπηση ε, και ουσιαστικά οδηγούνται σε δευτερογενή μετακίνηση. Για τα αποδεικτικά στοιχεία, γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά το οικογενειακό κριτήριο και ξέρω πως το θέμα της τεκμηρίωσης έχει τεθεί από κράτη-μέλη. Κλείνω εδώ. Ναι, σας παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί πρέπει να περάσουμε στον επόμενο πάνελist. Ο κύριος Ward Λούτεν, που εκπροσωπεί την υπηρεσία υποστήριξης ε, για το Ευρωπαϊκό Άσυλο. Σε 10 λεπτά θα προλάβετε. Ναι, θα προλάβω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγητρία, την κυρία Κελέρ, για την πρόσκληση. Ε, μου ζητήθηκε να παρουσιάσω την ε, υποστήριξη που, προσφέρει ο οργανισμό μα για την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνου 3 με δράσει, κατάρτιση και εκπαίδευση. Γρήγορα, γρήγορα λοιπόν, βάσει του ιδρυτικού μα ε, κανονισμού, ρόλο τη ΕΑΖΟ είναι να ασχολείται με την εφαρμογή του κοινωνικού συστήματο ασύλου, να ενισχύει την ε, συνεργασία των κρατών μελών για το άσυλο και να προσφέρει επιχειρησιακή υποστήριξη στα κράτη-μέλη που υπόκεινται σε ιδιαίτερε πιέσει. Αυτό ακριβώ έχουμε κάνει και σε σχέση με τον κανονισμό του Δουβλίνου. Ε, πιο συγκεκριμένα, Έχουμε δημιουργήσει ένα ε, δίκτυο των υπηρεσιών για το Δουβλίνο, όπου προσπαθούμε να έχουμε αρμονισμένη εξέταση των διαδικασιών για τις αιτήσει ασύλου και το Δουβλίνο. Είναι τουλάχιστον 13 υπηρεσίες, μάλλον 30 υπηρεσίες των καταμελών για το ε, άσυλο, μαζί με τα κράτη-μέλη δηλαδή, Νορβηγία και Λεχτενστάιν και κοιτάζουμε να έχουμε συντονισμό, ανταλλαγή πληροφοριών και των πρακτικών μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών ασύλων, ασύλου στις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης Plus. Δηλαδή. Και αυτό για να ενισχύσουμε και το κλίμα μηδέα εμπιστοσύνη που ακούσαμε και προηγουμένω αναφέρεται. Οι δραστηριότητε στο δικτύο μα ε, ε, προβλέπουν συνεδριάσει των ομάδων, των ομάδων που είναι ομάδες κατεύθυνση των steering groups κάθε δύο χρόνια περίπου, αλλά και θεματικές των εμπειρογνωμόνων για διάφορα ζητήματα, όπως λόγω χάρη τα παιδιά ε, βάσει του κανονισμού Δουβλίνου. Πολλέ φορέ έχουμε διεξοδικέ συζητήσει για το πώ τα κρατη μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα και να αναχαιτήσουν τι διάφορε ε, απειλέ. Επίση, κάτι θέλω να παρουσιάσω ε, λεπτομερέστερα είναι τα πρακτικά μα εργαλεία, όπω ο πρακτικό οδηγό του ΕΑΖΟ για την υλοποίηση του κανονισμού Δουβλίνο 3, ιδίω για τι προσωπικέ συνεντεύξει και τα αποδεικτικά στοιχεία και την αποτίμησή του. Αυτό δημοσιεύθηκε πρόσφατα τον Οκτώβριο του 2019. Και Έχουμε και ένα πρόγραμμα ανταλλαγή πληροφοριών ε, Δουβλίνου για του υπαλλήλου που εργάζονται με τα θέματα του Δουβλίνου και για σκοπού αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έτσι μπορούν οι περιεχόμενοι από τα διάφορα κάτι μέλη να συγκεντρωθούν και να επισκεφθούν την υπηρεσία Δουβλίνου των ε, ε, ομολόγων του σε άλλα κάτι μέλη, να μάθουν από τι ιδέε του, τι καλύτερε πρακτικέ του και να δουν πώ θα πάνε οι άλλοι για να δουν αν και οι δικέ του πρακτικέ είναι κατάλληλε ή όχι. Επίση, κάτι που πρέπει να αναφέρω είναι ο πρακτικό οδηγό για το καλύτερο συμφέρον του παιδιού στι διαδικασίε ασύλου. Το, ε, στο συμφέρον του παιδιού, κάτι που ανέφεραν προηγουμένω και άλλοι ομιλητέ, είναι κάτι που διατίθεται στον ιστοτοπό μα. Η πρακτική αυτή οδηγή για την υλοποίηση του κανονισμού Δοβλίνου 3 συντάχθηκαν από τα κράτη-μέλη και μια ομάδα εργασία, αλλά πήραμε συνεισφορέ και από την ομάδα αναφορά όπου συμμετείχαν και οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολούνται με την πολιτική άκρη. Επίση, ασχοληθήκαμε με την, κοιτάξαμε την πείρα των υπαλλήλων που ασχολούνται με τι διαδικασίε του Δουβλίνου για όσου έχουν πρακτική εμπειρία, ιδίω από προσωπικέ συνεντεύξει. Έχουμε ερωτηματολόγια, checklist για τι πληροφορίε που πρέπει να παρέχονται στον Ετούντα ε, σε σχέση με την αίτηση ασύλου βάσει του κανονισμού Δουβλίνου 3 και τι προσωπικέ συνεντεύξει με του Ετούντε, που είναι μέρος της διαδικασίας. Πολύ σημαντικό επίσης, το ακούσαμε ήδη αρκετά, η αποτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων είναι ένα ζωτική σημασία στοιχείο. και το κοιτάζουμε και αυτό με ιδιαίτερη προσοχή. Επίση, έχουμε εκπαίδευση και κατάρτιση για τα θέματα του Βλήνου. Ιδιαίτερω, έχουμε συναντήσεις ε, εκπαιδευτικές για όσους ε, είναι υπάλληλοι που ασχολούνται με τα θέματα των δικασίων Δουβλίνου και έχουμε και εκπαίδευση για, την, ε, για τον εντοπισμό ενδεχόμενων περιπτώσεων Δουβλίνου για τους υπαλλήλους πρώτης επαφής. Δηλαδή να ξέρουν τι ε, δείγματα να εντοπίζουν για να ε, κοιτάζουν κατά πόσο μια υπόθεση είναι υπόθεση Δουβλίνου σε προκαταρκτικά στάδια. Κάποιε επίση από τι υποθέσει πρέπει να πηγαίνουν στη διαδικασία οικογενειακή παρένωση βάσει του Δουβλίνου. Επίση, οι ασκούμενοι μαθαίνουν καλύτερα πώ να εργάζονται εντό των υπηρεσιών Δουβλίνου για να είναι πιο δίκαιοι και σωστή, ισόρροπη όλη η διαδικασία. Ακόμη, Προσφέρουμε υποστήριξη, επιχειρησιακή υποστήριξη σε τέσσερα κράτη-μέλη, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Μάλτα και την Κύπρο. Αλλά στο πλαίσιο αυτή τη επιχειρησιακή υποστήριξη προσφέρουμε επίση υποστήριξη στα θέματα Δουβλίνου. Στην Ιταλία Έχουμε συνεργαστεί στενά με την υπηρεσία Δουβλίνου και κοιτάζουμε να υποστηρίξουμε την διαχείριση και την ε, ε, τελική εξέταση των αιτήσεων Δουβλίνου. Ε, επίσης, κοιτάζουμε στις υπεύθυνε αρχές τις διαδικασίες Δουβλίνου και τις αιτήσει ασύλου στην Ελλάδα σε σχέση με το Δουβλίνο, προσφορά πληροφοριών στους ετούντας ε, επίσης επίκαιρος εντοπισμός, έγκαιρος εντοπισμός υποθέσεων Δουβλίνου και υποβολή φακέλων υποψηφιότητα στην υπηρεσία Δουβλίνου. Καθώς και οι αιτήσει που φεύγουν από την υπηρεσία της Αθήνα. Τώρα στη Μάλτα και την Κύπρο είναι πολύ πρόσφατο. Ασχολούμαστε με την οικοδόμηση δυνατοτήτων, ε, στέλνοντα εμπειρογνώμονε Δουβλίνου στι ε, τεχνικές υπηρεσίε. Θα πάψω εδώ Νομίζω ότι έχω μένει στα όρια του χρόνου. Απλώ να σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία να παρουσιάσω τι ε, δυνατότητέ μα και την επιχειρηματική μα ε, υποστήριξη για την αναμόνιση των πρακτικών και την σωστή υλοποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε απευθεία στον επόμενο πανελίστ, η κυρία Κάρεν Μέτ, ε, που είναι από το Save the Children. Εσείς ευχαριστώ να κάνετε λίγη υπομονή μερικά λεπτά ακόμα και θα τα καταφέρουμε. Χαίρομαι πολύ που είδα πολύ κόσμο να αναφέρονται στα δικαιώματα των παιδιών, τα, τους ασυνόδευτους ανηλίκους, ανησυχούν για το καλό των παιδιών. Ε, είναι κάποιες φορές πονοκέφαλο το όλο ζήτημα και χάρηκα που ξαναδιάβασα τον κανονισμό Δουβλίνου 3 και πώς ε, ε, εχέγγυα περιλαμβάνονται για την προστασία των παιδιών. Έχει πολεμήσει το Κοινοβούλιο για να έχει τι διασφαλίσει αυτέ και θα συνεχιστεί ο αγώνα. Πρώτα απ' όλα μια επισκόπηση. <clears throat> Ένα στου τρει ετούντε άσυλο που φτάνουν στην Ευρώπη είναι παιδί. Ε, από το 2013 έως 2016 είχαμε 225.000 ε, παιδιά που έφτασαν στην Ευρώπη και από το 2014 έως το 2017 περίπου 30.000 παιδιά μεταναστών που αγνοούνταν από τους αριθμούς αυτούς που είναι λίγο ενδεικτικοί διότι η συλλογή των δεδομένων είναι πολύ δύσκολη, έχει να κάνει με το ποιο κάνει τη συλλογή, πού συλλέγονται, είναι όλα τελείω αποσπασματικά. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που συλλεγονται ειναι ολα τελειω αποσπρωματικα ομως βλεπουμε οτι υπαρχει φτάνουν να αγνοούνται. Ε, εδώ λοιπόν τι κάνουμε στην πράξη και όταν λέω στην πράξη ε, θα σας εξηγήσω λίγο τι βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και πώς όλα αυτά σχετίζονται με το Δουβλίνο από τη στιγμή που φτάνει στα σύνορα ε, ένα παιδί και εργαζόμαστε στα σύνορα της Ιταλίας και της Ισπανίας, την Βοσνία ε, Ζεγοβίνη και την ε, Σλοβενία και σε χώρες που έχουν πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες όπως η Σουηδία και η Γερμανία. Θα σα παρουσιάσω λίγο τι συμβαίνει, διότι όλοι οι υπόλοιποι μίλησαν για οικογενειακή επανένωση. Εγώ όμω θα μιλήσω για το τι συμβαίνει πριν την οικογενειακή επανένωση, στο πρώτο στάδιο. Το πρώτο άτομο που συναντά ένα παιδί, το πρώτο άτομο το οποίο έρχεται σε επαφή είναι ο συνοροφύλακα. Και να πω ότι αυτό είναι σημαντικό, διότι ο συνοροφύλακα παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των παιδιών. Λόγου χάρη, στην Ιταλία βλέπουμε ε, κορίτσια από την Ιγυρία που φτάνουν στην Ιταλία και λένε στους συνηροφύλακες ότι είναι άνω των 18, αυτό τους έχουν πει οι έμποροι να πούνε, ε, τις έχουν καταγράψει ε, φυσικά εσφαλμένα και λανθασμένα και θελημένα ως ενήλικες, προχωρούν την όλη διαδικασία ως ενήλικες, ενώ είναι ξεκάθαρα ανήλικες και θα έπρεπε να τις μεταχειριζόμαστε ως παιδιά. Αυτό δημιουργεί πολλές ε, απειλές εις βάρος τους. Επίση, πρέπει να εγγράφονται σωστά οι άνθρωποι στα σύνορα. Βλέπουμε πολλοί κόσμο να φτάνει στα σύνορα στην Κροατία που δεν έχει την δυνατότητα ούτε καν να εγγραφεί. Και αυτά πιέζουν και προωθούν τα παιδιά στα χέρια των εμπόρων, των λαθρεμπόρων. Είναι σημαντικότατη λοιπόν η δουλειά των σύνοροφυλάκων και τη εγγραφή κατά την άφηξη. Αυτό που κάνουμε τώρα και αυτό που έχει να κάνει με την πρόληψη τη δευτερογενή μετακίνηση, όπω λέγεται. Έχουμε περισσότερου ανθρώπου στα σύνορα. Συνεργαζόμαστε με τα παιδιά, με την αστυνομία για να ξεχωρίσουμε τα παιδιά και τι ευπαθεί ομάδε του πληθυσμού. Συγκεντρώνουμε και προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του. Του εξηγούμε τη διαδικασία προκειμένου να γίνει αντιληπτό. Εξηγούμε την εμπορία ανθρώπων. Εξηγούμε πού είναι τα προβλήματα και απειλέ, τι δικαιώματα έχουν και ε, έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό αυτό. Έχουμε κερδίσει αρκετέ φορέ την εμπιστοσύνη του και έχουμε εμποδίσει την περαιτέρω μετακίνηση. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των παιδιών και που δεν έχει σχολιαστεί ιδιαίτερω, πιστεύω, είναι το θέμα τη εκπροσώπηση ή τη κυδαιμονία. Αυτό καλύπτεται επίση από τον κανονισμό του Δουβλίνου. Δηλαδή, έχουμε δει να υπάρχουν κάποιε σχετικέ βελτιώσει στα θέματα τη κυδαιμονία ε, κάποιο ενήλικο που προστατεύει τα ασυνόδευτα ανήλικα. Κάποιε φορέ όμω έχουμε πάνω από 3.000 και δεν μπορούν να Η Ελλάδα έχει ορίσει ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο για του υπευθύνου ε, ενηλίκου. Αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά κενά και ελλείψει. Ε, Εφαρμόζεται πλημελώ. Στην Ισπανία βλέπουμε πολλά κενά επειδή οι περιφερειακέ κυβερνήσει ασχολούνται με τα θέματα τη κυδαιμονία και ε, τα κέντρα υποδοχή ορίζουν ποιο εκπροσωπεί το παιδί. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα ε, το σύστημα κυδαιμονία ε, είναι διαφορετικό από κράτο μέλο σε κράτο μέλο. Και πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα αυτό, διότι είτε είναι οικειοθελή κυδαιμονία ή επαγγελματική. Είναι ε, ζωτική σημασία για να είμαστε βέβαιοι ότι τα παιδιά προστατεύονται και λαμβάνουν τι σωστέ πληροφορίε. Φανταστείτε όμω ότι είστε παιδί. Τελικά καταλαβαίνετε τη διαδικασία. Έχετε και κυδαιμόνα, κάποιον που σα εκπροσωπεί. Και όλα πάνε καλά αλλά έχετε μέλη της οικογένειάς σας που κατοικούν, διαμένουν σε άλλο κάτω μέλος. Μπορεί να πάρει ένα χρόνο, τα γνωρίζετε όλοι. Μπορεί να πάρει ένα χρόνο να πάει το παιδί στην οικογένειά του τελικά. Πολλοί κόσμοι το σχολείο αυτό όμω. Ε, φανταστείτε τι είναι ένα χρόνο τη ζωή ενό παιδιού. Όταν ήσασταν εσεί παιδιά, σκεφτείτε το, σκεφτείτε τα δικά σα τα παιδιά. Πόσο τεράστιο χρονικό διάστημα είναι ένα χρόνο για τη ζωή παιδιού. Για την παιδική ψυχούλα. Αν πει ο λαθρέμπορο, μπορώ να σε πάω στο παιδί σου, στο, στην οικογένειά σου, συγγνώμη, σε μια εβδομάδα, φυσικά το παιδί θα πει ναι. Ε, γιατί θέλει να πάει στου ανθρώπου που εμπιστεύεται και αγαπάει. Ε, είναι τεράστιο αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο. Έχει διαφορετικέ πιέσει η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Σουηδία. Αλλά ελπίζω ότι αν σκέφτεστε την προστασία των παιδιών, θα σκεφτείτε τη δική του προστασία πρώτη όταν μιλάτε για τα ζητήματα αυτά. Επίση, κάτι που είδαμε και θέλω να το επαναλάβω, είναι σημαντικότατο μέτρο, παρόλο που δεν καλύπτεται από τον κανονισμό Δουβλίνου είναι το σύστημα τη μετεγκατάσταση. Είναι ένα πολύ εξυπηρετικό σύστημα, ακόμη και για τα παιδιά. Ε, το σύστημα που εφαρμόστηκε από του συναδέλφου μα του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, το DAB, έχει επίση φανεί καλό για την μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ε, παιδιών. Ε, όταν σταμάτησε το πρόγραμμα αυτό, είδαμε παιδιά να αρχίζουν να εξαφανίζονται από τα κέντρα μα στην Ιταλία. Αυτού του είδου οι κανόνε, οι κανονισμοί έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνη η Επίτροπο Γιώχανσον ε, μίλησε πολύ για την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών. Είναι πραγματικά σημαντικό αυτό. Διότι αν θέλουμε ο κόσμο να χρησιμοποιεί το ισχύον σύστημα, θα πρέπει το σύστημα ε, να λειτουργεί και να υπάρχει εμπιστοσύνη. Ε, και όσο καλύτερα λειτουργεί, τόσο περισσότερο θα το εμπιστεύονται. Όταν όχι, δεν θα το εμπιστεύονται σημαντικά στοιχεία τώρα για την πρόληψη της εξαφάνισης των παιδιών μεταναστών, το πώ μπορούμε να ε, εντοπίσουμε παιδιά ε, και το αν παιδιά ή όχι ανήκουν στη διαδικασία Δουβλίνου. Υπάρχουν πολλά διασφαλίσει εδώ, εγγυήσει. Ε, στο άρθρο 6, στο άρθρο 8 υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για του ανηλίκου. Είναι στην νομοθεσία όλα. Η υλοποίηση είναι το πρόβλημα. Τι συστήνουμε τώρα να βεβαιωθούμε ότι τα συστήματα προστασία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενδυναμώνονται. Διότι πρέπει να δώσουμε ε, έμφαση και στα σύνορα και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και κυρίω εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το σύστημα για το άσυλο και τη μετανάστευση, ε, το σχετικό ταμείο που παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Οι ε, συνοφύλακε παίζουν σημαντικό ρόλο και για την υλοποίηση του Δουβλίνου πρέπει να είναι σωστά καταρτισμένοι και να μπορούν να παραπέμπουν τον κόσμο στα σωστά συστήματα, να αποταθούν κάπου που θα τους βοηθήσουν. Επίσης, πληροφορίες να είναι ε, ε, φιλικές προς τα παιδιά, για να το πω έτσι. Το αν θα καταλάβουν τις πληροφορίες είναι σημαντικό για να μπορούν τα παιδιά να καταλάβουν τα δικαιώματα που θα έχουν, τότε χρειάζονται προσώπηση και να δουν τι εμπόδια υπάρχουν για την οικογενειακή επανένωση πιστεύω και πιστεύουμε στο Save the Children ότι όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στο να ε, δείξει ο κόσμο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο σύστημα και να λειτουργήσει ευρυθμότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία, κυρία Μέτς. Περνάμε τώρα στον τελευταίο ομιλητή, σε αυτό το δεύτερο κύριο, ο κύριος Φραντσέσκο Μαγιάννη, από το δίκτυο Οδυσσέας. Παρακαλώ, το πολύ 9 λεπτά για να έχουμε μετά χρόνο και για συζήτηση. Έχουμε ακόμα μια ώρα. Ε, το λόγο ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρευρεθώ εδώ. Ε, μου ζητήσατε να παρουσιάσω την υπόθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το κανονισμό Δουβλίνο 3 υπήρξαν τρεις ε, αποφάσεις, 19 συγγνώμη, αποφάσεις που συνδέονται άμεσα και τρεις ακόμα σχετίζονται έμεσα. Ακόμα περισσότερες από ό,τι είχαν να κάνουν με το Δουβλίνο 2 ε, που αφορούσε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο σημαίνει ότι το Δουβλίνο 3 έχει οδηγήσει και έχει γύρει πάρα πολλά ερωτήματα που έχουν φτάσει στο δικαστήριο. Τα ζητήματα που εξέτασε το δικαστήριο έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι και τα πιο τετριμένα τεχνικά ζητήματα ε, του κανονισμού Δουβλίνο 3. Ε, φυσικά δεν υπάρχει ο χρόνο να επισέλθουμε σε λεπτομέρειε για αυτή την ομολογία. Θα προσπαθήσω μόνο να παρουσιάσω τρει ε, σημαντικέ τάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ελπίζω να μου συγχωρήσετε τις ε, τα κενά που θα έχω σε αυτή την παρουσίαση, η λήψη χρόνου. Πρώτον, έχουμε το υψηλό επίπεδο προστασία. Αυτή είναι η πρώτη τάση. Η Κάρεν προηγουμένω είπε πολύ σωστά ότι ο κανονισμό Δουβλίνο 3 προστατεύει πολύ περισσότερο τα δικαιώματα και συμφέροντα των ατόμων από ότι ο Δουβλίνο 2. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην ε, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αναδιατύπωση του 2013. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, τήρησε αυτή την ε, αλλαγή. Έχει αλλάξει τον τρόπο ερμηνεία του συστήματο. Παλιότερα ε, έβλεπε το σύστημα ω ένα σύστημα αλληλεπιδράσεων μεταξύ κρατών μελών μεμονωμένα. Ενώ τώρα ο ετών είναι βασικό παράγοντα στο σύστημα. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση ανάμεσα στο να δίνουμε έμφαση σε εγχέγγυα και δικαιώματα και στην διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, όπως παρουσιάζεται συχνά. Μία από τις βασικές πηγές αναποτελεσματικότητα του συστήματο είναι το γεγονό ότι οι ετούντε ε, εξαναγκάζονται να ακολουθήσουν ένα σύστημα που δεν κατανοούν και ε, πρέπει να τους βοηθήσουμε να ε, συνεργαστούν με το σύστημα. Αυτό θα καταστήσει το σύστημα πιο αποτελεσματικό, όχι πιο αναποτελεσματικό. Δεύτερη τάση που προκύπτει από την ομολογία, πιο ισορροπημένη προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει με την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Υπό το Δουβλίνο 2, ιδίω στην απόφαση Αμπτουλάη, υπήρχε μία ε, επιμονή στο τι σημαίνει αμοιβαία εμπιστοσύνη ε, η αμφισβήτηση της ε, μεταφοράς ή μετακίνησης ε, που να έχει να κάνει με την απόδειξη της συστημικής ανεπάρκειας στο κράτος μέλος, το οποίο οδήγησε σε εντάσεις με, το, με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, γιατί από ό,τι φαίνεται αντιβαίνει στις θεμελιώδεις εγγυήσεις που έχουμε στην πολιτική μας κληρονομιά και είχε την ευκαιρία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διορθώσει αυτή την ε, αδικία στην ε, υπόθεση Αντζάβο για παράδειγμα. Ε, υπάρχουν και επικρίσεις και θετικά λόγια, όμως το δικαστήριο προσπάθησε να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά ζητήματα του Δουβλίνου σε ό,τι έχει να κάνει με την δικαιοδοσία του δικαστηρίου ε, σε ό,τι έχει να κάνει με τούντες που ζουν σε ε, χώρες ε, με ακραία φτώχεια και φεύγουν για να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής. Τρίτον, το δικαστήριο έχει προσπαθήσει να ε, τιμήσει τον νόμο σε περιπτώσεις κρίσης. Και πάλι υπάρχουν επικρίσεις και έπαινοι. Όμως βλέπουμε ότι μια κατάσταση κρίσης δεν επιτρέπει την αλλαγή του νόμου, είτε παράκαμψη του νόμου. Αρκεί να δείτε την υπόθεση Τζαφάρη για να δείτε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι εννοώ. Και σε άλλες υποθέσεις το δικαστήριο ήρθε αντιμέτωπο με ε, διάφορες ε, διαδικαστικές παρακάμψεις και παραθυράκια που εκμεταλλεύτηκαν τα κρατημέλη για να αντιμετωπίσουν ε, δυσκολίες που είχαν ε, σε Ανά πάσα στιγμή όμως πρέπει να τηρούνται οι διατάξει του κανονισμού. Αυτό είναι σαφές. Και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τώρα, όπου υπάρχουν τεράστιε πιέσεις για την συμμόρφωση επιτόπου με τα εγχέγγυα που προβλέπει η νομοθεσία. Γιατί ακούμε ότι υπάρχουν όλα ένα και περισσότερα φαινόμενα αποθήσεων, άτυπων, ανεπίσημων ε, προσεγγίσεων και πρακτικών παρακάμψεων του κανονισμού το μήνυμα που αποστέλει το δικαστήριο όσο μπορεί είναι ότι αυτό δεν συνάδει με το γράμμα και το πνεύμα ε, του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και της σχετικής νομοθεσίας. Φτάνω στις τελευταίες μου παρατηρήσεις. Παρότι μπορεί να ε, φάνηκε ότι έχω σκεγγραφίσει μια ρόδινη εικόνα, αλλά έχω και μόνο 10 λεπτά. Υπήρξαν και κάποια αγκάθια βέβαια στην νομολογία, αλλά ε, συνολικά έχουμε μια θετική συνεισφορά. Δυστυχώ, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο χωρίς επιφυλάξει για την συμβολή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπό τον κανονισμό Δουβλίνο 2. Υπήρξε λοιπόν μια σαφή ε, αλλαγή προσέγγισης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια ερμηνείας και εφαρμογής του Δουβλίνο 3 με πιο ανθρώπινο τρόπο. Και θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στην ε, πρακτική εφαρμογή του κανονισμού σε ό,τι έχει να κάνει με την οικογενειακή ένωση υπό τον κανονισμό του Δουβλίνου. Κάτι ακόμα καθώς το δικαστήριο έχει την ευκαιρία να διευκρινίζει τις διάφορες πτυχές του κανονισμού Δουβλίνου και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάει χρόνια ή και δεκαετίες. Αν δείτε την νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, ε, μας πήρε δεκαετίες να διευκρινίσουμε ορισμένα σημεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό ε, σύστημα οι αιτίε ανεπάρκεια δεν έχει να κάνει μόνο με τι αμφιβολίε προ την ερμηνεία, πάνε πολύ βαθύτερα στην δομή του συστήματο. Έχω ακόμα 3,5 λεπτά, οπότε καλά τα πάω από χρόνο, μπορώ να πω κάτι ακόμα. Μια αντίρρηση που θα μπορούσε να φέρει κανεί είναι εντάξει, θετική η συμβολή του δικαστηρίου, αλλά δεν φτάνει. Χρειάζεται μεταρρύθμιση του συστήματο. Έστω Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα ζητήματα που ακούσαμε για την μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. Σίγουρα θα ήταν καλή κίνηση η μεταρρύθμιση του συστήματος, όμως θα πρέπει να γίνει μια ε, μεταρρύθμιση προς το καλύτερο του συστήματος, να μην κάνουμε τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Και σε αυτό το πλαίσιο να θέσω τα εξή ερωτήματα. Πρώτον, θα μπορούσε να λειτουργήσει κάποιο σύστημα κατανομής των ευθυνών, εάν δεν μπορούμε ακόμα να ε, αποδείξουμε ότι είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε τα κοινά μας πρότυπα. Μήπως είναι άλλη προτεραιότητα η κύρια. Πρώτα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα πριν φέρουμε τον ασθενή και πάλι στο χειρουργείο. Δεύτερον, είμαστε σε θέση να έχουμε ένα σύστημα κατανομής αρμοδιοτήτων που είναι ε, ικανό να λειτουργήσει όταν όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να υποστηρίξουν οικονομικά το κόστος ε, όλων των ετούντων, όταν δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτό το κόστος από κοινού. Αυτοί είναι οι παράγοντες που δίνουν το λάθος κίνητρο σε όσους συμμετέχουν στο σύστημα και δεν επιτρέπουν τη δίκαιη λειτουργία και υλοποίηση του συστήματος του Δουβλίνου. Κάτι άλλο. Ε, ας ξεχάσουμε ότι υπάρχει ε, η μαγική λύση από νομικής άποψης. Πρόκειται η κατανομή των ευθυνών είναι εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα. Δεν μπορούμε να έχουμε την ε, εσφαλμένη αντίληψη ότι με μια νομική διόρθωση θα τα όλα. Εγώ είμαι υπέρ της δίκαιης κατανομής και ισότιμης κατανομής των ετούντων άσυλο στη θεωρία, αλλά το ερώτημα είναι στην πράξη είναι εφικτό κάτι τέτοιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης, όταν έχουμε εκατοντάδε. χιλιάδες ε, πρόσφυγες και πώς θα τους κατανείμουμε στα κράτη-μέλη, ε, χωρίς μάλιστα να μας ενδιαφέρει η συνεργασία τους. Και ένα αφελές ερώτημα για το τέλος, γιατί το ακούσαμε στη συζήτηση. Γιατί είναι σημείο εστίαση οι δευτερογενεί μετακινήσει. Αν δείτε το άρθρο 78 τη συνθήκη, το σημείο εστίαση είναι η Ευρώπη στο σύνολό τη να τιμήσει ε, τις τι υποχρεώσει τη σε ό,τι αφορά τη διεθνή προστασία, να διεκπαιρεώσει τα αιτήματα εγκαίρω, να επιστρέψει όσου δεν, δεν ε, ε, δικαιούνται άσυλο και να ενσωματώσει στην κοινωνία τη αυτούς που το δικαιούνται. Σε αυτή την περίπτωση δεν μας βοηθά καθόλου αυτό το ping-pong μεταξύ κρατών μελών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάνατε ό,τι μπορούσατε. Αλλά πραγματικά υποδείξατε μία σειρά προβλήματα τα οποία τα μέλη τα οποία θα λάβουν τώρα το λόγο θα σχολιάσουν. Η κυρία Κέλλερ, παρακαλώ να ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις παρουσιάσεις. Σας ευχαριστώ για τη συντομία. Σας ευχαριστώ για το ότι είπατε πράγματα συμπληρωματικά. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε τη δυνατότητα να δούμε ολόκληρη την εικόνα που δεν είναι καλή, τα είπατε και τα ξαναείπατε, αλλά να βάλετε ο καθένας το δικό του στοιχείο για να αναλύσουμε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καταλαβαίνω πόσο εκνευριστικό είναι για καθένα σας που είστε εμπειρογνώμονες να πρέπει να τα πούτε τόσο ε, συνεκτικά. Καταρχήν, Ευχαριστώ πολύ το PRS που είναι το εσωτερικό κέντρο ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κάνανε καταπληκτική δουλειά για μια μελέτη που θα εκδοθεί στα τέλη της εβδομάδας και που θα προσθεθεί στην αξιόλογη δουλειά που έχει κάνει η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και που παρουσιάστηκε το 2017 με επιπλέον στοιχεία ε, στο ξεκίνημα του ε, της χρονιάς. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δώσουμε αριθμητικά στοιχεία γιατί πρέπει να σας πω πως τα στοιχεία που έδωσε η Κομισιόν εμένα με σοκάρισαν. Λοιπόν, αν μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία αριθμητικά, μια και δεν έχουμε ε, πρόσφατη αξιολόγηση, μας δώσατε απλώς κάποιες ενδείξεις για, τις, ε, για την ανάληψη ευθύνης και για την επιστροφή. Αριθμητικά στοιχεία σας παρακαλώ πολύ, γιατί αυτό θα ήταν χρήσιμο. Για τη διακυβέρνηση που πολλοί από εσάς ανέφεραν, το να δουλέψουμε μαζί, να υπάρχει εμπιστοσύνη, να έχουμε ανάλυση που θα μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε ένα τον άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ εκπρόσωποι της ΕΑΣΟ. Μπορείτε να μας κάνετε προτάσεις για να πάμε πιο κάτω. Και θα το πω, οι θεματικοί μυρογνώμονε του Δουβλίνου συναντιόνται. Αλλά δύο φορέ το χρόνο δεν είναι σε επιχειρησιακό επίπεδο αρκετό. Για παράδειγμα, εμφανίζεται καινούρια ε, οδός. Ε, ε, επικαιροποιούνται διμερεί συμφωνία. Συμφωνίες. Αλλάζουν οι διαδρομές που ακολουθούν. Μπορούμε να πάμε λίγο πιο μακριά στη συνεργασία, η οποία μοιάζει να είναι έτσι κι αλλιώς πολύ ε, καρποφόρος. Μία φορά το χρόνο φτάνει. Είμαστε στο ρυθμό που θα μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που ακούγονται. Για τη Save the Children και για όλους σας. Είπατε πως υπάρχει το συγκεκριμένο θέμα των ανηλίκων. Είναι το τρίτο από τα τέσσερα σημεία που θέλω να θίξω. Όλοι, όλοι συγκινηθήκαμε από τα όσα είπατε. Κορνέλια, δεν ξέρω αν είσαι εδώ ακόμα, αλλά έχει κινητοποιηθεί ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Δεν το έχετε πει, αλλά ίσως γι' αυτό, παραπάνω από ότι για τα υπόλοιπα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί μιλάμε πια για την προστασία του παιδιού σε κάθε κράτος μέλος και της παιδικής ζωής. Έχετε προτάσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μια πεποίθηση. Ζήτησα από το Ερευνητικό Κέντρο του Κοινοβουλίου να το κάνει, αλλά ακόμα δεν έχουν προλάβει πώς μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τη διαδρομή αυτών των ανθρώπων. Με τις μαρτυρίες που ξεκινήσαμε σήμερα και που μας φώτισαν αρκετά, γιατί κανείς ε, μηχανισμός δεν λειτουργεί αν δεν λάβει υπόψη την πραγματικότητα που είναι αναλόγως με τη χώρα κατογής αρκετά διαφορετική για κάθε άνθρωπο. Τι κινητοποίησε, ποια είναι η οικογενειακή κατάσταση, τι ηλικία είναι, όλα αυτά επηρεάζουν. Ίσως λοιπόν δεν θα μπορούσαμε με τον τρόπο αυτό να είμαστε πιο ρεαλιστικοί σε αυτά που θεσπίζουμε, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία, την κινητοποίηση το κίνητρο, την ανθρώπινη πραγματικότητα, τον χρόνο που χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα ξεκινάει η δουλειά. Και όλες οι προτάσεις για βελτίωση είναι καλοδεχούμενες. E Ευχαριστούμε. Και τώρα εσείς κύριε Τομπέ, ε, του ΕΛΚ, Σκιώδης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τις ε, συνεισφορές σας. Για μας είναι πολύ χρήσιμο να τα βλέπουμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες τα πράγματα. Και πιστεύω ότι εδώ δεν είναι ακριβώς οι ίδιες οι μας, αλλά θέλουμε βεβαίως να γίνουν αλλαγές, γιατί ως πολιτική δουλειά μας είναι να βλέπουμε τα πράγματα θετικά να πω δύο πράγματα. Θέλουμε μια μεταναστευτική πολιτική με έναν κανονισμό του Δουβλίνου που να λειτουργεί καλά αλλά ουσιαστικά θα διακρίνει καλύτερα μεταξύ όσων έχουν δικαίωμα στο άσυλο και αυτών που είναι οικονομικοί μετανάστες. Μπορεί κανείς να τους πει και παράτυπους μετανάστες. Εάν θέλουμε να γίνει αυτή η σοβαρή διάκριση, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με, πρόταση, με την πρόταση να εξετάζονται οι αιτήσει ασύλου απευθεία στα εξωτερικά σύνορα. Θα το θεωρούσατε εξυπηρετικότερο από τη δική σας την προοπτική ο καθένας ή ότι δεν θα λειτουργούσε το σύστημα καλύτερα. Πρώτη ερώτηση για τους ελέγχους, την εξέταση των αιτήσεων απευθεία στα εξωτερικά σύνορα και δεύτερον, Όλοι γνωρίζουμε ότι θα έρθει που να είναι πρόταση νέου συμφώνου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γνωρίζουμε ότι θα γίνει συζήτηση για μεταρρύθμιση του συστήματος ως έχει. Επίσης γνωρίζουμε ότι υπήρχε το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαφορών θεσμικών οργάνων, ιδίως στο Συμβούλιο και κυρίως για την υποχρεωτική ανακατανομή το είδαμε από τις επιστολές ε, των ε, εντολών που έχουν μοιραστεί για την απέτηση περί αλληλεγγύης. Εδώ έχω λοιπόν δύο πολιτικά ερωτήματα και ας πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει προτάσει για νέε μορφέ αλληλεγγύη μεταξύ των 100 μελών από τι δικέ σα διαφορετικέ οπτικέ γωνίε. Πώ θα ορίζατε αυτή την αλληλεγγύη, τι θα ήταν εξυπηρετικό, τι θα σα βοηθούσε. Θα το δέχεστε, θα μπορούσατε να το δεχτείτε αυτό ως πρόταση. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο αντιπρόεδρός μας, ο κύριος Μπάρτολο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όσους παρενέβησαν σε αυτό το δεύτερο πάνελ. Ευχαριστώ για τη δουλειά που γίνεται. Άκουσα αριθμού, στατιστικά στοιχεία πολύ σημαντικά και είναι πολύ καλό για να τα επεξεργαστούμε. Όμω, ε, για την ε, μεταρρύθμιση του Δουβλίνου είδαμε ότι το σύστημα μέχρι τώρα είναι δυσλειτουργικό. Ιδίω ε, στι φάσεις που υπάρχει συγκέντρωση και αύξηση των ροών. Γι' αυτό μια δύο ερωτήσει που στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλο ιδιαίτερο, για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση. Γνωρίζουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρξει μηχανισμό υποχρεωτική ανακατανομή. Αλλά πώ μπορείτε να μα καθησυχάσετε ότι θα υπάρχει μια ισότιμη κατανομή των ευθυνών, έστω και αν δεν υπάρχει αυτό ο μηχανισμό. Και πώ θα αποφύγουμε οι ευθύνε ε, να πέφτουν και να βαραίνουν ε, τι χώρε πρώτη εισόδου. Τι συνέπειες θα προκύπτουν, λέτε, ότι θα υπάρχει μια διαδικασία φιλτραρίσματος, screening των ανθρώπων που φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα. Πώς θα γίνεται αυτό, πώς θα γίνεται προσεκτική εξέταση της κάθε περίπτωσης και πώς θα ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας, πώς δεν θα αποδυναμωθεί η θέση τους. Και τι είναι ότι θα δημιουργηθούν κέντρα κράτησης όπου άντρες, γυναίκες, παιδιά θα περιμένουν μπλοκαρισμένοι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ε, Εξηγήστε μας. Ίσως έχουμε ακόμα χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το δημοκρατικότερο θεσμικό όργανο του κόσμου. Α σκεφτούμε του ιδρυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έδωσαν ένα παράδειγμα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι προσωπική έκκληση από κάποιον που εδώ και 30 χρόνια ασχολείται με τα άτομα αυτά και έχει δει νεκρούς. Έχω κάνει ιατροδικαστική εξέταση χιλιάδων ε, πτωμάτων. Ε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ζήσει ε, φρικαλές καταστάσεις, καταστάσεις που κανείς δεν πρέπει ποτέ να περάσει. Ε, πραγματικά πρέπει να έχουμε και καρδιά κάποιες φορές, να τη χρησιμοποιούμε πότε πότε, γιατί πρέπει να παραμένουμε πάρα πολλά άνθρωποι. αυτή είναι η δική μου έκκληση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος, η κυρία Γκαρντίνο.

Ευχαριστώ. Η εικόνα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μετανάστευση είναι κάπω σαφή. Όλα πάνε καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλληλεγγύη, υπάρχει σωστή υποδοχή, ανακατανομή. Όμω όσα λέγονται γύρω του φαίνεται ότι είναι μια βρώμικη προπαγάνδα. Πρώτα λέμε μεταξύ μα γιατί είμαστε εντό και κλεισμένων θυρών. Η μετανάστευση και η υποδοχή είναι ε, περιπτώσεις με παταγώδεις αποτυχίες. Ο κανονισμός του Δουβλίνου αναθέτει τις ευθύνε και το κόστος σε χώρες όπως η Ιταλία. Χώρες που είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν και να εγγράφουν τους μετανάστες που αποφευάζονται. Εδώ τα είπε και η κυρία Φόντε Λάιεν στην αρχή της θητείας της. Ε, το είπε στις αρχές Σεπτεμβρίου και αυτά θα έπρεπε να έχουν και κάποιες συνέπειες. Στην πράξη, η μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου είναι ω σήμερα μπλοκαρισμένοι. Γιατί οι χώρε αυτέ που είναι τόσο αλληλέγγυε, που έχουν τόσο καλέ προθέσει όπω η ε, Γερμανία, ε, θέλουν να παραμείνει το βάρο στι χώρε πρώτη εισόδου. Ακόμα και η συμφωνία τη Μάλτα ήταν ένα μεγάλο, ε, μια μεγάλη αποτυχία. Η ανακατανομή ίσχυσε μόνο για κάποιε δεκάδε μετανάστε, οι οποίοι ήταν ελάχιστοι και μετά είχαμε και τον χρόνο με τα λιμάνια. Όποιο θέλει να μου εξηγήσει και να μου αποδείξει ότι δεν είναι αλήθεια, να τον ακούσω. Στην Ιταλία όμω με την αλλαγή της κυβέρνησης είδαμε να αυξήνονται 700% οι αφήξει και αποβιβάσεις. Χαίρομαι που σηκώνονται οι συνάδελφοι και φεύγουν. Ε, και αυτή την εβδομάδα αποφασίστε να σταματήσετε την επιχείρηση η Σοφία. Στη Σοφία τα προηγούμενα, χρο... η Σοφία, ε, τα προηγούμενα χρόνια μας έφερε 4.500 μετανάστες τουλάχιστον. Και έχουμε ε, πολύ λίγα ποσά διαθέσιμα γι' αυτό. Έχω λοιπόν τις εξή ερωτήσεις. Δεν θα είχε περισσότερα λογική να ε, περιορίσουμε τις αφήξεις αντί να το στέλνουμε πίσω. Επίσης δεν θα είχε νόημα να γίνεται η έγκαιρη, ο έγκαιρος εντοπισμός των αιτήσεων ασύλου ή τουλάχιστον να ξεχωρίζουμε τους οικονομικούς μετανάστες, να φτιάξουμε χάμπ στη Βόρεια Αφρική και όχι να φτάνουν όλοι ε, ατάκτος στην Ευρώπη. Δεν θα είχε περισσότερο νόημα και λογική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους να πάρει σοβαρά το θέμα της μετανάστευσης και να μην μας κάνει την καλή και αλληλέγγυα που μετά όμως θα τα πετάει τα κόστη και το, ε, το βάρος της υποδοχής σε χώρες όπως η Ιταλία. Ευχαριστούμε κύριε Καρέμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους διάφορους ομιλητές. Να σταθώ και σε ορισμένες έννοιες ε, που αναφέρθηκαν στη μελέτη ΕΚΡΕ, όπως είναι η ελλειπής, η πλημελή ε, συνοχή με τα όσα προωθούνται και με την ε, προβληματική προσέγγιση ότι έχει να κάνει με τον κανονισμό του Δουβλίνου και μας οδηγεί σε αυτό τον όρο, του δούβλενοποιημένους που λέγαμε και προηγουμένως. Θα ήθελα να σταθώ και στα αριθμητικά στοιχεία που μας ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί δεν είναι μόνο νούμερα, είναι άνθρωποι πίσω από τα νούμερα. Περάσαμε από τις 28.000 το 2012 στις 94.000 ε, πρόπερση. Ε, Φαίνεται μια τεράστια... Ένα τεράστιο αριθμό. Αλλά από το 0,00056 πήγαμε στο 0,01% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Ε, ούτε για εισβολή πρόκειται, ούτε για λαοθάλασσα, ούτε για τίποτα άλλο τέτοιο δραματικό που προβάλλεται. Είναι μικρή από 0,018 σε 0,05. Η Ευρώπη μπορεί να κάνει διαφορετικά τα πράγματα από τη σήμερα, με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια, με υπευθυνότητα να υποδεχθεί αυτούς τους ανθρώπους και από το 0,0 να πάμε στο 0,06 σε ό,τι αφορά την ανάληψη ευθύνη. Ήθελα να αναφέρω αυτά τα στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με την κλίμακα του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Ε, στη Γαλλία, για παράδειγμα, να σταθώ μόνο, το 2016, ε, στο πλαίσιο του Δουβλίνου, ε, στείλαμε 1.293 άτομα και υποδεχθήκαμε 1.253. 40 άτομα διαφορά, λοιπόν που υποδεχθήκαμε όλους αυτούς που δεν ήθελαν να έρθουν στην Ευρώπη και απορρίψαμε 1.273 αιτήσει ε, ανθρώπων που ήθελαν να μείνουν στη Γαλλία και δεν τους τα επιτρέψαμε. Και αυτό δείχνει ε, το Δουβλίνο και την έλλειψη ανθρωπιάς του. Τέλος, μιλώ για τα δικαιώματα των ανηλίκων, τα, των παιδιών που πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας, τα δικαιώματα των παιδιών και η ανάληψή τους, η φροντίδα τους. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ένστ. Äh, ναι, άκουσα με προσοχή τον ομιλητή μου από την ε, μετάφραση. Λοιπόν, έχω τις εξής ερωτήσεις. Το μεγάλο θέμα της οικογενειακής επανένωσης. Η οικογενειακή επανένωση είναι στην Γερμανία κάτι που Υποτίθεται ότι υλοποιείται ευρέω. Είναι χιλιάδε αυτοί που έρχονται στη Γερμανία για λόγου ε, οικογενειακής επανένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό όμω, γιατί μιλάμε για το συμφέρον των παιδιών. Τι πρέπει να γίνεται στην οικογενειακή επανένωση, πώ θα πρέπει κατά την άποψή σα να οργανωθεί το νέο σύστημα, τι διευθετήσει να υπάρχουν. Ε, πολλά προτάθηκαν. Εγώ όμω θέλω να μου πείτε νομικώ τι πρέπει να γίνει. Το δεύτερο είναι τα δικαιώματα των προσφύγων. Ε, τα κράτη-μέλη που έχουν το μεγαλύτερο φόρτο και βάρος στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, πρέπει να τα βοηθήσουμε. Ε, θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Τα εξωτερικά σύνορα δεν μπορεί να πιέζονται κατά αυτόν τον τρόπο και να επομίζονται εκείνη την ευθύνη όλοι. Όμως ένα άλλο θέμα είναι το τι γίνεται με τους ε, πρόσφυγες. Οι πληροφορίες, η απομάκρυνση πώς θα πρέπει να ε, ρυθμιστούν αυτά, ώστε να υπάρχει μια σχετική δικαιοσύνη, όχι μόνο ως προς τα κράτη-μέλη που πιέζονται, αλλά και προς τους πρόσφυγες, τους ανθρώπους αυτούς που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Και το τρίτο είναι αυτή η διατύπωση ότι χρειαζόμαστε πρώτερους ελέγχους, φιλτράρισμα, screening στα εξωτερικά σύνορα. Ε, όλοι λένε ότι δεν ξέρω από πού να το πιάσω το θέμα, γιατί δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε, το θεωρείτε σωστό, το θεωρείτε λογικό ε, και εφικτό να υπάρχουν τέτοια έλεγχη και αν το θεωρείτε εφικτό, τι προϋποθέσεις θα πρέπει να υπάρχουν, ε, τι ε, όροι να πληρούνται για να θεωρούμε ότι υπάρχει και ίση μεταχείριση των προσφύγων. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα βλέπω ότι έχουμε κάποιο ακόμα συνάδελφο που ε, θέλει να σχολιάσει. Σας παρακαλώ, κύριε Εντέλη, για ένα λεπτό. Μία σύντομη ερώτηση προς τον κύριο Λούτιν από την ΕΑΣΟ. Έχετε σκοπό να διευρύνετε το κέντρο γνώσης έτσι ώστε να καλύπτει και τους υποψήφιες χώρες από τα Δυτικά Βελκάνια για τους γνωστούς λόγους. Μιλήσατε για την Νορβηγία και για την Ελβετία και όλες οι υπόλοιπες χώρες. Πιστεύω ότι αυτή η πρακτική τεχνική βοήθεια είναι πραγματικά ε, πολύ ενδιαφέρουσα για τις υποψήφιες χώρες, κυρίως ε, επειδή τρέχουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 2024, οπότε καλό θα ήταν ε, να ευθυγραμμιστούν τουλάχιστον με το δικό μας νομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω και κάποιον ακόμα να θέλει να μιλήσει. Ε, ένα λεπτό, όχι παραπάνω, αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαρητήρια στο πάνελ. Ε, χαίρομαι πολύ που υπάρχει και πάλι ε, ομόνοια σε αυτή την Επιτροπή. Στο τέλος η τελευταία παρέμβαση μας είπε ότι πρέπει να έχουμε περισσότερους πρόσφυγες, να τους υποδεχόμαστε καλύτερα. Η κυρία Μέτσα από τους ε, σοσιαλιστές πρώην συνάδελφός μας που αναφέρει ε, την μαζική μετανάστευση ως ένα κύμα... παιδιών και ανηλίκων που έρχονται εδώ ανεσπεράσπιστοι, το 80% είναι νεαροί άντρες. Το έψαξα μάλιστα εδώ στο κινητό μου για να σας τα πω. Για παράδειγμα, ο κύριος Τούφικ Τσέι, Μαροκινός που μένει στην Αμβέρσα. Ε, εκπορνεύει νέες γυναίκες και μάλιστα καταδικάστηκε για το βιασμό μιας 14χρονης και φυλακίστηκε μόλις τρία χρόνια. Στη Γαλλία πέρυσι καταδικάστηκε ε, τον άσυλος για την ε, δολοφονία της Γιωχάννα Μπλάνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστώ. No, no, no. I will ask my... Όχι, όχι, θα θέσω την ερώτησή μου κιόλας στην κυρία Ντεμέτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, ναι. Σωστά φέρομαι. Απλώς παίρνω το δικαίωμα και εκμεταλλεύω το δικαίωμα που έχω να με μιλήσω. Έχω ένα ερώτημα συγκεκριμένα. Ναι, αλλά βλέπω ότι και άλλοι... What are you trying to make a footnote on some... Τι θέλετε να σχολιάσετε κάτι άλλο? Γιατί θέλω να έχω κατά νου τον χρόνο πάντα, έτσι. Θα είμαι πιο σύντομος όμως από εσάς. Ναι, βεβαίως, θα ακούσετε την απάντηση. Πρώτα απ' όλα, Πρόεδρε. Πιστεύω και δεν είμαι σίγουρη και ίσως μπορείτε να το επιβεβαιώσετε πως είναι κατά των κανόνων να έχεις ε, σημαία στο τραπέζι μπροστά σου, οπότε ας αφαιρεθεί. Και δεύτερον θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ, δεν ξέρω ποιος είναι ο κανόνας, διαμαρτύρομαι κατά του συνδέσμου που έγινε μεταξύ, σε σχέση με του συνδέλφου μεταξύ μετανάστευσης και βιασμού γυναικών. Είναι ε, πραγματικά α, απεχθές και είναι και κατά των κανόνων μας. Frau Ernst, you also wanted to comment. The same. Κυρία Ernst, ναι, το ίδιο θέλω να πω κι εγώ. Okay, yes. Well, I am to remind you... Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ακριβώς το ίδιο, όπως και ολομέλεια. Παρακαλώ να συμπεριφέρεστε σωστά, όλοι το κάνουμε. Και το λέει, τα μέλη δεν διακόπτουν και δεν συμπεριφέρονται και δεν σχημονούν και δεν έχουν ε, σημαίες. Θα κάνω την ερώτησή μου, αλλά σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, κατεβάστε το σημαίακι, βγάλτε το σημαίακι. Δεν είναι σημαία το banner στα αγγλικά. Όχι. Σημαίακι είναι. No, please. Please, it's okay. It's okay. Please, please. I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, I mean. You have in mind, you have in mind just... Σας παρακαλώ. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να κάνετε τσαμπουκά και να προκαλείτε και να, να ε, χαλάσετε την ατμόσφαιρα. Σας έχω προειδοποιήσει ξανά και ξανά. Όχι σημαίε. στις κοινοβουλευτικές μας εργασίες και εσείς φέρνετε σημαία εδώ πέρα. Κάνετε ακριβώς αυτό που λέει το άρθρο να μην κάνετε. Τα μέλη δεν θα διακόπτουν την εύρυθμη διεξαγωγή των συζητήσεων. Όχι σημαίε, παρακαλώ. Κάντε ό,τι υπόλοιποι. Να απαντήσω. Όχι, σας παρακαλώ. Έχω δικαίωμα, έχω δικαίωμα. Έχω κάθε δικαίωμα, διότι μπορώ να, ε, θα μπορούσα να φέρω την Ευρωπαϊκή Σημαία και να μην έχω καμία ποινή. Όχι. Ε, διαταράστε την ομαλή διεξαγωγή τη συνεδρίαση. Και δεν είναι κόσμια η συμπεριφορά σα. Παρακαλώ. Περνάμε στον επόμενο μιλητή, ε, ο, και ο κύριος Παναγιώτης. Γκόφας Παναγιώτης. Είμαι μέλο τη Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Σα ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δίνετε. Θα ήθελα να ε, τονίσω δύο-τρία σημεία. Ε, άκουσα όλου του ομιλητέ. Θεωρώ καταρχήν ότι ε, το πρόβλημα το οποίο συζητείτε είναι οι λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, βάζοντας βέβαια τη διάσταση τόσο τη νομική όσο και τη συναισθηματική θα έλεγα. Εκείνο όμως που δεν έχει αποφασιστεί νομίζω ακόμα είναι ότι δεν έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν θέλουμε μετανάστες, εάν χρειαζόμαστε μετανάστες και απλά το αντιμετωπίζουμε ως δεδομένο ότι έχουμε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους μετανάστες τους οποίους έχουμε. Το δεύτερο το οποίο πρέπει σίγουρα νομίζω να αποφασιστεί είναι ποιοι είναι μετανάστες και ποιοι είναι πρόσφυγες. Γιατί συνεχώς κάνουμε έναν διαχωρισμό. Ε, είναι πρόσφυγες δηλαδή αυτός ο οποίος μετακινήθηκε δια της βίας από τη χώρα του λόγω πολέμου, αυτός λόγω κλιματικής αλλαγής, αυτός λόγω οικονομικών συνθήκων ή είναι όλοι αυτοί τελικά ή μήπως τελικά είναι όλοι πρόσφυγες. Νομίζω ότι δεν έχουμε αποφασίσει ποιοι τελικά είναι πρόσφυγες και φυσικά το επόμενο ερώτημα είναι ποιοι έχουν δικαίωμα να παραμείνουν. Διότι λέμε ότι δικαίωμα να παραμείνουν έχουν αυτοί οι οποίοι δικαιούνται να έχουν άσυλο. Ποιοι δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι πρόσφυγες. Μήπως όμως τελικά μπαίνουμε σε έναν κύκλο μέσα στον οποίο δεν μπορούμε να βρούμε τις λύσεις οι οποίες προτάθηκαν σήμερα εδώ πάρα πολύ εύστογα από όλους τους προηγούμενους ομιλητές. Εάν λοιπόν λέμε ότι κάποιος δεν έχει δικαίωμα να παραμείνει και πρέπει να επιστραφεί. Να επιστραφεί πού? Στη χώρα την προηγούμενη από την οποία εισήλθε, για παράδειγμα ενδεχομένως την Τουρκία ή την Αφρικανική χώρα, ή στη χώρα από την οποία έρχεται τελικά. Ποιος θα τον επιστρέψει, η χώρα πρώτης εισδοχής ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε αμέσω. Διότι η χώρα πρώτη εισδοχή αδυνατεί να κάνει συμφωνία, για παράδειγμα, με το Αφγανιστάν, με το Πακιστάν, με άλλε χώρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Okay, now let's, let's, let's try to save... Εντάξει, να κερδίσουμε λίγο χρόνο για να δώσουμε και χρόνο στους ε, ομιλητέ μας να απαντήσουν, όπως είναι και το σωστό. Ξεκινούμε λοιπόν με την ίδια σειρά. η κυρία Γούλαρτ και ο κύριος Παπαγιόργόπουλο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια από τα ζητήματα που μας ε, στρέφουν περισσότερο προς το μέλλον που ενδέχεται να είναι στο σύμφωνο και τι ακριβώς προσδοκούμε. Ξέρουμε ότι ε, εκατοντάδε ΜΚΟ έχουν, μάλλον ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν ε, υπογράψει ένα εγγραφό που αναφέρει ακριβώς αυτό που θέλουμε και εμεί στο σύμφωνο. Μία από τις προτάσεις είναι μία εκτεταμένη υποχρεωτική διαδικασία στα σύνορα που κατά τη γνώμη μα εισάγει σημαντική διαδικασία που θα ήταν άδικη και αναποτελεσματική και θα οδηγούσε σε μαζικές κρατήσεις σε κέντρα στα σύνορα, κυρίως ανθρώπων που δεν μπορούν να επιστραφούν οι αιτίε που δεν μπορούν να επιστραφούν αυτοί οι άνθρωποι έχουν να κάνουν συνήθω με τι χώρε προέλευση. Αυτή η πρόταση για επέκταση ή υποχρεωτική χρήση των συνοριακών διαδικασιών ε, ενισχύει και αυξάνει τι ευθύνε των ε, χωρών που βρίσκονται στα σύνορα. Επιπροσθέτω, θα λέγαμε ότι οι πρόσφυγε ε, θα πληγούν περισσότερο, γιατί εκείνοι είναι που πρέπει να διέλθουν τα σύνορα για να αναζητήσουν προστασία. Αντιθέτω, εμεί προτείνουμε μια έμφαση στη συμμόρφωση με το υφιστάμενο δίκαιο ασύλου, ε, με όλες ε, τις διατάξει πέραν του Δουβλίνου, διαδικασίες ε, ταυτοποίηση και κάλυψη των κενών που έχουμε εντοπίσει. Και έτσι βελτιώνουμε τα πράγματα με τη βελτίωση των διαδικασιών για το Δουβλίνο πρέπει να υπάρξει μια σωστή και εύλογη μεταρρύθμιση της διαδικασίας που θέτει και το ζήτημα της, του επιμερισμού των ευθυνών. Παράλληλα, τα προσωρινά μέτρα αλληλεγγύης και το σχέδιο μετεγκατάσταση που προτείνουμε στο άρθρο 17 για την ανάληψη ευθυνών και αποφάσεις πολιτικής που βασίζονται σε μια συμμόρφωση με βάση τα δικαιώματα. Είναι κάτι το οποίο έχουν αναφέρει πολλοί ομιλητέ προηγουμένω, όπου το περιθώριο διακριτικής ευχέρεια ε, των κρατών μελών μπορεί να τύχει διαφορετικών ερμηνεών. Επιπλέον, ε, με το σύμφωνο μπορούμε να καλύψουμε νόμιμες διόδους ε, ασύλου και μετανάστευσης και μεγαλύτερη έμφαση στην συμπερίληψη με βάση τα δικαιώματα και την ε, πολιτογράφηση των ε, ατόμων αυτών στην Ευρώπη. Καλύτερα να κάνουμε όλα αυτά παρά να αρχίσουμε αυτό το παζάρι με ανεπαρκή μέτρα αλληλεγγύης ε, προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα. Ο κύριος Δεσσαλού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σε σχέση με τα κυρία Σκέλ, φτάσω επί κυρία Κέλλερ για την συμπερίληψη των ε, ατόμων που ε, έχουν βιώματα αυτή τη διαδικασία ασύλου στην Ευρώπη. Στην έκθεσή μα έχουμε συμπεριλάβει πάνω από 100 τέτοιε ε, εμπειρίε ετούντων άσυλων για να βασιστούμε σε συγκεκριμένε αποδείξει. Για το σύμφωνο, θα ήθελα να πω ότι βεβαίω και η Πατιαρμοστία του ΙΕ για του πρόσφυγε θέλει μια ιεράρχηση τη προτεραιότητα τη οικογενειακή επανένωση. Δεύτερον, με βάση και το έγγραφο του Ιανουαρίου για το νέο σύμφωνο. Ούτε εμεί πιστεύουμε ότι οι συνοριακέ διαδικασίε θα πρέπει να είναι υποχρεωτικέ. Εναλλακτικά στι ε, διαδικασίε ε, ε, παραδεκτότητας θα πρέπει να ακολουθήσουμε ταχύτερες διαδικασίες για να εντοπίσουμε τις σωστά τεκμηριωμένες και τις αβάσιμες, τους αβάσιμους ισχυρισμούς προκειμένου να αποφασίζονται τελικά τι, τι μελγελέστε με τις αιτήσει ε, με βάση ε, τα στοιχεία. Και σε άλλο έγγραφο ε, της ΥΠΑ τη Αρμοστία, το Fair and Fast, τα μέσα του 2018 τα αναφέρουμε όλα αυτά. Μπορούμε να τα στείλουμε αν σας ενδιαφέρουν. Για τον επιμερισμό και όχι τη μετατόπιση της ευθύνη, εμείς προτείνουμε τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσανάλογα αυξημένο αριθμό αφήξεων να υποστηριχθούν με μέτρα αλληλεγγύης και να λάβουμε υπόψη μια εργαλειοθήκη που μπορεί να δημιουργηθεί με, τους, με τα είδη υποστήριξη και αλληλεγγύη που μπορούν να δείξει ένα κράτο μέλο σε άλλο, ότι έχει να κάνει με την έρευνα αναζήτηση, το σύστημα ασύλου, οικονομική υποστήριξη στου ευρωπαϊκού οργανισμού και τέλο ενώ μπορεί να έχουμε μέτρα και εσωτερικά και στην εξωτερική διάσταση, είναι σημαντικό η εξωτερική διάσταση να μην ιεραρχηθεί ως προτεραιότητα σε σχέση με τα διευρωπαϊκά μέτρα αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε. Η κυρία Νταρμανίν τώρα. Um, thank you, Chair, and... Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και πάλι ε, κύριε Σιγητά. Θα ήθελα για τα δεδομένα τα οποία σας έδωσα, κυρία Συγήτρια, με συγχωρείτε, ε, μπορώ να τα μοιραστώ με το προσωπικό σας και θα ήθελα να μου πείτε το εξή για να αποκριθούμε σε μία άλλη παρατήρηση. Από το 28.000 στο 94 έχει να κάνει με τις αφήξεις που αυξήθηκαν από το 12 και μετά μέχρι το 18 για την Επιτροπή ε, Επαφών δύο φορές το 15 που είναι καλύτερο το 16 κατέθεσε την πρόταση αναθεώρησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε η περισσότερη δράση ασχολήθηκε με αυτό. Για το μέλλον τώρα, πιστεύω πως γνωρίζετε και εσείς πως ο Αντιπρόεδρος κύριος Χινάς και η Επίτροπος ε, κυρία Γιώχανσεν θα κάνουν ένα γύρο πρωτευουσών στα κράτη-μέλη. Έχουν κάνει τα δύο τρίτα ήδη και έχουν κάνει και διμερείς συναντήσεις και το σχέδιο είναι μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου τις επόμενες εβδομάδες οι συναντήσεις αυτές να κλείσουν είναι σημαντικές για να γίνουν κατανοητές οι θέσεις των κρατών μελών και αυτό προετοιμάζοντας την συμφωνία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή ακόμα να πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Είναι όλο τμήμα των συνεχιζόμενων ε, προβληματισμών, αλλά η συμφωνία αυτή θα αντιμετωπίσει τη μετανάστευση και το άσυλο με σφαιρικό τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το κλειδί. Η αλληλεγγύη η οποία δεν θα αποτελεί απλή εναλλακτική λύση. Αυτά. Και νομίζω αργότερα ο Επίτροπος θα μπορέσει να σας τα πει. B, Mr. παρακαλώ. Η κυρία Κέλλερ μας ρώτησε κάτι για το τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Να διευκρινίσω πως εμείς κάνουμε παραπάνω συνεδριάσεις από αυτές τις δύο. Έχουμε δύο της ε, Διευθύνουσας Επιτροπής ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης τέσσερις θεματικές και συν δύο ε, σειρές ανταλλαγών επισκέψεων. Οπότε πολλά γίνονται, γίνονται και σε τεχνικό επίπεδο με τα κράτη-μέλη. Να σας πω πως προσπαθούμε πολύ συχνά να εστιάζουμε στο τεχνικό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα με τις ε, ε πρακτικές, ε, με τα εγχειρίδια πρακτικών που δείχνουμε. Οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε βγάλει από το 18 θα χρησιμοποιηθούν, είναι πολύ ε, σύντομα για να αξιολογηθούν, αλλά δεν είναι βέβαια δεσμευτικέ αυτές οι κατευθύνσεις που δίνουμε. Συντάχθηκαν βέβαια μαζί με τα κράτη-μέλη, οπότε έχουν κάποιο κύρος και χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Δεν έχουμε εντολή, αλλά μπορούμε να δούμε τα χαλαρά μέτρα. Τώρα, για τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Γίνονται πολλά έργα για την οικοδόμηση θεραμικού στα Δυτικά Βαλκάνια, για τα συστήματα ασύλου και υποδοχής. Βέβαια για το Δουβλίνο δεν δεσμεύονται από τον κανονισμό. Έχουμε λοιπόν τα ε, σχέδια έκτακτων ε, περιστάσεων και στις διαδικασίες ασύλου εν ώψη και της προσχόλησης ε, έχουν κάνει πάρα πολλές προσπάθειες και βελτιώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Save the Children. Σας ευχαριστώ πολύ που ενδιαφέρεστε για τα πραγματικά παιδιά που συναντάμε εμείς κάθε μέρα στη δουλειά μας για το θέμα της αλληλεγγύης. Αυτό που δείχνει η αλληλεγγύη είναι η περαιτέρω εναρμόνιση των συστημάτων. Και αν εναρμονιστείτε προς τα υψηλότερα πρότυπα, αυτό θα βοηθήσει. Ένα εργαλείο είναι το Ταμείο Ένταξης ε, για τους ετούντες άσυλο και για τους μετανάστες. Το Ταμείο δηλαδή για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο, από το οποίο επιστρέφουν πολλές φορές κονδύλια τα κράτη-μέλη γιατί δεν θέλουν να το, το χρησιμοποιήσουν. Να το ανοίξετε στις περιφέρειες, στους Δήμους. Αυτή είναι επιτόπου και αυτή αυξάνουν τα επίπεδα προστασίας. Είναι ένα καλό εργαλείο το Ταμείο αυτό και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το Δουβλίνο 4 έκανε κάποιες καλές προτάσεις για την προστασία των παιδιών με ένα νέο μηχανισμό αλληλεγγύης. Γίνεται δηλαδή επανένωση fast track. Και ένα παράδειγμα που είπα είναι το καθεστώς DUB, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο μετεγκατέστησε παιδιά από την Ιταλία και από την Ελλάδα που είναι μια βέλτιστη πρακτική, γιατί λαμβάνει υπόψη το, ε, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Αυτά για τα παιδιά λοιπόν το να συμπεριλάβουμε τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές στους μηχανισμούς αλληλεγγύης είναι κομβικό. Και το έχουν πει σε πολλές χώρες. Θέλουν να συνεισφέρουν. Ας τους δώσουμε την ευκαιρία. Για την εξωτερική διάσταση και εμεί είμαστε στη Βοσνία, Γοβίνη, στη Σερβία, στην Τουνησία. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο στο να ενισχύσουμε τα συστήματα ε, προστασίας αυτέ τι χώρε. αλλά θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίζουν τους ζητούντε άσυλο. Στη Βοσνία, Γοβίνη ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο. Ελάχιστοι έχουν καταφέρει να μπουν στο σύστημα αίτηση ε, ασύλου, οπότε πρέπει οι χώρε αυτέ να είναι έτοιμε για να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Και μια τελευταία παρατήρηση για τι επιστροφέ, γιατί είναι κάτι το οποίο ε, συζητήσαμε, μιλήσαμε με το Αφγανιστάν και γράψαμε για το τι συμβαίνει με τα παιδιά που τα επιστρέφουν στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, αν πάω εγώ στην ε, χώρα, θα δείτε ότι από το Ιράν και από το Πακιστάν χιλιάδες επιστρέφονται στο Αφγανιστάν και οι σειράξει όλο και ενισχύονται. Αυτέ οι, τρίες, οι τρίτες χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και το να δημιουργήσουμε συστήματα ασύλου για τους που επιστρέφουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτού πραγματικά δεν αποτελεί προτεραιότητα. Αν του επιστρέφουμε εκεί λοιπόν, ε, αυτό να το έχουμε κατά νου. Επίσης υπάρχει και θέμα εθνική κυριαρχία με τι χώρε αυτέ. Σα ευχαριστώ. Ο καθηγητής κ. Μαγιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω από τις παρατηρήσεις της συζήτριας ότι πρέπει εμείς να κατανοήσουμε καλύτερα τη διαδρομή των ε, ατόμων για να λειτουργήσει το σύστημα καλύτερα. Πράγματι, πράγματι. Ξεκάθαρα ναι. Το, ένα από τα προβλήματα του συστήματος του Δουβλίνου είναι ότι έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σχεδόν αυτόματα και σε μαζική κλίμακα. Το σύστημα δεν ε, είναι σωστά εξοπλισμένο δηλαδή για να διαχειριστεί διαφορετικά. Δεν έχει να κάνει με, με τις ομάδες ε, Δουβλίνου ε, εγώ γνωρίζω τους ανθρώπους που λειτουργούν εκεί, κάνουν το παν για να λειτουργεί καλά το σύστημα. Και πράγματι βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία να περνάει τους ανθρώπους μέσα από το σύστημα πολύ γρήγορα και χωρίς δεύτερη σκέψη. Και αυτό δημιουργεί ε, ε, παρεξηγήσεις, δημιουργεί έλλειψη εμπιστοσύνη ε, και ούτω καθεξής. Μετά, τα ερωτήματα που μου που έθιξε ο κύριος Τομπίας ο τον Στομπέ, Μήπως θα βοηθούσε μια εξέταση ε, στα σύνορα να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Να σας πω, αυτή η διάκριση γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου αυτό είναι ο σκοπό τη διαδικασία ασύλου. Το να στείλουμε, να μετακινήσουμε την διαδικασία ασύλου στα σύνορα δεν επιλύει το ζήτημα, απλώ το μετατοπίζει. Και φυσικά μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και πάλι όμω θα έχουμε προκλήσει. Πώ θα αποτρέψουμε τις μαζικές ε, κρατήσεις σε πολύ άσχημες συνθήκες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από πλευράς δηλαδή υλικοτεχνικής υποδομής δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε ότι δεν θα καταντήσουμε κάπως έτσι. Δεύτερον, ποιος αναλαμβάνει το κόστος. Προτείνουμε οι χώρες στα σύνορα να επομιστούν όλο το κόστος της διαδικασίας ασύλου στην Ευρώπη. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μήπως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει αυτό το κόστος. Και πάλι όμως αυτό ενέχει πολύ σημαντική δουλειά. Και τέλος, τι γίνεται με αυτούς που χρήζουν προστασίας, πού θα πάνε, πώς επιλέγουν πού θα πάνε, επιλέγουν πού θα πάνε ή απλώς μετακαθίστανται κάπου που δεν γνωρίζουν καν ε, και δεν γνωρίζουν καν που πάνε. Ε, δεν λύνει κάτι λοιπόν αυτό, δημιουργεί και γύρει πολλά ερωτήματα και ανάλογα με το πώς θα απαντήσουμε μπορεί να είναι ένα βιώσιμο σύστημα ή όχι. Σίγουρα όμως δεν πρόκειται για μια de facto λύση του ζητήματος αν είχατε κατά νου μία διαλογή πριν από το σύστημα ασύλου, να σα πω ότι εγώ δουλεύω στην Ελβετία. Έχουν κάνει πολλέ διαφορετικέ μεταρρυθμίσει τη ε, ε, νομοθεσία ε, ασύλου. Δεν την άφησαν την έρημη νομοθεσία ήσυχη ούτε για δύο χρόνια. Προσπάθησαν με, με διάφορα είδη ε, διαδικασιών μη παραδεκτού, ε, άλλε διαδικασίες διαλογής και τελικά είδαν ότι απλώς χάνουν χρόνο και χρήματα. Ήταν πολύ πιο απλό να έχουν πολύ λίγες αιτίε ε, μη παραδεκτού και να έχουν μια καλή διαδικασία ασύλου. Δεν πρέπει λοιπόν να χαθούμε σε αδιέξοδες καταστάσεις. Άλλο ερώτημα. Υποχρεωτική ανακατανομή. Αν δεν θέλετε κάτι τέτοιο, πώ θα βελτιώσουμε την ελληνική. Βέβαια είναι δύσκολο να απαντήσει κανεί μέσα σε ένα λεπτό σε αυτό το ερώτημα. Έχω ε, γράψει μακροσκελή κείμενα για αυτό το ζήτημα και βεβαίω μπορώ να αποστείλω αυτά τα γραπτά μου στη γραμματεία. Κάποια από αυτά τα απίφθηνα και προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σας πω ότι το μείζον ε, ερώτημα εδώ είναι πώς θα ελεγχιστοποιήσουμε το κόστος και τον χρόνο που χρειάζεται από τη στιγμή της άφηξης του ετούντος μέχρι την ε, ένταξή του στη διαδικασία. Για να γίνει αυτό θα έπρεπε να υπάρχει αυτό ο κανόνα που είχε ζητήσει η Πατιαρμοστία εδώ και 20 χρόνια. Η αίτηση εξετάζεται εκεί που υποβάλλεται, Εκτό και αν μπορούμε να μεταφέρουμε το πρόσωπο με τη συγκατάθεσή του σε ένα μέρο ε, όπου διαμένει η οικογένειά του ή σε ένα κράτο που δεν επομίζεται τι ίδιε ευθύνε. Αλλά και πάλι με τη συνένεσή του, με τη συγκατάθεσή του. Αλλιώ ξαναμπαίνουμε σε ένα ολόκληρο τέτοιο κύκλωμα νομικών ε, διαδικασιών, εξαναγκασμού και ούτω Φυσικά αυτό ε, διαφέρει σε πολύ μεγάλη ανισοκατανομή του κόστους και των ευθυνών. Αλλά γι' αυτό έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, έτσι δεν είναι. Προς το παρόν, οι οικονομικές μεταφορές είναι απειροελάχιστες και δεν καλύπτουν το κόστος ε, που ε, επισύρει η υποδοχή και ταυτοποίηση των προσφύγων. Αν είχαμε την δημοσιονομική ισοδυναμία, δεν θα ίσχυε όμως κάτι τέτοιο. Τέλο, μία από τι πηγέ ένταση είναι το γεγονό ότι οι ετούντε φοβούνται ότι θα μείνουν εγκλωβισμένοι για πάντα σε ένα μέρο όπου δεν έχουν ούτε δεσμού ούτε οικογένεια καμία σχέση. Αν του υποσχεθούμε ότι θα λάβουν καθεστώ προστασία, τελικά θα καταφέρουν να πάνε σε ένα μέρο όπου έχουν δεσμού, δυνατότητε απασχόληση κ.ο.κ. Σε τελική ανάλυση, στο άρθρο 78 δεν αναφέρεται ρητός ε, ότι έχουμε ένα τέτοιο καθεστώς το οποίο θα ισχύει σε όλη την επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθούσε. Μπορεί να κάνω λάθος. Είμαι στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε. Κάτι τελευταίο προς την κυρία Ernst. Για τις ρήτρες οικογενειακής επανένωσης. Τι κάνουμε στο νέο κανονισμό. Είναι σαφές. Αν έχετε ακούσει όλες τις παρεμβάσεις, διευρύνουμε τις ε, ρήτρε κατά τι προκειμένου να τις ε, καταστήσουμε εφαρμοστέ όχι μόνο σε εξαιρετικέ περιπτώσεις. Πρώτον, και για να έχουμε πιο σαφείς ε, κανόνες ό,τι έχει να κάνει με την τεκμήριωση, με τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό που λέω εγώ για τις δυνατότητες ε, του κανονισμού Δουβλίνου είναι ότι ήδη είναι πολλέ για την βελτίωση του συστήματος δεν θέλω να διαφημίσω το έργο μου και να περιευθολογήσω, αλλά για τους σκοπούς ε, της σημερινή ε, συζήτηση. έχω δημοσιοποιήσει μια μελέτη πρόσφατα για τις ε, ερμηνείες που δίνονται στις ρήτρε οικογενειακή επανένωσης. Με τα χαράς να την αποστείλω στη γραμματεία. Το βασικό μήνυμα είναι ότι υπάρχουν πολλά δόγματα και προσεγγίσεις ότι έχει να κάνει με τα αποδεικτικά στοιχεία και την οικογενειακή επανένωση. Και όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε πολύ περισσότερε περιπτώσει από ό,τι γίνεται σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να θυμίσω στους συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα ότι θα ξαναρχίσουμε στις 3. Και έχουμε πάρα πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη και το απόγευμα. Έχουμε διαθωμένο διάλογο με την Αντιπρόεδρο Γιούροβα, μετά με τον Αντιπρόεδρο Σκίνα. Στις 3 θα είναι εδώ. Και μετά από αυτή τη συνεδρίαση έχουμε και τη συνάντηση των συντονιστών τελευταίος που θα πάρει το λόγο για τις καταλεκτήριες παρατηρήσει, εσείς. Ω εισηγήτρια για το θέμα, κυρία Κελέρ, έχετε το λόγο. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συμμετέχοντες, ε, τους υπαλλήλους, τους βουλευτές, όσοι ετοίμασαν το πάνελ τα διάφορα πάνελ, τους προσκεκλημένους μας, με μια εξαίρεση από εκείνη την πλευρά βέβαια, που ευτυχώς σκόθηκα και έφυγαν εκείνοι οι συνάδελφοι. Θέλω να τονίσω την καλή διάθεση όλων ε, για να συνεργαστούμε. Όλοι έχουν διάθεση να παρουσιάσουν την δουλειά τους στα όρια που μπορεί να υπάρχουν πρακτικά και να μοιραστούν τις ε, πρακτικές τους για να κάνουμε όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε μαζί. Ευχαριστώ για αυτό το κλίμα συνεργασίας λοιπόν, ε, γιατί αυτό ακριβώς ε, μας εμπνέει όλους και διέπει τη δουλειά μας, εμένα και των υπόλοιπων σκιωδών συγκητών. Κάποιες ιδέες, σημεία, ε, εντάχει, αν και άλλα αναφέρθηκαν πάλι στην ε, συζήτηση, η διακυβέρνηση, η διαχείριση του θέματος, πώς θα συνεργαστούμε μεταξύ μας για να τονώσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τους παράγοντες που δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνη. Ε, μετά πώς θα ασχοληθούμε με τα κίνητρα για τις βασικές ροές και πώς θα κοιτάξουμε να εφαρμόσουμε καλύτερα την οικογενειακή επανένωση και την ε, μετανάστευση για λόγους επαγγελματικού. με πτυχία, με δεξιότητες ή χωρίς δεξιότητες. Επίσης το θέμα των ε, χρονικών διαστημάτων, της προθεσμίας και του χρόνου. Ε, το χρόνο. Δεν χρειάζεται λίγος χρόνος για να εξετάσει κανεί, καλά κανείς μια αίτηση ασύλου. Υπάρχει όμως και το πρόβλημα των καθυστερήσεων με τις διάφορες ατέλειες επικοινωνίας. Πρόεδρε, αυτές ήταν οι παρατηρήσεις. Με ευχαριστώ πολύ που οργανώσατε τη συνεδρίαση σήμερα το πρωί. Πραγματικά δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει την πορεία μα και ευχαριστώ πολύ για την ενέργεια, τον ενθουσιασμό σα, για όλη τη δουλειά που κάνουμε για να εφαρμόσουμε καλύτερα το δίκαιο περί σε σεβόμενοι πλήρω τι διεθνεί υποχρεώσει και δεσμεύσει μα. Απέναντία, κυρία Κελέρ, εσά ευχαριστούμε. Είστε εισηγήτρια και είναι απολύτω φυσικό να εξετάσουμε αυτό το κατεπήγον θέμα το οποίο συζητήθηκε και με καμάρι θα έλεγα από την Επιτροπή Λίμπε. Αφιερώσαμε ολόκληρο πρωινό σε αυτή την ακρόαση. Να σας θυμίσω, η συνεδρίαση πρέπει... Α, εδώ θα γίνει η συνάντηση των συντονιστών. Ανακοινώνω ότι σε αυτήν ακριβώ την αίθουσα στι 3 θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μα. Προηγουμένω όμω έχουμε και τη συνεδρίαση των συντονιστών τώρα, ευθύ αμέσω.